Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Χτες ε, διακόπη η συνεδρίασή μας, διακόπη συνεργασία μας πιο σωστά και ξεκινάμε ε, με την ε, σημερινή μας ημερήσια διάταξη που σήμερα προβλέπεται η συζήτηση για το Γενικό προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και χαιρετίζω θερμά τον Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου μας, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον ε, προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναφέρομαι βέβαια στον κύριο Τζάνι Πιτέλα. Σας καλωσορίζουμε θερμά στην Επιτροπή μας. Και εξίσου θερμά χαιρετίζω και το Γενικό Γραμματέα του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Κλάους Βέλε, όπως επίσης και τον ε, εσωτερικό ελεγκτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Γκάλβιν. Καλωσορίσατε και επίσης κύριε Μπαντήλιο το Μερούζα. Η συγγήτρια για αυτό το θέμα της μερίσιας διάταξης ε, είναι η συνάδελφος Εύα Ότης Βιλέα και θα ήθελα να της δώσω το λόγο για να κάνει την εισαγωγή. Εύα, παρακαλώ, αν θέλετε έχετε το λόγο. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να χαιρετήσω και όλα τα πρόσωπα τα οποία ανέφερε ο Πρόεδρος. Και ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Βέλη που βρίσκεται ενώπιον μας σε αυτή την Επιτροπή για να μας μιλήσει για τον προπολογισμό του Ευρωκοινοβουλίου και τον, ε, του 2011 για την απαλλαγή αυτού. <coughs> Λόγω της περίοδου που διανύουμε θέλουμε να εξετάσουμε σε βάθος ε, τις εξελίξεις. Οι συνεδριάσεις που είχα αυτόν τον καιρό με τους Γενικούς Διευθυντές του Ευρωκοινοβουλίου και τον εσωτερικό ελεκτή είχε ως στόχο να διασφαλίσουν ότι το δημόσιο χρήμα δαπανάται με τρόπο ποδοτικό και ικανοποιητικό. προτίθεμε να πετύχω μια απαλλαγή η οποία θα τύχει πλήρους έγκρισης και ενδεχόμενα να διασκεδάσω ενδεχόμενε ανησυχίε ε, που έχουν Θα ήθελα να ευχαριστήσω για, την για τον επαγγελματισμό και την ε, διαθεσιμότητα όλων ε, όσων συνάντησα. Θα έπρεπε να πω ότι όλε οι συναντήσει μου ήταν ιδιαίτερα καρποφόρε και διευκρινιστικέ. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το γεγονό ότι μου αναθέσατε την να είμαι για τον προπολογισμό 2011. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις προτάσεις και για τα τελικά του σχόλια, καθώς επίσης και τη συνεργασία της ομάδας εργασία που με συνόδεψε σε αυτό το σημαντικό έργο μου. Θα ήθελα να σχολιάσω διάφορα θέματα τα οποία θεωρήσαμε σημαντικά κατά τη διάρκεια των εργασιών μας. Το 2011 εγκρίθη ένα επιπλέον ε, σύνδελο μέτρων για την ε, δαπάνη των πόρων. Επίση εξετάζουμε θέμα της μετάφραση ε, των γράφων, τη σημερινή αποζημίωση ε, για τι αποστολέ. και όλε τι συγκρίνουν με τις αποστολές των, των συναδέλφων. Όλα αυτά όμω, δεν μα επέτρεψαν να κάνουμε τι απαραίτητε ε, οικονομίε για, τι τις, για τις εργασίες μας. Θα ευχαριστήσω όμω και τον κύριο Βέλε για την προσπαθία του. Θα ήθελα να πω ότι ακολουθήσαμε τις ε, διάφορες συστάσεις ε, που είχαν ληφθεί υπόψη κατά την απαλλαγή του 2010. Συγχαρώ για την ε, επιτυχία του Βαλεμετάριου που από την έναρξη των εργασιών του φαίνεται ότι λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά, αποτελεί ένα πόλο έλξη εξέλιξης ε, τουριστικές της Βρυξέλλες ε, και το feedback ήταν ιδιαίτερα θετικό για όλους όσοι το επισκέφθηκαν και από αποτελεί με αναφορά για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα του 2011 είδαμε πως ε, συμπεριφθήκε και το ζήτημα της εσωτερήκευσης στο Λουξεμβούργο, στις Βρυξέλλες αλλά και το Στρασβούργο. Βρισκόμαστε λοιπόν πιο κοντά στην πλήρη εσωτερήκευση των ε, θεμάτων αυτών στο Κοινοβούλιο, κάτι το οποίο διασφαλίζει και την ασφάλεια του οίκου μας. Το θέμα λοιπόν είναι σημαντικό και πάντα ήταν ε, στόχος διαφόρων ε, κριτικών που είχαν ασκηθεί τα τελευταία χρόνια. Μας είπαν ότι με το νέο αυτό σύστημα, πέραν του ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια, αυτό θα κοστίζει και λιγότερο. Ζήτημα πολύ σημαντικό στους, στους καιρούς μας ε, κάναμε πράγματα πολύ σημαντικά και σας συγχαίρω γι' αυτό, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την περαιτέρω τα πράγματα. Έτσι, συνεχίζοντας με το θέμα της ασφάλειας, θα πρέπει να βελτιωθούμε. Το Κοινοβούλιο είναι ένα σώμα το οποίο επισκέπτονται αρχηγοί κυβερνήσεων ε, κάθε εβδομάδα θα έλεγα. Θα ήθελα λοιπόν να διευκρινιστεί κατά πόσον θα υπάρξει η υποχρεωτικότητα, υποχρεωτικός χαρακτήρας ε, της χρήσης μαγνητικών badge ε, και για του βουλευτέ. Θα θέλαμε κύριε Βέλη να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες του σχεδίου και ελπίζω να μην ε, δυσκολέψει την κινητικότητα των βουλευτών προκειμένου να κυκλοφορούν ελεύθερα και άνετα αλλά και ασφαλώς στα κτίρια μας. Ο υψηλός αριθμός ευρωβουλευτές, επισκέπτες και υπάλληλοι. Όπως καταλαβαίνετε επηρεάζονται από αυτές τις διαδικασίες. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα του catering που σε κάποιες ώρες πραγματικά ε, ε, βρίσκεται στα όρια του. Ένα άλλο ζήτημα έχει σχέση με τον οίκο της ιστορίας. Ε, φαίνεται ότι το ζήτημα προχωράει και θα ανοίξει τις πόρτες του το κτίριο του Σεπτέμβριο 2014 με ενισχύει η χρηματοδότηση αυτού του σχεδίου, αυτού του προγράμματος γι' αυτό. Τον Νοέμβριο 2012, όπως θυμόσαστε, το συζητήσαμε το ζήτημα, αλλά θα ήθελα τώρα με την ευκαιρία της απαλλαγής Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε την επιθυμία τη να συμμετάσχει στην κόστο αυτού του σχεδίου. Υπάρχει επιστολή του Προέδρου Μπαρόζου στον πρώην πρόεδρο του Βουλίου Μπούζεκ, όπου εκφράζει την πρόθεσή του να συμμετέχει η Κομισιόν στι δαπάνε και θα ε, αφορά το έτος ε, και τον προπολογισμό του 2013. Τι έγινε τελικά, έχει προχωρήσει το ζήτημα, ήταν μια ε, δήλωση προθέσεων, πού ακριβώς βρισκόμαστε σε ό,τι φορά τον ε, αριθμό των εργαζομένων ε, φαίνεται ότι θα πρέπει να προσληφθούν επιπλέον ε, εννέα άτομα. Από πού θα, προσληφθούν βρεθούν τα άτομα αυτά, πώς θα προσληφθούν, θα είναι προσωρινοί υπάλληλοι, θα είναι επισυμβάσει, τι. Επίσης, ποια θα είναι η συμμετοχή της βελικού κράτους σε αυτό τον ευρωπαϊκό οίκο. και θα, θα θέλαμε να γνωρίζουμε λοιπόν πώ θα συμβάλλει η βελική κυβέρνηση. Στην αρχή τη παρεμβάσεώ μου μίλησα για την καρποφόρα και αποδοτική συνάντηση που, συναντήσει που είχα τι προηγούμενε εβδομάδε. ε, μία από αυτέ ήταν με τον κύριο Γκάλβιν, τον εσωτερικό ελεγκτή και μου έπεσε την προσοχή στην ανάγκη για ένα καλύτερο προγραμματισμό των γενικών διευθύνσεων διότι ε, συχνά συμμετέχουν σε έκτακτες ε, διαπραγματεύσεις και αναφέρθηκε επίσης στις συμβάσεις ε, οι οποίες έχουν συναυθεί για τα ζητήματα αυτά τα πάντως κύριε Βέλε δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε μια, ένα κακό προγραμματισμό διότι αυτό αποτελεί σπατάλη πόρων αν και διαπίστωσα ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά, αλλά θα ήθελα να το αναφέρω για μια ακόμα φορά. Θα ήθελα να γνωρίζω επίση δεν υπάρχει κάποια ημερομηνία για την ε, ψήφιση τη ε, έκθεση, σχετική έκθεση στην Ολομέλεια, διότι με τα προβλήματα τη ε, αίθουσα Ολομέλεια και με τη μήνυ σύνοδο ξέρουμε, ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να ψηφιστεί κανονικά πριν από τα τέλη Μαΐου. Απλά πότε θα γίνει αυτή η ψήφιση. Έχετε υπόψη σα για κάτι ακόμα χωρίς να έχουμε τη μελέτη για το κόστος των εργασιών και την ενίσχυση της μεταλλικής δομής του ημιτικλίου Και πότε προβλέπεται να δημοσιευθεί η, η σχετική δήλωση σε ό,τι αφορά τώρα την ασφάλεια των ε, κτηρίων μετά από το ότι συνέβη με τον ε, ημικύκλιο στο Στρασβούργο, θα έπρεπε να ελεγχθούν όλα τα κοινοβουλευτικά κτίρια για να βελτιώσουμε την ασφάλεια τους. Επίσης, ε, να πω ότι θα πρέπει να λυθούν τα προβλήματα με την υπηρεσία ηλεκτρονικών, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διότι ε, ε, η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εξεπλάγει όταν την περσμένη εβδομάδα υπήρχε, υπήρξε πρόβλημα με το mail του Κοινοβουλίου λέγοντας ότι δεν υπήρχε έλεγχος με τον πάροχο. Θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να χάσει αυτόν τον έλεγχο και αυτές τις ε, γνώσεις που θα πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι στον τομέα αυτό. Και τέλος, ε, να σας πω κάτι το οποίο παρατήρησα, ότι αν δεν σφάλω, το ίμιση των ε, ζητημάτων οι υπηρεσίες αναφέρθηκαν ότι αφορούν στον απολογή του προβλησμού 2011. Δεν είναι έτσι σε όλες τις περιπτώσεις όμως μόνο ότι αυτέ ήταν οι απαντήσει τη γραμματεία. Η ερώτηση 20 παραδείγματο χάρη για την ε, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματο. Διότι θίγεται το θέμα τη διαχείρισης, οικονομική διαχείριση του 2011. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε όμω ε, τον προπολογισμό και να τον εξετάσουμε μονομερός. Λοιπόν, εγώ φρόντισα να περιλάβω όλε τι ερωτήσει των πολιτικών ομάδων και να τι περιλάβω στο ερωτηματολόγιο και κάτι ακόμα. Ε, οι δύο τελευταίες ερωτήσεις ε, θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς. Η πρώτη από αυτέ αναφέρεται στην ε, ε, στο Γραφείο Ταξιδίων. Πολλοί παραπονιούνται ότι είναι ιδιαίτερα ακριβή και μπορεί να αγοράζει κανείς ε, πολύ φθηνότερα ειστήρια χρησιμοποιώντας το ίντερνετ. Ε, υπόθηκε ότι αυτό δεν αφορά το 2011, αλλά εγώ επέμεινα στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις αλλά και σε άλλες. Θα πρέπει να εξεταστεί περισσότερο το θέμα του γραφείου ταξιδίων ε, αν θα μπορούσατε να μας ε, μιλήσετε περισσότερο για το καθεστώς ε, των βοηθών των βουλευτών και μια ακόμα ερώτηση για τα intergroups στο Κοινοβούλιο. Να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου που βρισκόσαστε σήμερα εδώ ενώπιόν μας για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο και σε όλους τους γενικούς διευθυντές και υπεύθυνου που συνεργάστηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Διευθυντή του Ελεγκτικού Συνεκνητρίου, τον κύριο Τόμι Ρουκουρούχφα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της ε, Επιτροπής Ελέγχου Προεπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το κεφάλαιο 9 της αιτής ετέξης του Ελληνικού Συνεδρίου παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ειδική αξιολόγηση διοικητικής δαπάνης ε, των οργάνων και άλλων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομάδα πολιτικής, διοικητικές και λοιπές δαπάνες εκπροσωπεί 7,6% των συνολικών πληρωμών του 2011 και συμπεριλαμβάνει κυρίως τις δαπάνες για τους ανθρώπινους πόρους όπως μισθούς, επιδόματα και συντάξεις, ε, δαπάνες για κτίρια, εξοπλισμό, ενέργεια, πληροφορία, ε, τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίες. Το ε, συνέδριο έλεγξε αντιπροσωπευτικό δείγμα συναλλαγών που καλύπτουν διοικητικέ και λοιπέ δαπάνε όλων των οργάνων και υπηρεσιών και αξιολογεί ε, την συμμόρφωση των εποπτικών και ελεγκτικών συστημάτων ε, κάθε οργάνου με του, τις απαιτήσει του δημοσιονομικού κανονισμού. Επίσης, το ελεγκτικό συνέδριο επέλεξε θέματα όπως ο υπολογισμός και πληρωμή κοινωνικών επιδομάτων ε, για το προσωπικό όλων των οργάνων, τις διαδικασίες παράτασης και τροποποίησης των συμβάσεων των προσωρινών και συμβασιούχων, όπως επίσης και συμβάσεις προμηθειών στα περισσότερα όργανα. Όπως και τα προηγούμενα έτη, το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης είναι θετικό. Το Ελεκτικό Συνέδριο συμπεραίνει ότι οι συναλλαγές διοικητικών και λοιπόν δαπανών το 2011 ήταν ε, σε κάθε, από, από απόψεως σημαντικότητας ε, νόμιμες και τυπικές. Ε, συγκεκριμένα 7% των 56 συναλλαγών ε, είχαν σφάλμα και το πιο πιθανό ε, ποσοστό σφάλματος είναι 0,1%. Επίσης, διαπιστώνουμε ότι τα εποπτικά και ελεγκτικά συστήματα των διοικητικών δαπανών συνάδουν με τις απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, και μέλη του Κοινοβουλίου. Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη ε, ότι το Ελεκτικό συνέδριο γνωμοδοτεί για όλου, όλα τα όργανα ε, και όλους, όλες τις υπηρεσίες ε, συνολικά και δεν γνωμοδοτεί ξεχωριστά για καθένα από αυτά. Παρόλα αυτά, ε, προβαίνει σε ειδική επιπλέον εργασία ε, για κάθε όργανο και υπηρεσία και παρουσιάζει κάποιες παρατηρήσεις για κάθε ένα από αυτά. Τα πορίσματα δεν θέτουν ένα αμφιβόλο την ειδική αξιολόγηση του ελεκτικού συνεδρίου. Οι συστάσεις προς ε, κάποια όργανα και υπηρεσίες ήταν οι εξής τρεις. Πρώτον, το προσωπικό πρέπει ε, σε τακτά χρονικά διαστήματα να υποβάλει έγγραφα που επιβεβαιώνουν την προσωπική κατάσταση ε, των οργάνων και των υπηρεσιών ε, ε, όπως επίσης και εφαρμογή ενός συστήματος της καλής παρακολούθησης του συστήματος. Δεύτερον, τα όργανα και οι υπηρεσίες πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες για την σύναψη, παράταση και τροποποίηση συμβάσεων με μη μόνιμο προσωπικό. Και τρίτον, τρίτον τα όργανα και οι υπηρεσίες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι συγκεκριμένοι ε, ε, υπεύθυνοι βελτιώνουν τον συντονισμό, προγραμματισμό και επίδοση και αποτελέσματα των διαδικασιών προμηθειών μέσω σωστών ελέγχων και καλύτερης καθοδήγησης. Επίσης βρέθηκαν ε, δυναμίες στις πληρωμές των κοινωνικών επιδομάτων σε δύο περιπτώσεις από τις, πέντε, που ελέγχθηκαν η κατάσταση δεν ήταν σωστά ενημερωμένη, ούτε είχε γίνει σωστή επεξεργασία και σε πολλές περιπτώσεις υπήρξαν υπερβολικές καταβολές ποσών. Επίσης βρήκαμε κάποιες παρατυπίες ε, στο σύστημα των εξουσιοδοτημένων ε, βοηθών. Ε, στις πέντε από τις δέκα περιπτώσεις τα ιατρικά πιστοποιητικά παρουσιάστηκαν πολύ αργά και σε καμία από τις 10 περιπτώσεις δεν υπήρξαν έγγραφα που να δείχνουν ότι έχουν γίνει ιατρική ή έλεγχη ε, σε σχέση, είχαν γίνει έλεγχοι σε σχέση με την γνώση των γλωσσών. Επίσης, ε, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των εκ των προτέρων ελέγχων, υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί σε σχέση με την ε, πρόσληψη 9 εκ των 10 βοηθών που ελέγχθηκαν. Επίσης, υπήρξαν κάποια προβλήματα στις δύο διαδικασίες προμηθειών από τις 10 όσον αφορά τα κριτήρια απονομής και επιλογής για την συντήρηση κτηρίων όπως επίσης και για τις υπηρεσίες εκτύπωσης. Στην ετήσια έκθεσή του το Συμβούλιο επίσης σχολιάζει τις εξελίξεις σε σχέση με τις συστάσεις που έγιναν τα τελευταία σε σχέση με τις συστάσεις που έγιναν στις τελευταίες εκθέσεις, προηγούμενες εκθέσεις και μία από αυτές έχει να κάνει με το, την παρακολούθηση, τη συνέχιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το follow-up. Όσον αφορά την, ε, τις πληρωμές των κοινωνικών επιδομάτων ε, στο προσωπικό, δείχνει ότι υπήρχε, υπάρχει ένας κίνδυνος ε, λανθασμένων και αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Κύριε Πρόεδρε και ε, αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, ε, πρόκειται για μια σύνοψη των πορισμάτων του ελεκτικού συνεδρίου. Ευχαρίστω να απαντήσω σε ερωτήματα, ε, αν θέλετε να μου θέσετε, και σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τομέμου Κουρούθα για την θέση του Ελεκτικού συνεδρίου και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πιτέλα, στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, καταρχήν να σας ε, καλημερίσω, να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα, τα μέλη του Ελεκτρικού Συνεδρίου και όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Ε, καλημερίζω και την κυρία Εισηγήτρια, κυρία Εύα Όρτης Μιλέια και τους υπόλοιπους σκιώδεις ηγητέ. και θα ήθελα να διαβεβαιώσω την εισηγήτρια και τους υπόλοιπους σκιώδεις ηγητέ ότι η ε, ανησυχία και η υποχρέωση για μια υγιή και αποτελεσματική διαχείριση του προπολισμού είναι και δικό μας μέλημα και δική μας υποχρέωση. Χαιρετίζω τον δόκτωρα Μουγκρούτ από το ελεγκτικό συνέδριο και Εκφράζει την ικανοποίησή μου για τις θετικές απόψεις που, που εκφράζει μέσα από την έκθεσή του σχετικά με τις εργασίες. Καλημερίζω και τον κύριο Ρόμπερτ Γκάλβιν, που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο του Κοινοβουλίου και όπως καθέμισα και σε προηγούμενες συναντήσεις, εγώ είχα την τιμή να είμαι μέλος της Επιτροπής σας κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου και θυμάμαι και έχω πολύ καλές αναμνήσεις από εκείνη την εποχή. Όσοι ήθιστε, σήμερα με συνοδεύει ο Γενικό Γραμματέα Κλάου Βέλε και ο Δ. Γκάλιν που συμμετέχουν σε αυτήν την ανταλλαγή ε, απόψεων που θα βρίσκονται στη διάθεσή σα ε, από. Ε, και η ανταλλαγή αυτή απόψεων είναι να εξετάσουμε τα εγγεγραμμένα ποσά στον προβλεσμό αλλά και τις πιστώσεις που προέρχονται από αποφάσεις που έχει λάβει το Προεδρείο του Κοινοβουλίου και που είχαν επιπτώσεις στον προϋπολογισμό. Νομίζω ότι λάβατε ήδη τον κατάλογο αυτών των αποφάσεων και έτσι δεν θα τις επαναλάβω. Επίσης πρέπει να έχετε λάβει και τι απαντήσει του Γενικού Γραμματέα για το ερωτηματολόγιο περί της απαλλαγής που αποτελούν απάντηση στα ερωτήματα που θέσατε και θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω ερωτήσεων. Προτού να δώσω το λόγο στου στους ε, αγορητές θα ήθελα να τονίσω ένα σημείο που μα είναι ιδιαίτερα ε, ενδιαφέρον, δηλαδή διαφάνεια, συνεργασία και διάλογος είναι και παραμένουν σταθερές θεμελιώδεις ε, για τις εργασίες μας. Το Προεδρείο ενεργεί προκειμένου οι σχέσεις ανάμεσα στους ε, εμπλεκόμενους ε, στα ζητήματα προϋπολογισμού του σώματός μας να είναι διάφανα και να την χάνουν υγιούς διαχείρισης, χρηστής διαχείρισης. Νομίζω ότι είναι κοινό μέλημα να μην υπάρξει υπερβάλλον ζήλος στα αυτά τα ζητήματα, διότι αυτό θα έρχονταν σε αντίθεση με το πνεύμα της απαλλαγής. Η συγκεκριά είπε, αλλά και η έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου, ότι υπάρχουν κάποιες κριτικές που έχουν σκεφτεί. και αν υπάρχουν κριτικές, τότε σίγουρα θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει να το πράξουμε με πνεύμα συνεργασίας και παράλληλα αποφεύγοντας την δημαγωγία και την ε, αδιαφορία. Ε, ο Γενικό Ρωματέας θα δώσει απαντήσεις και προφορικά για κάθε σημείο και εγώ θα ήθελα να εκφράσω επισήμως και να επαναλάβω προς τον Γενικό Γραμματέα και προς όλες τις γενικές διευθύνσεις του Κοινοβουλίου την ε, μέγιστη εκτίμησή μου και εμπιστοσύνη που φέρω από κοινού με τον Βίνταλ Κουάντρας και τους άλλους συναδέλφους στο Προεδρείο για τις εργασίες τους. Μαζί με τον κύριο Βίνταλ Κουάντρο επαναλαμβάνω την πρόθεσή μας για ε, περαιτέρω συνεργασία. Κάθε φορά που οι ερωτήσεις σας θα αφορούν τη χρηστή διαχείριση και τη διαφάνεια, σίγουρα θα λάβουν τις κατάλληλες απαντήσεις ε, με ειλικρίνεια και ορθότητα. Δίνω το λόγο στον Γενικό Γραμματέα. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πιτέλα και για τα πολύ φιλικά ε, λόγια που βρήκατε για την ε, δουλειά των ανθρώπων που εργάστηκαν σε αυτή την Επιτροπή. Βεβαίως επειδή υπάρχουν διάφορα θέματα που διακυβεύονται, αυτά που είπατε κύριε Πιτέλα ήταν πολύ ενθαρρυντικά και σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Κλάους Βέλε, το Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώντας ε, την ε, παρουσίασή μου θα μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω και να σας υπενθυμίσω ορισμένα βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού του 2011 γιατί σήμερα ε, για αυτή την απαλλαγή μιλάμε. Το 2011 ήταν καθοριστικό έτος γιατί από τη μια πλευρά ήταν η χρονιά εκείνη όπου ε, αφήναμε την παλιά μέθοδο και έπρεπε να προσαρμοστούμε στην συνθήκη της Λισαβόνας. Επιπλέον προσθέθηκαν 18 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πήραμε 35 θέσεις ε, για την περίφημη Policy Department, δηλαδή για να ενισχύσουμε τη δυνατότητά μας ε, διαβούλευσης. Επίσης ένα αριθμό ε, θέσεων στη βιβλιοθήκη, για υποτροφίες και πολλά άλλα. Ε, παράλληλα, άνοιξε και το Παρλαμεντάριουμ, το κέντρο επισκεπτών. Το επισήμανε αυτό η συγγήτρια. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μας έχει απασχολήσει επανειλημμένα ε, και στην Επιτροπή Προπολογισμών υπήρχαν πολλέ προσδοκίε, αλλά μερικέ φορέ εκφράστηκαν και φόβοι. Εν τω μεταξύ, μπορούμε να πούμε ότι το Παρλαμεντάριο μετά από πάνω από ένα χρόνο λειτουργίε, σημειώνει ιδιαίτερη επιτυχία. Ε, την πρώτη χρονιά είχαμε περίπου 200 ε, τόσες χιλιάδες επισκέπτες ε, πάνω από τις προσδοκίες μας και εντωμεταξύ νομίζω ότι το Παρλαμεντάριο έχει γίνει σημαντικό εργαλείο βοήθειας και για τους βουλευτές. Είναι και ένα ιδιαίτερα ελκυστικό σημείο στις Βρυξέλλες που τραβά πολλούς τουρίστες. Πολύ επιτυχημένο λοιπόν. Επίσης είχαμε και το πρόγραμμα της διεύθυνση πόρων. Αυτό εφαρμόστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που σημαίνει ότι τώρα ε, όλες οι μεγάλες και οι μεσαίες μεγάλες ε, διευθύνσεις ε, έχουν δικό τους προσωπικό που ασχολείται με τη διαχείριση του προσωπικού και με θέματα πληροφορικής. Αποτέλεσμα αυτού είναι ιδιαίτερα καλές τεχνικές γνώσεις και έτσι οι γενικές διευθύνσεις έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται οριζόντια, να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να είναι αποτελεσματικό συνεργάτης για άλλες γενικές διευθύνσεις. Και αυτό το μέτρο λοιπόν αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένο. Στο τέλος του έτους 2011 ε, ανανεώσαμε τη συνεργασία μας με το Λουξεμβούργο ε, στο θέμα της χρηματοδότησης του ε, κτηρίου Κόνατ Αντενάουρ. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου η οποία ανέλαβε επιπλέον υποχρεώσεις και η κυβέρνηση λοιπόν αυτή όχι μόνο θα μας στηρίζει κατά την υλοποίηση αυτού του προγράμματος αλλά θα προσφέρει και οικονομική βοήθεια παραδείγματο χάρη εγγύησης μισθώσεως κάτι το οποίο μας επιτρέπει να συνεχίσουμε την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Πιστεύω λοιπόν ότι από το πρίσμα των βουλευτών αλλά και των ε, συνεργατών ε, το Wi-Fi είναι καθοριστική σημασίας. Ήταν μια πολύ μεγάλη επένδυση ε, και βεβαίω και εσείς μας διαθέσατε τα απαραίτητα κονδύλια. Βασική προϋπόθεση ήταν βέβαια να μπορούμε να ε, χρησιμοποιήσουμε την ε, πληροφορική και τα κινητά τηλέφωνα και τα, τους κινητούς ε, υπολογιστές, τους, τα PC. Όλα αυτά όμως μπορέσαμε να τα ολοκληρώσουμε την περασμένη χρονιά. Η συγγήτρια επίσης αναφέρθηκε στην ανάληψη εκ μέρους μας, στην περίφημη εσωτερικοποίηση των ε, ε, διαπιστεύσεων. Γνωρίζετε ότι είχαμε κάποια επεισόδια και γι' αυτό το λόγο λάβαμε τα απαραίτητα μέτρα. Είμαι λοιπόν απόλυτα πεπισμένος ότι δεν αρκεί απλά να προσλαμβάνουμε ένστολους ε, για να διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Χρειαζόμαστε συνεργάτες οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι οι οποίοι γνωρίζουν πολλά χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νιώθουν αφοσίωση απέναντι σε αυτό. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το περιμένει αναγκαστικά από συνεργάτες με συμβάσεις ε, έργου, με συμβάσεις. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ε, Ξάγαμε τα απαραίτητα συμπεράσματα και όπως σας είπα η διαπίστευση εντωμεταξύ έχει ολοκληρωθεί. Το ίδιο ισχύει και για την ανάληψη εκ μέρους μας ε, το θέμα, ε, το θέμα αυτό, την εσωτερήκευση, όπως σας είπα, όπως αποκαλείται. Εφαρμόζεται λοιπόν στην πράξη αυτή η προσπάθεια και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του 2013 θα μπορούμε να την ε, έχουμε ολοκληρώσει, έτσι ώστε η διαπίστευση να έχει πλήρως εσωτερικευτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πριν περάσω στα συγκεκριμένα ερωτήματα της εισηγήτριας, θα ήθελα να σας παραπέμψω στο πρόγραμμα βελτιστοποίησης στον τομέα της παροχής γλωσσικών υπηρεσιών. Στον τομέα αυτό πραγματικά επιτεύχθηκαν εντυπωσιακά αποτελέσματα και αυτά σε συνεργασία με τους άμεσα θυγόμενους συνεργάτες προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα στον τομέα της μετάφρασης, της γραπτής μετάφρασης. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχαν ε, πολλές ε, διαφορές ε, στον όγκο της μετάφρασης αναεργαζόμενο και γι' αυτό αυτό ε, αναζητήσαμε και είδαμε που μπορούμε να κάνουμε μετακινήσεις ε, με φιλόδοξους στόχους, όχι βέβαια υπερβολικά φιλόδοξους, 100 ε, θέσεις εργασίας, περίπου δηλαδή το 10% του συνόλου σε δύο χρόνια χρησιμοποιήθηκαν σε άλλη θέση. Και με τον τρόπο αυτό μπορέσαμε να επανδρώσουμε τη νέα διεύθυνση για τη μελέτη αντικτύπου χωρίς να εισάγουμε νέες θέσεις εργασίας εμβας Εν πάση περιπτώσει, είμαστε και στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι και για το σπίτι της ευρωπαϊκής ιστορίας δεν προσθέσαμε θέσεις εργασίας στο οργανόγραμμα. Θα καλυφθούν οι θέσεις από μετατάξεις, από εκεί όπου υπάρχουν ε, περισευούμενοι πόροι και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη διαχείριση. Εξάλλου έχουμε μια νέα προσέγγιση και στον τομέα της γραπτής μετάφρασης. Δηλαδή, <clears throat> περνάμε σε μια άλλη μορφή εργασίας. Προσφέρεται η υπηρεσία εφόσον ζητείτε on demand. Έχουμε τα πρακτικά των ε, ολομελιών ε, σε όλες τις γλώσσες. Το κατά το παρελθόν γινόταν αυτόματα σε όλες τις γλώσσες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με υπέρογκο κόστος. Τώρα το σύστημα το αλλάξαμε και είπαμε ότι ακόμα και αν ένας και μόνο ευρωβουλευτής επιθυμεί τη μετάφραση των πρακτικών στη γλώσσα του θα του την προσφέρουμε. Όμως δεν θα κάνουμε τη μετάφραση αν δεν γνωρίζουμε ότι θα χρησιμοποιηθεί. Αποτέλεσμα αυτού το 2012 δεν έγινε δεν ζητήθηκε ούτε μία γραπτή μετάφραση των πρακτικών. 8,4 εκατομμύρια ευρώ εξοικονομήσαμε από το γεγονός αυτό. Το ποσό επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και δεν υπήρξε καμία απώλεια παροχής υπηρεσίας ε, για ευρωβουλευτή. Γιατί αν κάποιος ευρωβουλευτή το είχε ζητήσει θα του είχε προσφερθεί. Αυτή λοιπόν είναι μια σημαντική βελτίωση. Και στον τομέα της διερμηνίας. Το 2011 και εκεί λάβαμε σημαντικές αποφάσεις. Ε, πολιτικές αποφάσεις, κατά κύριο λόγο τρεις. Δηλαδή παρακαλέσαμε τις επιτροπές και ξέρω ότι αυτό στην αρχή ήταν λιγάκι επίμαχο. Τους είπαμε να συνεδριάζουν είτε Δευτέρα Τρίτη είτε Τετάρτη Πέμπτη. Αλλά όχι όλοι Τρίτη και Τετάρτη. Αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα ότι στον τομέα της ε, διερμηνίας χρησιμοποίησαμε πολύ περισσότερο τους υπαλλήλους διερμηνείς οι οποίοι είναι στη διάθεσή μας από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και δεν χρειάστηκε ε, να καταφεύγουμε στους ε, ελεύθερους συνεργάτες που τους προσλαμβάναμε για τις ημέρες εχμής Τρίτη και Τετάρτη. Εξοικονομήσαμε λοιπόν 10 εκατομμύρια ευρώ από την κίνηση αυτή και στο τέλος του 2012 ε, διαπιστώσαμε ότι η πραγματική εξοικονόμηση δεν ήταν 10 αλλά 15 εκατομμύρια ευρώ. Και επιπλέον προέκυψε και το εξής. Τώρα μπορούμε να χρησιμοποιούμε καλύτερα τη διερμηνία, άρα δηλαδή οι ελεύθεροι συνεργάτες διερμηνής έχουν όχι μόνο δύο ημέρες εργασίας προσφορά, αλλά συμβάσεις τεσσάρων ημερών. Και για τις τέσσερις ε, ημέρες καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να προσλαμβάνουμε καλύτερους διερμηνείς και με τον τρόπο αυτό μειώνεται και το κόστος των εισιτηρίων και γιατί όχι και οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα το 2012 στον τομέα λοιπόν της μετάφρασης και της ε, διερμηνίας εξοικονομήσαμε συνολικά 24 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ε, να ε, μειωθεί η παροχή υπηρεσιών στους ευρωβουλευτές και αυτά θα επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. Στον τομέα της μετάφρασης αυξήθηκε η παραγωγικότητα των μεταφραστών κατά 50%. Αυτά τα στοιχεία είναι πολύ ενθαρρυντικά και καταδεικνύουν ότι υπάρχουν αποθέματα στη διοίκηση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς ε, να επιδεινώνεται η παροχή υπηρεσιών στους ε, συνεργάτες αλλά και στους, ε, στους ευρωβουλευτές με συγχωρείτε, αλλά και για τους συνεργάτες τους. Τώρα, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στις ερωτήσεις της εισηγήτριας της κυρίας Όρτης. Ευχαριστώ θερμά για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και με εκείνη και με τον εσωτερικό ελεγκτή. Επίσης, ευχαριστώ πολύ για τις ε, θετικές παρατηρήσεις ε, τις οποίες έκανα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τα συγκεκριμένα ερωτήματα ο υποχρεωτικός έλεγχος των ευρωβουλευτών στην είσοδο του Κοινοβουλίου. Επ' αυτού το Προεδρείο δεν άλαβε καμία απόφαση που να αλλάζει το ισχύον σύστημα. Προσπαθούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε τη σύγχρονη τεχνολογία και να ελέγξουμε στην πράξη ένα σύστημα το οποίο θα μας επιτρέπει ο Ευρωβουλευτής χωρίς να εμποδίζεται στην είσοδο να ελέγχεται η ταυτότητά του με το εξή σύστημα. η φωτογραφία του Ευρωβουλευτή με το που διασχίζει την πόρτα θα προβάλλεται σε μία οθόνη. Βέβαια το σύστημα αυτό δεν έχει ακόμα τελειοποιηθεί για να πω ότι θα το εφαρμόσουμε, αλλά ε, καταλαβαίνετε ότι αναζητούμε ένα σύστημα όπου οι ευρωβουλευτές ε, πράγματι να πιστοποιούνται ως ευρωβουλευτές και χωρίς αυτοί να παρεμποδίζονται κατά την είσοδό τους. Το δεύτερο ερώτημα που τέθη, ε, πότε ε, θα εφαρμοστεί αυτό το περίφημο zooming, δηλαδή το να υπάρχουν διάφορες ζώνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εισαγωγή αυτών των ζωνών αποφασίστηκε πέρυσι από το Προεδρείο και εμείς λάβαμε την εντολή να εφαρμόσουμε ένα ειδικό σχέδιο για τις διάφορες αυτές ζώνες. Αυτό λοιπόν το σχέδιο έχει κατατεθεί και προβλέπεται ότι το Κοινοβούλιο θα διαιρεθεί σε πέντε διαφορετικές ζώνες ασφαλείας και ε, θα έχουμε και κλιμακούμενα μέτρα ασφαλείας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι στον, στη ζώνη εκείνη που θα είναι προσπελάσιμη για όλους, εκεί ε, θα υπάρξει κάποια ελάφρυνση κυρίω κυρίως των επισκεπτών εφόσον γνωρίζουμε ότι στους ευαίσθητους τομείς μπορούμε να προσφέρουμε μεγαλύτερη ασφάλεια. Εσείς ε, ε, ρωτήσατε σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Πότε λοιπόν θα ληφθεί η σχετική απόφαση. Και εγώ πρότεινα στον Πρόεδρο αυτό το θέμα να το θέσει στην ημερήσια διάταξη του Προεδρείου για να ληφθεί η απόφαση την επόμενη Δευτέρα στο Στρασβούργο, δηλαδή την 4η Φεβρουαρίου. Προφανώς θα πρέπει να προηγηθεί συζήτηση, αλλά νομίζω έχουμε βάσιμες ελπίδες να πιστεύουμε ότι θα ληφθεί τελικά η απόφαση. Ο στόχος είναι οι αλλαγές που θα υπάρξουν στα κτίρια, αυτές οι αλλαγές να λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και του διαλύματος που μεσολαβεί ανάμεσα στις δύο κοινοβουλευτικές θητείες, έτσι ώστε να μην υπάρξουν εμπόδια για τους ευρωβουλευτές αλλά και για όλους τους άλλους χρήστες, που σημαίνει μετά το καλοκαίρι όταν θα έλθει ε, το το καινούριο κοινοβούλιο θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα κατάσταση. Τρίτον, όσον αφορά το θέμα της καντίνας, ε, το, το εστιατόριο. Ε, και εκεί έχουμε αρκετά προβλήματα, όπως και σε άλλους τομείς. Δηλαδή, τα κτίρια μας ή αν θέλετε η υποδομή μας δεν είχε προβλεφθεί για τον αριθμό των χρηστών στον οποίο εντωμεταξύ έχουμε φτάσει. Παράδειγμα, ε, το είπα αυτό όταν ρωτήθηκα ξανά για το εστιατόριο. Πριν από 10 χρόνια είχαμε 1,4 εκατομμύρια χρήστες του εστιατορίου. Τώρα 3,7 εκατομμύρια χρήστες του εστιατορίου, που σημαίνει υπερδιπλασιασμός, χωρίς όμως ε, να αυξηθεί ουσιαστικά το προσωπικό του εστιατορίου, με μικρές βελτιώσεις. Άρα δηλαδή η υποδομή επιβαρύνεται τα μάλα. Το ίδιο ισχύει και για τους ανελκυστήρες. Έχουμε ανελκυστήρες οι οποίοι μετακινούνται πάνω από 2.000 φορές την ημέρα. Αυτό λοιπόν σημαίνει τεράστια επιβάρυνση. Και γιατί ε, η επιβάρυνση προκύπτει ε, μάλλον η επιβάρυνση προκύπτει διότι έχουμε πάρα πολλούς ε, μετακινούμενους ε, ανθρώπους στο κτίριό μας που είναι και επισκέπτες και συνεργάτες. Όσον αφορά στους επισκέπτες ισχύει το εξής. σήμερα οι επισκέπτες, όπως είχε αρχικά προβλεφτεί, δεν μετακινούνται μόνο σε ένα συγκεκριμένο τομέα, όπου να έχουμε ειδικό εστιατόριο για αυτούς, ειδικέ αίθουσε, έστω ε, να μπορούν να μπουν και στην Ολομέλεια. Βλέπουμε ότι πάρα πολλές ομάδες επισκεπτών ε, μετακινούνται παντού στο Κοινοβούλιο και στο κύριο κτίριο. Όταν λοιπόν έχουμε ομάδες επισκεπτών που περιμένουν τον ανελκυστήρα, καταλαβαίνετε ότι οι ανελκυστήρες αυτοί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεύτερον, στον τομέα των συνεργατών εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε την εξή ε, κατάσταση. Ε, έχουμε ένα γραφείο για του ευρωβουλευτέ και ένα γραφείο για του συνεργάτε. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει τρει συνεργάτε και μερικέ φορέ και άλλου τρει μαθητευόμενους που κάνουν πρακτική άσκηση. Δηλαδή ε, σε 70 τετραγωνικά μέτρα πάνω από 7 άτομα. Αυτή λοιπόν η κατάσταση για μένα είναι απαράδεκτη και δεν νομίζω ότι είναι πολυτέλεια το να σκεφτούμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Κάναμε μια ε, μελέτη συγκρισιμότητας με το Γερμανικό Κοινοβούλιο, το Bundestag. Το Bundestag είναι το κοινοβούλιο του μεγαλύτερου κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρετε κάτι, τώρα το Bundestag πρόκειται να προσφέρει τέταρτο γραφείο γραφείο στους βουλευτές, για αυτούς και τους συνεργάτες τους. Εμείς έχουμε δύο γραφεία, παρότι συνεδριάζουμε περισσότερο από το Bundestag, διπλάσιος αριθμός των συνεδριάσεων των δικών μας. Ε, εμείς ε, ε, έχουμε και εκτελεστική εργασία. Πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει και ελπίζω κατά τη νέα θητεία να μπορέσουμε να επιτύχουμε βελτιώσεις. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ε, αυτή τη στιγμή στη διοίκηση προβαίνουμε ε, σε κάποιες βελτιώσεις. Επανέρχομαι στο θέμα του εστιατορίου. Πρότεινα στον πρόεδρο το θέμα αυτό να το συζητήσουμε στις περίφημες away days, εκεί που συνεδριάζει δηλαδή το Κοινοβούλιο σε κεκλεισμένο των θυρών, μετά από τέσσερις εβδομάδες που θα συνεδριάσουμε. Βεβαίως δεν θα καταστεί δυνατόν εκεί να ληφθεί η τελική απόφαση, όμως το θέμα θα συζητηθεί διεξοδικά και χρειαζόμαστε κάποιες εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα μας επιτρέψουν να καταλήξουμε στην τελική λύση. Πάω τώρα στο σπίτι της ευρωπαϊκής ιστορίας. Η χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος ε, ρυθμίζεται σε ένα business plan ε, το οποίο έχει συμφωνηθεί από την Επιτροπή Προπολογισμών και από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τηρούμε απαρέγκλητα τις προποθέσεις αυτού του προγράμματος. Εν τω μεταξύ έχουμε τις ε, διάφορες προσφορές για την ανέγερση αυτού του κτηρίου και κινούμεθα μέσα στα κονδύλια που προβλέπονται στον προπολογισμό. Από πλευράς χρονοδιαγράμματος είμαστε καλά. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι την άνοιξη του 2014 ε, θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα κατασκευής και κατόπιν τίθεται το ερώτημα μήπως θα μπορούμε να το ανοίξουμε έστω εν μέρη αυτό το σπίτι της ιστορίας. Υπήρξαν κάποιες συζητήσεις ανάμεσα στην Επιτροπή Προπολογισμών και τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος λοιπόν έκρινε ότι δεν πρέπει να γίνει μια μερική εγγενίαση το 2014 αλλά να περιμένουμε να ολοκληρωθεί το εσωτερικό του κτηρίου, ο εξοπλισμός του και αυτό σημαίνει ότι η οικονομική επιβάρυνση ε, θα υπάρξει για ένα περαιτέρω έτος. Και αυτό σημαίνει ότι το κτίριο έτοιμο πλέον στην τελική του μορφή ε, θα είναι ε, το 2015. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεσμεύτηκε γραπτά με επιστολή του κυρίου Μπαρόζο να προσφέρει οικονομική χρηματοδότηση για τις τρέχουσες δαπάνες. Εμείς προσφέρουμε ε, την κατασκευή και ένα μέρος των ε, τρεχουσών δαπανών και το υπόλοιπο θα πληρώνεται από την Επιτροπή. Άρα δηλαδή η Κομισιόν δεσμεύεται πριν από το καλοκαίρι του 2014 ε, όταν θα κάνει την προσφορά της για τον προπολογισμό να αναφέρει συγκεκριμένα ποιο θα είναι το ποσό ε, με το οποίο θα συμμετέχει. Πάντως ε, σας είπα ότι τα επίσημα γένεια θα γίνουν το φθινόπωρο του 2015. Βεβαίως δεν έχουμε ακόμα κάνει εκτίμηση κόστους για το 2015. Ε, πάντως να το ξέρετε, το 2015 θα προκύψουν αυτές οι δαπάνες και βεβαίως και το 2016. Αυτό θα το συζητήσουμε με την Κομισιόν για να δούμε ε, όπως σας είπα, ε, ποιο θα είναι το δικό της το ποσοστό συμμετοχής. Όσον αφορά τώρα το θέμα των συνεργατών, σας είπα ότι δεν χρειάζεται να προσλάβουμε νέους υπαλλήλους για το σπίτι της ευρωπαϊκής ιστορίας, γιατί θα καλύψουμε τις ανάγκες μέσα από μετατάξεις. Ε, είμαι βέβαια πεπισμένος ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ε, συνεργατών θα πρέπει να είναι με συμβάσεις έργου συμβάσεις έργου. Γιατί? Ε, διότι χρειαζόμαστε ε, επιγόντως ε, τεχνοκράτες, ειδικού γνώστες, μουσιολόγους. Αυτούς χρειαζόμαστε για το σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Όμως μουσιολόγους δεν έχουμε εδώ στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτοί υπάρχουν στα 27 κράτη-μέλη. Επιθυμούμε λοιπόν και η γνώση τους να είναι επίκαιρη. Άρα δηλαδή ε, αυτοί να προσληφθούν για κάποια έτη. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε ένα μείγμα υπαλλήλων από συμβασιούχους αλλά και από άλλους ε, μόνιμους ε, υπαλλήλους οι οποίοι θα εργάζονται για το πρόγραμμα αυτό. Όσον αφορά τώρα το θέμα του διαγωνισμού ο κύριος Κέλβιν θα αναφερθεί εντός ολίγου στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι επιτύχαμε σημαντική πρόοδο με τον παλιό νέο δημοσιονομικό κανονισμό όπως αποκαλείται δεν υπάρχει πλέον ε, συγκεντρωτικό σύστημα αλλά αποκεντρωτικό που σημαίνει ότι υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές ε, οι οποίες ε, υπάγονται στις αρμοδιότητες του εκάστοτε ε, authorizing officer. Ε, βεβαίως και πρέπει να τηρούνται κάποια πρότυπα ποιότητας. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτές οι προδιαγραφές ε, ποιότητας να ισχύουν. Και για το λόγο αυτό με το Procurement Forum καταλήξαμε ε, σε κάποιες αποφάσεις, ε, σε κάποιες εξαιρετικές ε, αποφάσεις που θα πρέπει να λαμβάνονται. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι όχι ότι χάνει τις αρμοδιότητες του ο εκάστοτε authorizing officer, αλλά μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να καταφεύγει σε τεχνογνωσία. Αυτή είναι μια απόφαση την οποία έλαβα το, κατά το τέλος του 2011 και έκτοτε εφαρμόζεται. Όσον αφορά τις μήνυ ολομέλειες, μπορώ να σας πω ότι το 2013 δεν θα λάβουν χώρα μίνι ολομέλειες στις Βρυξέλλες. Άρα δηλαδή ε, για ολομέλειες ε, έχουμε προβλέψει μόνο τις ολομέλειες στο Στρασβούργο. Και ε, ποιος είναι ο λόγος? Είναι η κατάσταση του ημικυκλίου στις Βρυξέλλες που καθιστά απαραίτητο να προβλέψουμε μια νέα μεταλλική φέρουσα κατασκευή που θα σταθεροποιεί τη στέγη. Αυτά θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2013. Άρα δηλαδή, αν λέγαμε τώρα ότι θα προσπαθήσουμε ε, να έχουμε ας πούμε μείνει ολομέλεια το Νοέμβριο του 2013, ενδέχεται ε, βραχυπρόθεσμα να χρειαστεί να αναβάλουμε κάτι τέτοιο. Αυτό όμως δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί τους ευρωβουλευτές που πρέπει να προγραμματίζουν μακροπρόθεσμα τα ταξίδια τους. Ε, όσον αφορά την μεταλλική φέρουσα κατασκευή, ε, αυτό το σύστημα επέλεξε το Προεδρείο. Δηλαδή οι ξύλινοι δοκοί παραμένουν, αλλά αυτή αυτοί οι ξύλινοι δοκοί συμπληρώνονται με μεταλλικά στοιχεία και αυτή η φέρουσα κατασκευή αρκεί για τη στήριξη της οροφής. Αν θέλετε δηλαδή η παλιά φέρουσα κατασκευή, οι δοκοί συμπληρώνονται ολοκληρώνονται και αυτές, αυτή η μεταλλική πλέον δοκή ε, πρέπει να κατασκευαστούν με μία απόλυτη ακρίβεια, χιλιοστού. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι χρειαζόμαστε χρόνο. Αυτό όμω μας επιτρέπει επίσης ε, να αφήσουμε την οροφή, τη στέγη ως έχει. Δεν χρειάζεται να την απομακρύνουμε. Έχουμε επιλέξει αυτή τη λύση ε, των μεταλλικών δοκών. Εσείς ε, αναφερθήκατε επίσης ε, στο ημικύκλιο του Στρασβουργού πριν από ένα χρόνο και εκεί είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ποιες ήταν οι συνέπειες αυτού. Μπορώ να σας πω ότι όταν εγώ ανέλαβα το αξίωμά μου 16 Μαρτίου του 2009 συγκεκριμένα στις 18 Μαρτίου του 2009 κατέθεσα πρόταση στο Προεδρείο για την αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης εκτηρίων. δηλαδή μόνος μετά από δύο ημέρες. Και αυτή η αναδιάρθρωση προέβλεπε ότι θα έχουμε μια ειδική μονάδα για τη συντήρηση ε, των κτηρίων στο Στρασβούργο. Ε, να την σπάσουμε τη Γενική Διεύθυνση. Νέα κτίρια, μονάδα συντήρησης, ε, γιατί όταν μιλάμε για ένα εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα, καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε τεχνογνωσία για τη συντήρηση. Τότε η Επιτροπή Προεπολογισμών προς τη μήν ήταν πρόθυμη να διαθέσει τα απαραίτητα κονδύλια. 48 θέσει εργασία για τρία χρόνια και ένας αρκετά ένα αρκετά σημαντικό ποσό εκατομμυρίων που μας επέτρεψε να καταφύγουμε και στις γνώσεις εξωτερικών συνεργατών. Καταλήξαμε λοιπόν σε ένα πρόγραμμα το οποίο ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήρηματα τη συντήρηση των κτηρίων. Χάρη λοιπόν αυτού του προγράμματος μπορέσαμε να καλύψουμε τις ζημιές του ημικυκλίου στο Στρασβούργο. Αν δεν είχαμε αλλάξει τη Γενική Διεύθυνση και αν δεν είχαμε λάβει τα επιπρόσθετα κονδύλια από την Επιτροπή Προπλογισμών και από την Ολομέλεια, δεν θα είχαμε ανακαλύψει τη ζημιά και δεν θα μπορούσαμε να... και επίσης επειδή θα προέκυπτε και αυτό το πρόβλημα στις Βρυξέλλες έτσι κι αλλιώς, δεν θα μπορούσαμε να καλύψουμε αυτό το σύνολο της ζημιάς, ε, πόσο μάλλον ε, όλα αυτά που θα υφίσταντο οι συνεργάτες του Κοινοβουλίου. Εν ολίγης, οι αλλαγές που έγιναν τα τελευταία χρόνια στον τομέα της συντήρηση κτηρίων, το ότι μπορέσαμε να έχουμε ε, τεχνοκράτες, ειδικού στο Κοινοβούλιο, του Κοινοβουλίου υπαλλήλου αλλά και εξωτερικούς, αυτά τα χρήματα που διατέθησαν για αυτούς αποδείχθηκαν χρήσιμα. Όσον αφορά το ερώτημα που θέσατε σχετικά με τα email, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπάρχει ένα ε, πρόβλημα ε, που ε, προέκυψε από ένα λογισμικό antivirus που προσέφερε η Microsoft. Παρόλα αυτά, λύθηκε το πρόβλημα, αλλά υπάρχουν άλλα μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί όλο και περισσότερο φτάνουμε στα όρια των δυνατοτήτων μας. Ο όγκος των mail και ο όγκος της ε, κινητής επικοινωνίας τα τελευταία χρόνια εξεράγει. Μιλάμε για μια έκρηξη επικοινωνίας και δεν είχαν προβλεφθεί τα συστήματά μας για αυτά τα μεγέθη. Έπρεπε λοιπόν να προσαρμοστούν. Υπάρχουν όμως και θέματα που αφορούν και στον τρόπο συμπεριφοράς. Παραδείγματο χάρη γνωρίζουμε, έχουμε ένα χρήστη, ο οποίος στο δικό του το σύστημα mail αυτός και μόνο διαθέτει 90.000 επαφές. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όταν έχει κανείς 90.000 επαφές, ένας και μόνο, ε, τι πρέπει να κάνει οι άλλοι. Αυτό λοιπόν οδήγησε στο να υπάρξει πρόβλημα, γιατί με τον τρόπο αυτό το σύστημα φτάνει στα όρια του. Βεβαίως και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Νομίζω όμως ότι και εμείς ε, πρέπει να δείξουμε μια αυτοσυγκράτηση στην ηλεκτρονική μας, ε, στα ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και την επαφή μας. Ε, κατόπιν, το 2011 μπαίνω σε πολύ πιο συγκεκριμένα θέματα που άπτονται της απαλλαγής όπως κάθε χρόνο. Απαντήσαμε σε όλες τις ερωτήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την απαλλαγή με τη στενή έννοια και υπάρχουν άλλα θέματα ευρύτερα που αφορούν τη διαχείριση. Όλα αυτά τα ερωτήματα τα επαντήσαμε, αλλά όσον αφορά τα πολύ πιο ε, συγκεκριμένα συστήματα του 2011, επισημαίνω και πάλι τα απαντήσαμε και αυτά. Έρχομαι τώρα στο ταξιδιωτικό γραφείο. Το ταξιδιωτικό γραφείο νομίζω το θέμα το γνωρίζετε. Βεβαίως Όσον αφορά τα εισιτήρια, όταν ναι, κανείς ένας ε, φυσιολογικός χρήσης λέει θα αγοράσω ένα εισιτήριο οικονομικής θέσης ή business class. Ε, προφανώς ε, υπάρχουν ε, διάφορες τιμές εισιτηρίων. Έχω δει διάφορες τιμές εισιτηρίων και για την business και για την οικονομική θέση. Και ως αγοραστής στο διαδίκτυο δεν μπορεί κανείς να τα ξέρει όλα και να ξέρει όλες τις τιμές. Εμείς παρόλα αυτά αποφασίσαμε, επειδή προσπαθήσαμε να μειώσουμε το κόστος ταξιδίων κατά 5%, καλέσαμε το Γραφείο Ταξιδίων να κάνει ουσιαστικότερες έρευνες για τις τις ε, καλύτερες τιμές ε, και μπορέσαμε να εξοικονομήσουμε 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Ε, ελπίζουμε λοιπόν το 2013, προφανώς και εδώ εξαρτώμεθα από το πνεύμα συνεργασίας που θα επιδείξει το ταξιδιογραφείο, ελπίζουμε να υπάρξει και άλλη εξοικονόμηση. Βεβαίως εντωμεταξύ υπάρχει και ένας διαγωνισμός που αφορά όλα τα όργανα και ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα προκύψουν βελτιώσεις. Έρχομαι τώρα στο ε, καταστατικό των υπαλλήλων. Η αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα θετική. Γνωρίζουμε, ε, γνωρίζετε μάλλον ότι με το παλιό σύστημα προέκυψαν πάρα πολλά προβλήματα. Κυρίως όσον αφορά το καθεστώς των συνεργατών. Οι συνεργάτες είχαν συμβάσεις ε, απαράδεικτες. Σε μεγάλο βαθμό δεν είχαν κοινωνική ασφάλιση. Γι' αυτό λοιπόν τελήσαμε να βελτιώσουμε την κατάσταση κυρίως στα κράτη-μέλη. Και με τον τρόπο αυτό αυτό μπορέσαμε να προσλάβουμε ποιοτικά καλύτερους ε, βοηθούς συνεργάτες. Ο προϋπολογισμός, το ύψος του προϋπολογισμού παρέμεινε το ίδιο. Το 2009 υπήρξε μία ε, προσαρμογή προς τα πάνω δύο φορές λόγω της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. αυτό προφανώς είχε και κάποιο, κάποια διοικητική επιβάρυνση, αλλά άξιζε τον κόπο. Όσον αφορά τα intergroups, η τελευταία σας ερώτηση. Αυτά εμπίπτουν στη διακριτική ευχέρεια της πολιτικής ομάδας. Δηλαδή, η ίδια η πολιτική ομάδα, αν θέλει να στηρίξει αυτά τα intergroups, η πολιτική ομάδα μπορεί να προσφέρει αίθουσα και διερμηνείς που δεν χρειάζεται η ίδια. Άρα δηλαδή δεν προκύπτει επιπρόσθετο κόστος ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρία Συγγήτρια, ελπίζω να απάντησα ικανοποιητικά στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Γραμματέα από αυτά που μα είπατε. Κατέστη σαφέ. Ε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι και θα παραμείνει εργοτάξιο. Καλή αυτή η εικόνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ότι απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματά μας και πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση θα ήθελα να παρακαλέσω τον εσωτερικό ελεγκτή, τον κύριο Γκάλβιν, να μας πει και αυτός ε, την δική του την άποψη. Κύριε Γκάλβιν, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Uh, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε να ε, παρουσιάσω την ετήσια έκθεσή μου για το 2011. Στις 26 Ιουλίου έκανα κάποιες προσαρμογές ε, μετά από, μετά από διαβούλευση με τον Γενικό Γραμματέα γιατί μου ζητάτε μια ειδική έκθεση που αναφέρει τον αριθμό των εσωτερικών ελέγχων που γίνονται και το είδος ε, των ελέγχων αυτών, όπως επίσης και τις την, τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει αυτών των, των εκθέσεων. Οπότε σας, βλέπω, σας δείχνω το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων των εσωτερικών ελεκτών του 2011. Βλέπουμε λοιπόν ότι βάσει επαγγελματικών προδιαγραφών κάθε χρόνο υπάρχει ένα ετήσιο πρόγραμμα βάσει της αξιολογικής αξιολόγηση κινδύνου ολόκληρου του ε, οργανισμού. Και ο βασικός στόχο είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στο IAS να δώσει προτεραιότητες ε, στις, ε, τομεί υψηλού κινδύνου που χρήζουν μεγαλύτερη προσοχή. Το 2011 οι εσωτερικοί έλεγχοι εστιάστηκαν κυρίως στις μεσοπρόθεσμε στρατηγικέ για τις δημόσιες προμήθειες, την τεχνολογία των πληροφοριών, όπω επίση και τι δαπάνε για το προσωπικό και επίσης για τη συνέχιση των ε, ε, συμπεφωνημένων ε, προγραμμάτων και των μέτρων από τους προηγούμενους ελέγχους. Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω την κατάσταση του 2011 σε σχέση με τις δημόσιες προμήθειες. Ε, ένας από τους βασικούς στόχους είναι, η είναι το αποκεντρωμένο περιβάλλον εσωτερικών ελέγχων. Η συνολική πρόοδος υπήρχε σε μερικούς τομείς, χρειάζεται όμως περισσότερη ε, βελτίωση στην κεντρική ε, διαχείριση. Πρέπει να υπάρξουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάλυση και τη διαχείριση κινδύνου, την καταγραφή των εσωτερικών ελέγχων, όπως επίσης και τη βελτίωση της ε, ε, ομαλοποίησης του προϋπολογισμού. Ε, σε συνέχιση από το 2010 έχουμε βρει κάποια πρόοδο που έχει σημειωθεί σε κάποιους από αυτούς τους τομείς, στον τομέα ας πούμε των δημοσίων προμηθειών. Βασικό θέμα ήταν αφορούσε τη Γενική Διεύθυνση ITEC για την καινοτομία και την τεχνολογία των πληροφοριών βρήκαμε ότι υπήρξαν κάποιες σοβαρές αδυναμίες. Ε, έγιναν ε, έλεγχοι των βασικών συμβάσεων για τις υπηρεσίες ε, τετραετούς περίοδου για 250 εκατομμύρια ευρώ και βρήθηκαν κάποιες, παρατυπίες γενικότερα ε, στις συμβάσεις αυτές, κάτι το οποίο είχε ε, ε, σοβαρά, σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τις συμβάσεις αυτές. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με το ευρύτερο σχέδιο δράσης. Ούτως ή άλλως είχαν αρχίσει κάποιες αναθεωρήσεις από, για τη διαδικασία του 2008 για να μην ξαναυπάρξουν τέτοιου είδους προβλήματα στην ανανέωση της διαδικασίας αυτής στην Γενική Διεύθυνση ITEC. Έγινε ένας έλεγχος που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της αναλογίας των off-site ε, υπηρεσιών ε, τεχνολογίας πληροφοριών με μεθόδους εφαρμογής, ε, με προσυμφωνημένα αποτελέσματα για να μπορούμε να πηγαίνουμε σε περισσότερες, με, σε, να, να φτάνουμε πιο συχνά σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης. Επίσης βρήκαμε ότι υπήρχε μία ανάγκη βελτιώσεων σε, σε τομείς που υπήρχαν σοβαρά προβλήματα, βελτίωση των διαδικασιών, αξιολόγηση των προσφορών, και τον ε, προγραμματισμό των εσωτερικών ελέγχων σε σχέση με τις προμήθειες. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, είχαμε ένα σχέδιο δράσης 9, σημείων μέχρι το τέλος του 2012 ε, έχουν ήδη γίνει ε, θετικές ενέργειες ε, με μεγάλη αναδιοργάνωση του εσωτερικού οικονομικού συστήματος από τον Ιανουάριο του 2012. Επίσης, η IAS παρακολούθησε τη διαδικασία προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης ITEC που είχε ξεκινήσει από το 2009 και δόθηκε η δυνατότητα στις, ε, στον εσωτερικό έλεγχο να κλείσει τις οκτώ βασικές δράσεις που είχε εντοπίσει. Όσον αφορά τώρα τις δαπάνες του προσωπικού, είδαμε ε, τη μισθοδοσία και διαπιστώσαμε ότι το περιβάλλον ελέγχου και οι δραστηριότητες ελέγχου στις ε, ε, πληρωμές ε, συνάδουν με τους στόχους και επίσης υπάρχει κάποια συνέπεια. Η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού συμφώνησε να ενισχύσει περισσότερο τη διαδικασία ελέγχου και διαχείρισης για τη βελτίωση της αξιοποίησης των δεδομένων για το προσωπικό, όπως επίσης και του συστήματος διαχείρισης του προσωπικού για τη βελτίωση της ε, αποτελεσματικότητας κοινοποίηση των αποφάσεων. Επίσης, όσον αφορά τον ε, παράγοντα από πολλαπλασιασμού των ε, μισθών που είχε αναφερθεί στην μεταρρύθμιση του εσωτερικού κανονισμού του 2004, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με τα προβλεπόμενα μεταβατικά μέτρα και την προσέγγιση που έχουν ακολουθήσει άλλα όργανα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κοινοβούλιο αναφέρομαι γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει κάποια οικονομικά πλεονεκτήματα σε κάποια μέλη του προσωπικού που είχαν προσληφθεί πριν από το 1η Μαΐου 2004. Το συμπεφρονημένο σχέδιο δράσης ε, δείχνει ότι πρέπει να γίνουν κάποιες προσπάθειες βελτίωσης ε, της ε, διαδικασίας για να ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες ενός κινδύνου του πολλαπλασιαστικού παράγοντα ε, να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα ε, στις πληρωμές. Να δούμε δηλαδή σε ποιο βαθμό κάποια διορθωτικά μέτρα μπορούν ακόμη να ληφθούν για να ε, περιοριστεί, να διορθωθεί το οικονομικό ε, αποτέλεσμα ε, των δραστηριοτήτων αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το 2012 λοιπόν προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες διορθώσεις, μία από τις οποίες ήταν η συνέχιση των προσπαθειών των επιδομάτων για τους συνεργάτες, ένα σχέδιο 12 μέτρων, είδαμε ότι υπήρξε πρόοδο σε σχέση με την αντιμετώπιση των προβλημάτων των τομέων κινδύνου και ο εσωτερικός έλεγχων έκλεισε από τις 33 από τις 36 ε, ε, περιπτώσεις ε, που είχε ελέγξει. Λοιπόν, κάποια συστημικά προβλήματα είχαν αντιμετωπιστεί. Είδαμε επίσης ότι τα εφαρμοστικά μέτρα για το καθεστώς των βουλευτών και τα σχετικά μέτρα που είχαν προτείνει, είχε προτείνει η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ε, είχαν βελτιώσει πολύ το ελεγκτικό περιβάλλον. Τρεις τομείς επίσης σε σχέση με τις ανοιχτές δράσεις ήταν μια, ε, ε, εξακολουθούσαν να εκτίθενται σε κίνδυνο. Μπορεί οι συνέπειε να είναι μικρέ, όμω μπορεί να υπάρξει πολύ μεγαλύτερο ε, πολύ μεγαλύτερος κίνδυνο. Πρέπει να υπάρξει ένα νέο σχέδιο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ε, ελέγχων που γίνονται από τους επικεφαλείς των πληρωμών. Το 2011 το IAS επίσης παρακολούθησε την ε, εξέλιξη της διαδικασίας των πληρωμών και της προόδου που έχει σημειωθεί. Στην αρχή είχαμε πει ότι θέλουμε μεγαλύτερη αποκέντρωση της διαδικασίας με ενίσχυση των ελέγχων και των κατευθυντηρίων γραμμών, βελτίωση επίσης των χρόνων πληρωμών, όπως επίσης καλύτερη εφαρμογή ε, του σχεδίου εφαρμογής. Ήταν βέβαια ε, μικρό το ποσοστό της εφαρμογής, Πρώτον, ε, η μείωση των χρόνων πληρωμών από το 2008 και δεύτερον, η απόφαση που ελήφθη τον Ιούλιο του 2011 για τη δρομολόγηση ενός προγράμματος ε, εξυγχρόνησης του συστήματος ε, πληροφόρηση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Για αυτά τα δύο στοιχεία θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε παρά το γεγονός ότι θεωρούμε ότι ο κίνδυνος αυτού του δύο τομείς είναι μικρός. Υπήρχε επίση ένα σχέδιο δράση ε, για τις, ε, τη βελτίωση της διαδικασίας ε, στέγασης και ακινήτων. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και ειδικότερα η ενίσχυση των δομών μπορεί να χρειαστεί περισσότερη δράση σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα από αυτόν που είχε διαφανεί στην αρχή. Επίσης, Έχουμε ένα πρόγραμμα που εξηγεί ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι των υψηλότερων δυνατών προδιαγραφών και οι εσωτερικοί ελεγκτές ε, ε, κατήρτισαν ένα πρόγραμμα ε, που ακολουθήθηκε το 2011 βάσει των δράσεων που είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των εκθέσεων σαν αυτή που σας παρουσιάζω τώρα. Το αποτέλεσμα της έκθεσης για το 2011 δείχνει ότι έγιναν σημαντικές βελτιώσεις στο ρυθμιστικό και ελεγκτικό περιβάλλον που επιβεβαιώθηκε από το 2011, κάτι το οποίο προέκυψε από την αλλαγή που έγινε το, 2011, ε, το 2008. Συγγνώμη. Αυτό δείχνει ότι ε, η μεταρρύθμιση των ε, συστημάτων μας όντως μπορεί να επιφέρει αλλαγές και βελτίωση κάτι το οποίο φαίνεται από την ειδική μας έκθεση και δείχνει ε, πραγματικά πόσο καλύτερα μπορούμε να εντοπίζουμε τους κινδύνους. Επίσης, ο εσωτερικός ελεγκτής επιβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε πρόβλημα ανεξαρτησίας, ούτε παρεμπόδιση ε, της δουλειάς των εσωτερικών ελεγχών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό πάνελ, όπως επίσης και το Γενικό Γραμματέα για την υποστήριξή του και ε, τον εισηγητή για την κατανόησή του και θα ήθελα επίσης ε, να πω ότι ήταν εξαιρετική η συνεργασία μας με όλα τα τμήματα το 2011. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γκάλβιν, για την ε, εκθεσή σας ε, και θα ήθελα τώρα να καλέσω τους ε, συναδέλφους να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους μετά από αυτά που άκουσαν. Ο να φτιαχτούν από τους Σοσιαλδημοκράτες, Ντέρικ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ντέρικ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή, ε, ε, τον κύριο Πιτέλα και τον Γενικό ε, Γραμματέα θα γνωρίζω ότι είμαι ο εισηγητής για το προπολογισμό 2013, οπότε γνωρίζω ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδος ε, ως προς, προς τον εντοπισμό των ε, οικονομιών που μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ορισμένα πράγματα ήδη αναφέρθηκαν σε σχέση με τα επιδόματα ε, και τα έξοδα των βουλευτών. Έχουν γίνει λοιπόν κάποιες σημαντικές προσπάθειες, υπάρχει πρόοδος και θα δούμε πώς μπορούμε, όταν κάνουμε οικονομίε, θα το κάνουμε με έναν τρόπο που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην αποτελεσματικότητα του Κοινοβουλίου ούτε των Ευρωβουλευτών. Οπότε στο μέλλον νομίζω ότι χρειάζεται να, να φύγουμε από αυτή τη διαδικασία περικοπών για τους ευρωβουλευτές και να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε διαφορετικές οικονομίες που θα μας βοηθήσουν στο μέλλον. Ξέρω ότι έχει ξεκινήσει κάποια δουλειά προς αυτό και έχουν αναφερθεί κάποιες δυνατότητες όπως για παράδειγμα στις γραπτές απαντήσεις σας λέτε κατά τη διάρκεια της πράσινης εβδομάδας ε, μπορούμε να εξοικονομήσουμε 9.000 ε, ευρώ. 900.000 ναι. ευρώ. Αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ίσως ε, θα έπρεπε να ενημερώσετε τους ευρωβουλευτές για τη δουλειά αυτή που ε, συζητιέται με την ΕΚΟΣΟΚ και με την Επιτροπή Περιφερειών, γιατί πιστεύω ότι είναι ένας τρόπος να προχωρήσουμε, να έχουμε μια κοινή δουλειά ερμηνείας, ε, ε, μια κοινή δουλειά διερμηνίας και μεταφράσεων ε, με, τους, ε, με τα όργανα αυτά για να μπορούμε, μπορέσουμε να προβούμε στις οικονομίες που θέλουμε ή ας πούμε ή ε, βιντεοδιασκέψεις και αυτό είναι, είναι ένας πολύ καλός τρόπος ίσως έχουμε ήδη ξεκινήσει αλλά θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα γιατί νομίζω ότι έτσι θα κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη οικονομία τα γλωσσικά μαθήματα για το προσωπικό Κάποιοι πηγαίνουν στη Νότια Γαλλία ή στη Μόσχα για μαθήματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εξετάσετε αυτό και να βρείτε έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο για αυτά τα γλωσσικά μαθήματα ε, του προσωπικού. Και κάτι ακόμη κάποια χρήματα τα οποία ε, υποαξιοποιούνται, δεν χρησιμοποιούνται καθόλου. Ε, ίσως στο τέλος αυτής κάθε χρονιάς ε, να τα συγκεντρώνουμε και νομίζω να ξέρουμε ποια χρήματα δεν χρησιμοποιήθηκαν, γιατί έτσι θα ήταν πολύ καλύτερος και αποτελεσματικότερος ο προπολογισμό μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και ευχαριστώ πολύ που δεν χρησιμοποίησε και πάρα πολύ χρόνο. Δεν θέλω να σα περιορίσω, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό και η συζήτησή μα είναι πολύ σημαντική. Αλλά έχουμε και κάτι να συζητήσουμε από τη χθεσινή ημερήσια διάταξη. Οπότε θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε την συζήτησή μα για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ την κυρία Ορτής ε, και τον Αντιπρόεδρο και τον κύριο Κλάους Βέλλο αλλά και τον ε, κύριο Μουραγκούθα θα ήθελα να πω τα, τα εξή. Σε ό,τι αφορά τη σκεπή του Μητυκλίου να ρωτήσω πως πέραν των όσων ανέφερε, τα οποία τον συγχαίρω και συμφωνώ απόλυτα, χρειαζόμαστε μια υπηρεσία συντήρησης, ε, αυτό είναι προφανές, αλλά μιλήσαμε και για την ευθύνη των ε, επιχειρήσεων, των κατασκευαστών, των μηχανικών, διότι ε, προφανώς ότι χρειάζεται αποζημίωση, που έγιναν κακοτεχνίες, έχει δικαίωμα λοιπόν το Κοινοβούλιο να λάβει αυτές τις αποζημίωσεις. Επίσης το ζήτημα της σύγκρισης με άλλα κοινοβούλια. Είπατε πως έγινε μια σύγκριση με το Bundestag για να δείτε τι γίνεται εκεί. Θα μπορούσαμε κι εμείς ε, να βρούμε έναν παρα, παρα, παραπλήσιο τρόπο να λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες ε, και κάτι ακόμα. Ε, μιλήσατε για, εξωτερήκευση, για εσωτερήκευση σε ό,τι αφορά τους υπάλληλους ασφάλειας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και να σας ρωτήσω το εξής. Για όλους αυτούς τι έχετε προγραμματίσει αναφορικά με την είσοδο το κοινοβούλιο των, αυτών των υπαλλήλων δηλαδή. Προβλέπετε μια συνεχής εκπαίδευση, κατάρτιση αυτού του προσωπικού, διότι είναι κάτι το οποίο διαφοροποιείται από την ε, εκπαίδευση του προσωπικού άλλων επιχειρήσεων το θέμα τώρα των ε, διαδικτύου που χρησιμοποιούν οι αντιπροσωπείες. Ξέρω ότι είναι περίπλοκο το ζήτημα, μέρα με τη μέρα βελτιώνεται, αλλά θα μπορούσαν ε, και οι αντιπροσωπείες να κάνουν μια προσπάθεια βελτίωσης όταν πρόκειται να διαδώσουν την πληροφορία τόσο στο εσωτερικό σου και στο εξωτερικό του οίκου μας. Ο κύριος Ρούμπιχ έχει το λόγο και μετά ο κύριος Ντεγιούγκ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Και θα ήθελα να συγχαρώ το Γενικό Γραμματέα για τις ε, αλλαγές που έκανε στο Κοινοβούλιο και οδήγησαν σε θετικές εξελίξεις ε, το Παρλαμεντάριο με το Κέντρο Επισκεπτών, πολύ επιτυχημένο. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι έχει βελτιωθεί κατά πολύ η επικοινωνία μας με τους υπόλοιπους. Να σας πω και το εξής. Ε, το Αυστραλιανό Κοινοβούλιο έχει ένα σύστημα όπου μπαίνει κανείς, ε, μετριέται το κεφάλι του ε, και από το μέγεθος το σύστημα δίνει περαιτέρω στοιχεία ο υπάλληλο ο ελεγκτής ε, βλέπει τη φωτογραφία του Ευρωβουλευτή. Άρα βλέπετε υπάρχουν συστήματα που μπορείτε λιγάκι να τα δείτε. Τώρα, όσον αφορά τις δαπάνες για τη διερμηνία, εγώ προτείνω κυρίως στα ταξίδια εκτός των οργάνων του Κοινοβουλίου διερμηνείς ε, να προσφέρονται μόνο εφόσον το ζητήσει ο Ευρωβουλευτής. Αυτή τη στιγμή ε, οι διερμηνείς ε, έχουν ε, ε, γλώσσες που προσφέρουν, άλλοι θετικά, ε, άλλοι οι ευρωβουλευτές μπορούν να ακούσουν μερικές φορές τη γλώσσα τους, άλλες να μιλήσουν μερικές φορές και τα δύο, αλλά λέω αυτό να γίνεται μόνο εφόσον το ζητήσουν. Κατά τα άλλα, είπατε ότι ο σχεδιασμός των ευρωβουλευτών είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, κατά κανόνα, εμείς ξεκινάμε τον προγραμματισμό μας για μεγάλες εκδηλώσεις ένα χρόνο νωρίτερα και πριν από έξι μήνες ή για τους επόμενους έξι μήνες έχει κανείς κλείσει. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα να παρακαλέσω μόλις καταλήγεται στο πρόγραμμα να μας το δίνετε. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε καλό προγραμματισμό. Και κάτι άλλο πρέπει στο Κοινοβούλιο να συστήσουμε μία ομάδα η οποία θα ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την κατάργηση της γραφειοκρατίας. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε να συμπληρώνουμε όλο και περισσότερα έντυπα και χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο χρόνο για αυτή τη δουλειά. Εμείς όμως είμαστε εδώ για πολιτική εργασία και όχι για να καλύπτουμε τις όλο και μεγαλύτερες απαιτήσει των γραφειοκρατών του ελέγχου. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά ίσως μπορούμε να σκεφτούμε να περιορίσουμε το χρόνο ενασχόλησή μας ε, με τέτοιου είδου θέματα κατά 25%. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο που θα μπορούσε να εξετάσει μια ομάδα μεταρρύθμιση. Ευχαριστούμε τον κύριο Ρούμπιχ. Ο συνάδελφο κύριος Ντε Γιούγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. <clears throat> να ευχαριστήσω και τον κύριο Πιτέλα και τον κύριο Βέλε για την παρουσία τους. Φυσικά υπήρξαν βελτιώσεις και θέλω να υπενθυμίσω το ζήτημα της μετάφρασης των πρακτικών της Ολομέλειας, το οποίο είναι θέμα πολύ Εμείς θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι θα πρέπει να βελτιωθεί, τι χρειάζεται βελτίωση. Έχοντας υπόψη τις ε, ευρωεκλογές του 2014, ε, έχοντας υπόψη μου τις κάτω χώρες, στην πατρίδα μου και άμα ρωτήσουμε τους πολίτες το, η άποψή τους δεν είναι ιδιαίτερα θετική για την λειτουργία του οργάνου μας και την αποτελεσματικότητα. Ήδη συζητήσαμε το ζήτημα ότι περίπου 300 ότι κάποια εκατομμύρια προσφέρονται για την γενική λειτουργία, αλλά υπάρχουν όμως και πολλές ε, παρατυπίες και απάτες θα έλεγα. Οι πολίτες ε, αυτά δεν ε, κατορθώνουν να τα κατανοήσουν. Νομίζω ότι αυτό είναι λυπηρό. Ο κύριο Βέλης στο παρελθόν είχε απαντήσει στο ζήτημα αυτό των παρατυπιών και είχε δηλώσει πω ε, η έλεγχη είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για, τους, ε, για την Γενική Γραμματεία. Ε, εντάξει, τέτοιου απαντήσει δεν μπορώ να πω ότι με ικανοποιούν και θα ήθελα να με ακούσω και την άποψη του κυρίου Πιτέλα. Κύριε Βέλε, θα μπορούσατε να μας κάνετε μια πρόταση για ελέγχους και εφαρμογή των ελέγχων, να μας πείτε τι θα ε, σημάνει αυτό ως ε, επιπλέον προσωπικό για την ε, Γραμματεία του Κοινοβουλίου και για να έχουμε έναν συνολικό έλεγχο για όλες τις δαπάνες οι οποίες θα πρέπει να ελέγχονται στο τέλος της χρονιάς και ένα άλλο σύστημα να ελέγχουν αυτοί οι οποίοι έχουν δαπανίσει πάνω από το 50% του προϋπολογισμού. Θα έπρεπε να ε, επιστρέφονται κάποια κονδύλια στο Κοινοβούλιο. και αυτό θα μας επιτρέψει να επαναφέρουμε τους ελέγχους εκεί όπου πραγματικά υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ε, για απάτες εάν το 5% αυτών των κονδυλίων χρησιμοποιήθηκε ή όχι. Θέτω το ερώτημα στον κύριο Βέλε και στον κύριο Πιτέλα, το έξοδο ταξιδίων. το κάτι το οποίο συγκρίνεται με την απόσταση η οποία όμως είναι κάτω από κοπήν έχουμε ήδη μια ημερήσια αποζημίωση που λαμβάνουμε εμείς οι βουλευτές για κάποιες δαπάνες λοιπόν τι ε, έχουμε για την αποζημίωση αυτή της, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με την απόσταση πάντα για τα ταξίδια υπάρχουν διάφορα προβλήματα Έφυξα μερικά Ας λάβουμε υπόψη μας ε, το ποσό το οποίο ε, μας χορηγείται αν ε, ταξιδεύουμε με τρένο ή με αεροπλάνο για μακρινές αποστάσεις. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί 100%. Γι' αυτό κρίνω ότι κάποια μορφή ελέγχων θα πρέπει να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Χρειάζεται να ληφθεί απόψη, απόφαση από το Προεδρείο για το ζήτημα των αποστολών ε, του, που αφορούν στο Κοινοβούλιο και όχι για ιδιωτική φύση ταξίδια. Και θα έχουμε ένα point system. Κάτι ακόμα. Όταν ε, μας δίνονται επιστροφές και σε αυτό πολλές φορές εμπλέκονται οι ταξιδιωτικές εταιρείες ε, το έχω δείξει το ζήτημα και μου είπαν εντάξει αυτά τα, αυτά τα points τα οποία σας δίνουν οι αεροπορικές εταιρείε μπορείτε να χρησιμοποιείτε για ιδιωτικά ταξίδια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να χρησιμοποιηθούν. Για επαγγελματικούς σκοπούς και όχι για προσωπικούς. Τώρα το Web TV, οι εργασίες στην Ολομέλη μας παρέχουν την δυνατότητα να ε, χρησιμοποιούμε αυτή την υπηρεσία. Αλλά επειδή είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά της Web TV θα πρέπει να συνεχθούμε με άλλα τηλεοπτικά μέσα για να χρησιμοποιούν αυτό το υλικό. Ευχαριστώ. <clears throat> herzlichen Dank. Äh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Βέλε και εγώ θέλω να σας ε, συγχαρώ. Εδώ είμαι, <laughs> αν δεν με βλέπετε. Καταρχήν για τον τρόπο με τον οποίο δίνετε τις απαντήσεις. Ε, πραγματικά είσαστε παράδειγμα προς μίμηση και καλό θα ήταν ορισμένοι επίτροποι να δουν τον τρόπο που απαντάτε. Πάω στο θέμα ε, του κόστους μετάφρασης και διερμηνίας. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πώς προέκυψε αυτή η ιδέα. Δηλαδή, ποιος είχε αυτή την ιδέα, πώς προέκυψε αυτή. Αυτό με ενδιαφέρει. Και επίσης ε, με ενδιαφέρει και το κατά πόσον υπάρχει μια στάνταρτ διαδικασία, δηλαδή του πώς εσείς ακούτε μια ιδέα και την υιοθετείτε. Παραδείγματο χάρη ε, υπάρχει ένα σύστημα μπόνους επιμυστίων που δίδονται στους υπαλλήλου για να έχουν ε, έτσι καλές ιδέες, για να μπορείτε κι εσείς να βρείτε κάποια κενά χρηματοδοτικής ή οικονομικής φύσης και να τα καλύπτετε. Δεύτερη ερώτηση. Όσον αφορά τους ελέγχους για τους ευρωβουλευτές, πραγματικά το βρίσκω υπερβολικό. Ο κάθε ευρωβουλευτής ε, έχει αυτό το badge, ε, αυτή την κάρτα και πρέπει να την έχει συνεχώ επάνω του. Εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Τώρα, να πρέπει να αγοράσουμε εξοπλισμό, μηχανές, μηχανήματα ε, για να ε, διαπιστώνεται κατά πόσο ο ευρωβουλευτή είναι αυτός ή όχι, αυτό εγώ το βρίσκω λανθασμένο και από πλευρά κόστους και από πλευρά προστασίας των δεδομένων. Θέλω να σας υπενθυμίσω, παραδείγματο χάρη, ε, σε εμά, και σε άλλα κοινοβούλια ο έλεγχος γίνεται στην ήριδα του ματιού. Υπερβολικό, τραγικό αυτό. Απλά και μόνο για να μπει κανείς σε ένα κοινοβούλιο, είτε είναι ευρωπαϊκό είτε εθνικό. Ας προσέξουμε λοιπόν ε, κάθε βουλευτής να έχει πάντα επάνω του την μαγνητική του κάρτα και ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος τώρα να ασχολούμεθα με το να αγοράζουμε νέο εξοπλισμό και νέα μηχανήματα για αυτό το σκοπό, για την εξακρίβωση των στοιχείων. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Βαντάλεν έχει το λόγο. Eh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Βέλ ε, για τις απαντήσεις του. Νομίζω πως ε, ακολούθησε τον, τη σωστή οδό και τον ευχαριστώ. Τώρα, θα ήθελα να κάνω κάποιες προτάσεις ε, βελτιωτικής φύσης. Οι προτάσεις ε, δεν αφορούν μόνο στον κύριο Βέλε, αλλά και στην εισηγήτρια, την οποία και παρακαλώ να σχολιάσει. Πρώτον, ο κύριος Ντεγιόγκ ε, έθιξε ήδη το θέμα των αποζημιώσεων που λαμβάνει κάθε βουλευτής για τις οποίες ε, δεν απαιτείται κανένα αιτιολογικό. Πρόκειται για 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο Γενικός Γραμματέας ε, Βέλε διερωτάται αν ε, χρειάζεται να εφαρμόσουμε κάποιο σύστημα ελέγχων και εγώ ερωτώ, δεν θα μπορούσε να γίνει κάποια περικοπή σε αυτό, στις, στις μηνιαίες της τάξης του 5% και με αυτή την εξοικονόμηση να χρηματοδοτηθούν οι θέσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να συσταθεί ένα σύστημα ελέγχου. Δεύτερον, αυτά τα ταξίδια μεταξύ Βρυξελών και Στρασβούργο εμείς ε, έχουμε τις καντίνες μας, ε, αυτά τα κουτιά, τα οποία πήγαινε έρχονται πάνω κάτω, Στρασβούργο, Βρυξέλλες και κάθε βουλευτής ε, έχει στην διάθεσή του πολλά από αυτά τα κυβότια πάνω στα οποία μπαίνει μια ετικέτα. Εγώ προτείνω να καταργηθεί το σύστημα και μόνο όσοι ζητούν να έχουν ε, μια, ένα μπαούλο ένα κυβότιο το οποίο θα διαθέτουν στο Στρασβούργο να το δηλώνουν. Έτσι η διοίκηση θα γνωρίζει πώς ε, μπαούλα θα πρέπει να μεταφέρει από τις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο και έτσι ε, μπορεί να οργανωθεί καλύτερα σε επίπεδο επιμελητίας. Θα υπάρχουν λοιπόν αυτές οι καντίν μόνο μετά από συγκεκριμένο αίτημα του κάθε βουλευτή. Θα ήθελα πάνε σε τον Βέλη και την εισηγητή. Ευχαριστώ. Κύριε Σόνικ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να συμφωνήσω με τον πρώτο αγορητή, ο οποίος δήλωσε ότι οι πάνε οι εξοικονομήσεις δεν θα πρέπει να επηρεάσουν με κανέναν τρόπο τις δραστηριότητες των ευρωβουλευτών. διότι ναι, αυτό στην ουσία συνέβη, το γνωρίζαμε, με κάποιες ιδέες αναφορικά με περικοπές που έγιναν ε, στο κόστος ε, ταξιδίων. Και κάτι ακόμα, το θέμα της ε, διερμηνίας και των διερμηνέων σε περιπτώσεις αποστολών και δι σε άλλες υπήρους δεν μπορούμε να έχουμε διερμηνείς ε, που θα βρίσκονται επί τόπου, διότι στη Λατινική Αμερική παραδείγματος χάρη υπάρχουν οι ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες ε, ε, και πρεσβείες που έχουν διάθεσή τους διερμηνείς. Καταλαβαίνω ότι χρειάζεται κάποιος διαπιστευμένος διερμηνές, αλλά αναφίβολα μπορούμε να βρούμε κάποιους διερμηνείς επιτόπου και αυτό μας επιτρέψει να πληρώσουμε τα πάντα και θα έχουμε τα έξοδα ταξιδίου τους διευνείς θα τους αναστήσουμε μέσω των πρεσβειών μας. το κόστος ε, που αφορά στο Στρασβούργο. Θα ήθελα να γνωρίζω ποιο είναι το κόστος του Λουξεμβούργου, διότι ας μην ξεχνάμε ότι το Κοινοβούλιο έχει μια τρίτη έδρα στο Λουξεμβούργο. Και αν είμαι καλά πληροφορημένο, ε, προβλέπονται νέε επενδύσει ε, και νέε εγκαταστάσει στο Λουξεμβούργο. Έπειτα υπάρχει και κάτι ακόμα που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλέ δεν είναι θεμελιώδη ζήτημα, αλλά θα μπορούσε να προβλεφθεί η ύπαρξη μιας, ε, ενός μικρού βιβλιοπολίου, θα έλεγα, στο, σε μια γωνιά του Κοινοβουλίου, διότι όλοι αγοράζουμε βιβλία, να υπάρχει λοιπόν ε, ένα, ένα, ένα γραφείο που να αναλάβει αυτό το έργο. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση εκ μέρους του κυρίου Κερμπραντ που δεν μπορεί να είναι εδώ. Νομίζω ότι μια ερώτηση ήδη ετέθη. Μιλάω για το ψήφισμα το περσινό της Ολομέλειας που ψηφίστηκε στην Ολομέλεια το ανώτερο σώμα του Κοινοβουλίου με το συντομότερο δυνατό να γίνονται ηλεκτρονικοί έλεγχοι ε, των βουλευτών όταν μπαίνουν στο κτίριο. Μιλήσατε βέβαια για ένα νέο σύστημα, οπότε εν μέρη απαντήσατε. Όταν εμφανίστε, δηλαδή η εικόνα ενός ευρωβουλευτή, το ενός ευρωβουλευτή κάπου. πρέπει να καταργηθεί το Europal TV. Το είχαμε πει αυτό και γιατί δεν το κάναμε. Είναι ένας τρόπος εξοικονόμησης χρημάτων και αυτός και είναι και απόφαση της Ολομέλειας. Πραγματικά μου εντυπωσίασε η περιγραφή των οικονομιών από το Γενικό Γραμματέα. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει αυτή η τάση και υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσα να πω. Είμαι εντυπωσιασμένο, όχι πάντοτε θετικά, από τον αριθμό των ανθρώπων που δουλεύουν ε, στις ε, πρωτεύουσε των κρατών μελών ε, για το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Πολλοί κόσμος κάνουν καλή δουλειά σε γενικές γραμμές, οργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις και βραδιές στις οποίες μας καλούν και όλες και γενικά η προσέλευση είναι αθρώα Επίσης προσλαμβάνουν συμβούλους ε, για να ε, είναι τέλο πάντων υπεύθυνοι της βραδιάς και της εκδήλωσης. Θα μπορούσε κάποιος από εμά ε, να είναι υπεύθυνο των διαφόρων συζητήσεων και συντονιστής των συζητήσεων που γίνονται σε εκδηλώσεις αυτές ή τέλο πάντων από το προσωπικό των αντιπροσωπιών στην κάθε πρωτεύουσα. Δεν χρειάζεται να προσλαμβάνουν καινούριου. Και αυτό θα ήταν μια οικονομία. στο Ζάγκρεπ. Ανοίξαμε ένα καινούριο γραφείο από ό,τι άκουσα. τι γίνεται, πρέπει να αγοράσουμε ένα κτίριο εκεί, να μισθώσουμε ένα κτίριο, πρέπει να αγοράσουμε, πάση περιπτώσει, τα γραφεία μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποια είναι συνήθως η πολιτική. Για την Ολομέλεια, ελπίζω να μην είναι συμβολικό, αλλά μου φαίνεται πολύ εντύπωση ότι λίγο μετά ε, την οικοδόμηση του κτιρίου και, το, και η οροφή του κτιρίου στις, ε, στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες καταραίει. Τι εγγύηση έχουμε και ποιος θα την πληρώσει. Ποιο ήταν ο υπεύθυνο αυτού του έργου, φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνε. Είναι πραγματικά φοβερό ότι σε 10-20 χρόνια από την οικοδόμηση του κτηρίου πέφτει το ταβάνι. Και μάλιστα το περίεργο είναι ότι συμβαίνει και στο Στρασβούργο και στι Φρυξέλλε. Και το τελευταίο μου ερώτημα Είμαι υπέρ των εξοικονομήσεων όσο το δυνατόν περισσότερο και σε σχέση με τη διερμηνία νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλές μεγαλύτερες οικονομίες. Αλλά όταν βλέπω τις απαντήσεις που δίνονται σε ερωτήσεις των ευρωβουλευτών ε, είναι στα γαλλικά και στα αγγλικά. Και δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρο ότι ένας ε, ευρωβουλευτής ε, γνωρίζει πολύ καλά και τη γαλλική και την αγγλική. Αυτό μου φαίνεται λίγο υπερβολική υπερβολικό. Νομίζω ότι θα πρέπει να αρκεστούμε σε μία γλώσσα μόνο τα αγγλικά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μούλτε και η Αποσπάτα επόμενη. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να συμφωνήσω γενικά με τους συναδέλφους, αλλά εισαγωγικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους πήραν το λόγο. Εγώ είμαι υπεύθυνη για τα κτίρια. Και έχω κάποια πράγματα να πω, κάποιες επικρίσεις να διατυπώσω σε σχέση με το κτίριο του οίκου της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση που δεν ε, προσλάβατε νέους ε, εργαζομένους. Για τις ειδικέ εργασίες, ε, επειδή δεν έχουμε ιστορικούς, θα πρέπει να έχουμε εξωτερικούς συνεργάτες. Και χαίρομαι όλος ιδιαίτερος γιατί η Επιτροπή Προϋπολογισμών ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτό το θέμα και κυρίως το περιεχόμενο μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, όχι το ίδιο το κτίριο. Ο τομέας ε, της ε, τεχνολογίας των πληροφοριών ε, επεκτείνεται. Είναι ο τομέας μου και η σχέση κόστους και ωφέλους είναι πάρα πολύ δύσκολο να οριστεί. Ίσως αν είχαμε Wi-Fi θα κάναμε πάρα πολύ μεγάλες οικονομίες, ειδικότερα στις πράσινες εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια των ε, εβδομάδων των επιτροπών, πολλοί ε, κόσμος ε, είναι εδώ. Πολλές φορές έχω πρόβλημα με το δίκτυο του κινητού μου τηλεφώνου. Δεν μπορώ να πιάσω γραμμή. Οι υπεύθυνοι πληροφορικής ζητούν όσο το δυνατόν περισσότερα για να έχουν στη διάθεσή τους τις καλύτερες τεχνολογίες, γιατί όλοι θέλουν το καλύτερο όσον αφορά τώρα τη διερμηνία. Εγώ μιλάω τσεχικά, όπως ακούτε. Ε, είναι μια από τις μικρές γλώσσες. Εγώ πιστεύω ότι τα μέτρα οικονομίας είναι καλά. Ελπίζω να συνεχίσουμε να διαθέτουμε τη διερμηνία στις μικρές γλώσσες. Το σύστημα δεν μου δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Μερικές φορές υπάρχει ένα επιπλέον διοικητικό άχθος ε, για τους βουλευτές που έχουν μία μικρή γλώσσα ως μητρική γλώσσα, αλλά αυτό είναι κάτι που μπορεί να βελτιωθεί. Μου κάνει επίσης εντύπωση όσον αφορά τον έλεγχο στα κτίρια, Εμένα δεν μου, δεν με ενόχλησε ποτέ να περνάω από μια ειδική πόρτα στο ε, κοινοβούλιο Το να εμφανίζεται μία φωτογραφία νομίζω ότι δεν υπάρχει, δεν δημιουργεί πρόβλημα σε κανέναν. Γιατί αν γίνει διακοπή ρεύματο, α πούμε, μπορεί ο κόσμο να παραμείνει ε, καθυλωμένο μέσα στου ανελκυστήρε. Είναι περίεργο να μην ξέρουμε ανά πάσα στιγμή ποιο είναι μέσα στο κοινοβούλιο. Μπορεί να γίνει μια πυρκαγιά, ας πούμε. Πιστεύω ότι οι ευρωβουλευτές πρέπει να περνούν από τις ειδικέ πόρτες τις ελεγχόμενες και ελπίζω οι κάμερε εισόδου να μην είναι πάρα πολύ δαπανηρέ. Νομίζω ότι οποιοδήποτε εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανεξαρτήτω καθεστώτο, πρέπει να κάνει το ίδιο πράγμα. Έχουμε ένα νέο σύστημα ε, λογιστικό για τα ταξίδια. Από διοικητική απόψεω, εμένα αυτό με επιβαρύνει. Δεν είναι οικονομικό το ζήτημα πρόκειται για μία αύξηση του διοικητικού άχθους. Αν από μετά από δύο μήνες ε, η γραμμα, γραμματεία μπορεί να κάνει μια αξιολόγηση του κατά πόσο βελτιώθηκε η υπηρεσία, ίσως, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό τώρα. Äh, Αγαπητοί συνάδελφοι, όλες αυτές οι ερωτήσεις που ετέθησαν είναι πολύ σημαντικές. Επειδή όμως υπάρχει και άλλη μια ειδική έκθεση που πρόκειται για την απαλλαγή ε, των άλλων οργάνων και την εκλογή του Αντιπροέδρου και ε, έχουμε χρόνο μόνο μέχρι τις 12.30. Σας παρακαλώ πολύ, δυνατόν είσαστε σύντομοι. Θα λάβουν το λόγο οι ομιλητές που αναφέρω, ο κύριος Ντότς πρώτα και μετά θα κλείσει η συζήτηση. Ο κύριος Ντότς, λοιπόν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας καταστήσω σαφές. Υποστηρίζω τη χρήση όλων των κονδυλίων που χρειάζονται για τη συντήρηση των κτηρίων του Κοινοβουλίου. Αλλά κάθε χρόνο, εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών, κάθε φορά που συζητούμε την ετήσια απαλλαγή, πρέπει να απολαμβάνουν συνεχώ τα ίδια πράγματα. θα μπορούσαμε να καταργήσουμε τα πάντα, οπότε δεν θα είχαμε και κανένα ε, κόστος. Ή μπορώ να πω, ας πούμε, οι βουλευτές δεν θα έπρεπε να πληρώνονται, αλλά θα έπρεπε να πληρώνουν ε, μπαίνοντα ε, στο κτίριο στο Στρασβούργο ή στη Βρυξή, Μπορούσαμε να πληρώνουμε, ας πούμε, ε, μια συνδρομή ε, συμμετοχής. ώστε να μην υπάρχουν ταμπλόιτ στο Λουξεμβούργο ή σε άλλες χώρες ε, που ε, να ε, μας τραβοκοιτάνε και έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συμμετέχει στην χρήση των εσόδων από τους φορολογουμένους. Νομίζω λοιπόν ότι υπερβάλλουμε μερικές φορές τις οικονομίες που προτείνουμε ή κάποιοι συνάδελφοι υπερβάλλουν σε αυτό. σου πω, πλάκα κάνω. Δεν θέλω να πείτε ότι θέλει, να, θέλει ο κύριος Δόιτς να καταργήσουμε τις αμοιβέ των ευρωβουλευτών. Αστείο έκανα. Τώρα πιο σοβαρά. συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει μια θεσμική θεώρηση να δούμε ποιοι τομείς είναι πιο αποτελεσματικοί στη χρήση των κονδυλίων και σε ποιους τομείς μπορούμε να κάνουμε τις μεγαλύτερες οικονομίες. Το ερώτημα λοιπόν είναι τις οικονομίες που θέλουμε να κάνουμε στη διερμηνία. Τι νοσηδέα ήταν αυτή και πώς μπορεί να συμπεριληφθεί στην διαδικασία λήψη αποφάσεων. Αυτό είναι μια ιδέα. Να ξέρουμε δηλαδή ε, σε ποιου τομεί μπορούμε να κάνουμε οικονομίες. Εγώ θα συμμετείχα ευχαρίστω σε μια τέτοιου είδους ε, διαδικασία. Κάτι άλλο που δεν το λέω ηρωνικά, ούτε κάνω πλάκα. Οι τελευταίοι μήνες έδειξαν ότι μπορούμε μια χαρά να τα πάμε χωρίς τις μήνυ ολομέλειες στις Βρυξέλλες. Δεν είναι υπερφορτωμένο το πρόγραμμα στο Στρασβούργο, αν δεν κάνουμε μήνυ ολομέλειες στις Βρυξέλλες. Την περασμένη εβδομάδα δεν είχαμε υπερβεί τις ψηφοφορίες στο Στρασβούργο, δεν, δεν, δεν ε, ε, οι ψηφοφορίες πάνω από 30 λεπτά. Και το λέω αυτό για να σας πω ότι ίσως να μην χρειαζόμαστε τις μήνυ ολομέλειες Φρυξέλλες Δεν λέω να γίνει καφετέρια ή βιβλιοθήκη το, το, η αίθουσα της Ολομέλειας εδώ στις Φρυξέλλες Αλλά ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο χρειαζόμαστε αυτές τις μήνυ Ολομέλειες. Γιατί είδατε, με, με ανωτέρα βία φάνηκε και σε μένα και σε άλλους συναδέλφους ευρωβουλευτές ότι δεν είναι απαραίτητες αυτές οι μήνυ ολομέλειες στις Βρυξέλλες. Κάτι πρέπει να κάνουμε να έχουμε μία ε, αίσθηση της οικονομίας. Ο κύριος Ντέιβις, ευχαριστώ πολύ. Δύο θέματα κύριε Γενική Γραμματέα σε σχέση με την προαγωγή τα εθνικά γραφεία κοινοβουλίων οργανώνουν επισκέψει δημοσιογράφων εδώ στο κοινοβούλιο και εγώ έχω ενισχύσει, έχω ε, ενθαρρύνει πολλές, δημοσι, δημοσιογράφους να έρθουν εδώ και έχουμε καταλήξει έτσι σε άρθρα σε σχέση με το τι κάνει το κοινοβούλιο, ε, ευρωβουλευτές από τη δική μου περιφέρεια κλπ. Και καταλαβαίνω ότι θα πληρώσει όλα τα έξοδα των ε, δημοσιογράφων εκτός μόνο όμως αυτές τις περιπτώσεις. Τι γίνεται όμως στο Στρασβούργο. Και δεν καταλαβαίνω αν δεν καταλαβαίνει κανείς πώς δουλεύει το ε, ε, κοινοβούλιο, ε, το να ερχόμαστε σε αυτή την επιτροπή έχει, νόημα μόνο αν μπορούμε να καταλαβαίνουμε πώς δουλεύει το κοινοβούλιο. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί οι δημοσιογράφοι πληρώνονται μόνο όταν έρχονται στο Στρασβούργο ε, για να καταλάβουν πώς είναι οι καθημερινές ε, ε, εργασίες των ευρωβουλευτών. Υπάρχουν, υπάρχει επίση και προσωπικό δημοσίων σχέσεων, σχέσεων με τα μέσα ενημέρωση. Έχουμε επίση ειδικά τηλεοπτικά στούντιο, στα οποία έχουμε επενδύσει. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ε, οι εταιρείε μετάδοση πρέπει κάτι να πληρώνουν, να παίρνουν δηλαδή μια μετάφραση από τα δικά μα τα στούντιο για τι χώρε του. τις καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τα πληρώσουν, ε, αλλά μερικέ φορές ε, μας λένε όχι ευχαριστούμε δεν θα πάρουμε. Και τι να σας πω, δεν βλέπω κατά πόσο αυτό αποτελεί εξοικονόμηση. Ίσως είμαστε σε καλύτερη θέση να χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά τα τηλεοπτικά μας στούντιο, υποστηρίζοντας τις ε, μεταδόσεις όταν ζητούμε από τον κόσμο να πληρώνει για τις μεταδόσεις αυτέ. Ευχαριστώ. Uh, Η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επικροτώ όλες τις βελτιώσεις και τις εξοικονομήσεις που έγιναν ε, από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου, καθώς επίσης ε, ε, ακούω και τους συναδέλφους που κάνουν νέες συστάσεις για νέες εξοικονομήσεις. Θα ήθελα όλα αυτά να έχουν γίνει πρώτη αλλά ακόμα ε, είμαστε έγκαιρα. Πολλά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε αναφορικά με τις προτάσεις περί εξοικονομήσεων. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ στο θέμα τη διαφάνειας. Εμείς, ευρωβουλευτέ, αντιμετωπιζόμεθα από τα μέσα ενημέρωση στα εθνικά σχετικά με τις εργασίες μα εδώ και ιδιαίτερα με το τι εισπράττουμε και θεωρώ ότι θα ήταν πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο να δαπανίσει γέρος κάποια χρήματα ε, με προβάλλοντας το τι χρήματα λαμβάνουμε, τι ε, ε, χρήματα δαπανούμε εμείς ως βουλευτές, διότι πολλές αναλήθειες ακούγονται και κυκλοφορούν. Οι βουλευτές από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι μόνοι που πρέπει να δημοσιεύουν τις δαπάνες, τους βοηθούς που έχουμε, τις ε, διάφορα, τα ε, διάφορες, αποζημιώσεις που λαμβάνουμε κλπ. Γιατί αυτό να μην αποτελέσει κανόνα για όλους τους ευρωβουλευτές. Αυτό θα καταστήσει αναφίβολα πιο διάφανο το Κοινοβούλιο. Πρέπει να ελευθερθούν λοιπόν μια σειρά πρωτοβουλειών που θα αφορούν στην διαφάνεια και θα οδηγήσουν στην εξοικονόμηση χρημάτων και παράλληλα θα κάνει μια προπαγάνδα υπέρ του Κοινοβουλίου. Τώρα για το ε, ζήτημα της, ε, του κώδικα συμπεριφορά των βουλευτών. Αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σε πολλά κράτη Βλέπω πως έχει ξεκινήσει μια διαδικασία επιλογής και συγχαίρω τον Κλάους Βέλε για τις εξοικονομήσεις που πέτυχε το τομέα των μεταφράσεων και των διερμηνίας στην ε, έκθεση που μας ε, έδωσε πέρυσι η ε, είδαμε διάφορες προτάσεις που αφορούσαν την περαιτέρω εξοικονόμηση πόρων. Χαίρομαι που οι προτάσεις αυτές έχουν συμπεριληφθεί ή τουλάχιστον υπήρξε μια τηλεπάθεια και είχαμε και η ΜΕΝ και η ΔΕ τις ίδιες ε, ιδέες για την επίτευξη εξοικονομησεών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Οίκο Ιστορίας, εγώ είμαι κάπως προβληματισμένος. Έχουμε ήδη το παρλαμεντάριο μου ε, γιατί θα μπορούσαν να μας ρωτήσουν γιατί θέλετε να έχετε κι άλλο ένα κέντρο που θα απευθύνεται στους επισκέπτες. Τώρα, εάν κάτι πάει στραβά και το κόστος αυξηθεί, αυτό θα συμβεί του χρόνου που είναι έτος ε, ευρωεκλογών και βλέπουμε ότι ξαφνικά πως τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν στην Ευρώπη θα έχουν και ένα περαιτέρω πρόβλημα το κόστος αυτού του οίκου. Εάν τα πράγματα λοιπόν δεν πάνε όπως ε, δεν πάνε κατευχήν, τότε αυτό το σχέδιο θα μας δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Και θεωρώ, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχουμε ανάγκη από ένα κτίριο για το, που θα χρησιμοποιηθεί ο ε, της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Έχουμε το Παρλαμεντάριο τουλάχιστον τα εγγένεια θα προβλέπονται για το έτος 2014. Γι' αυτό επαναλαμβάνω για τρίτη φορά. Εάν κάτι πάει στραβά θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Και... Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταία ερώτηση. Συνάδελφος Σαβαμέ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο γιατί τα περισσότερα καλύφθηκαν από του συναδέλφου. Νομίζω όμω ότι παρόλα αυτά εξακολουθώ να θέλω από ορισμένα πράγματα για την ε, παρέμβαση του κυρίου Ντεγιόνγκ. Όταν μιλάμε πάντοτε για χρήματα που πηγαίνουν ε, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ευρωβουλευτών είναι κάτι για το οποίο δεν θέλει να μιλάει κανείς ε, πολύ ανοιχτά. Όταν ο κύριος De λέει ότι θα μπορούσε να είναι διαφορετικό το σύστημα για κάποιους ευρωβουλευτές ε, που ε, ε, χρησιμοποιούν λιγότερες ημερήσεις αποζημιώσεις και περισσότεροι έλεγχοι σε αυτούς που χρησιμοποιούν περισσότερες. Τι να σας πω, αν ακολουθήσουμε αυτήν την οδό, θα είναι πολύ μεγαλύτερο το χάος που θα δημιουργηθεί. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι διαφάνεια Δηλαδή πραγματικά θα γίνει, θα δημιουργηθεί πολύ μεγάλο χάος. Δεν λέω εγώ ότι είναι δυνατόν να κάνω υπολογισμού ε, ε, τέτοιους για το τι είναι και τι δεν είναι δυνατόν, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι διαφάνεια. Δεν θα μπορούσαμε, ας πούμε, να ελέγξουμε πάντα. Πολλοί ε, πολίτες, οι περισσότεροι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα χαίρονταν αν με τον πρωινό τους καφέ διαπίστωναν ότι γύρονταν περισσότεροι έλεγχοι στους ευρωβουλευτές. Αλλά η ουσία ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, μεγαλύτερο χάος. Αν θέλουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα και αν θέλουμε να έχουμε διαφανείς κανόνες, Α υπάρχει μια αποζημίωση, ένα χι ποσό ε, σε ευρώ. Ο Στάινμπρουκ είπε ότι όταν είπε για το μισθό του, ναι, έκανε αυτό το τεράστιο λάθος για, τα, για τους μισθούς που πρέπει να πληρώνονται στους ε, πολιτικούς. Και ο κύριος Ντόιτς το είπε. Αν δεν μπορούμε εμείς να ελέγξουμε το άλογό μας, ε, τότε τι να πω, ας ε, κλείσουμε για το Κοινοβούλιο. Vielen Dank. Äh, zum Abschluss sehr Πολύ ωραία. Τελευταία ερώτηση παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω την συγγήτριά μας Εύα που έχει πάρει το δρόμο να καταστεί μια από τις καλύτερες ευρωβουλευτές μας. Ευχαριστώ κύριε Γενική Γραμματεύ Συχνά στον Νίκο μας ε, κυκλοφορούν διάφορες φήμες ε, ειδικά με την υποβάθμιση της ασφάλειας κλπ. Πάντως όλες τις οι ε, είναι σημαντικές και σας ευχαριστώ τώρα για την πολυγλωσία. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι καταδικάζουν την πολυγλωσία. μα είπατε τα μέτρα που λάβατε και διερωτώ αν δεν έχει φτάσει η στιγμή προκειμένου να κάνουμε μια γενικότερη αξιολόγηση. Διότι επί των μεταφρασμένων εγγράφων των τροπολογιών που καταθέτουμε εμεί οι βουλευτές μας ε, επιβάλλουν να καταφέρουν τροπολογίε στα αγγλικά και όταν μας μιλάτε δεν νομίζω ότι επιδεινώνεται ο, η πολυγλωσία ενώ στην καθημερινότητα ω βουλευτές αισθανόμαστε την υποβάθμιση αυτού της πολυγλωσίας. Δεν δηλαδή μπορούσε να γίνει μια αξιολόγηση ανάμεσα στις μεταφράσεις και τις διερμηνίες, δεν είναι το ίδιο επάγγελμα πάνω στο ζήτημα αυτό της πολυγλωσίας και κάτι ακόμα για τα κτίρια τα κτίρια μας είναι καινούριο πλήστον, αλλά ξέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του βίου της γίνονται πολλές εργασίες κλπ. Έχουν προβλεφθεί αρκετά κονδύλια για τα μεγάλα έργα που θα πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια της χρησιμοποίησης αυτών των ε, ε, Πολύ ωραία λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, Αυτά τα θέματα αφορούν όλους εμάς τους ε, ευρωβουλευτές. Ε, τέθησαν ερωτήματα που δεν μπορούν ε, να απαντηθούν από τον Γενικό Γραμματέα. Είναι καθαρά δικά μας θέματα. Ίσως μπορεί να τα απαντήσει ο Αντιπρόεδρος. Εμείς ως ευρωβουλευτές καλούμεθα να τοποθετηθούμε ας πούμε επί του κώδικα συμπεριφοράς. Αυτό δεν είναι θέμα της διοίκησης και γι' αυτό λοιπόν, εξ ονόματος της Επιτροπής, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τη διοίκηση, γιατί η διοίκηση είναι εκείνη που ε, εφαρμόζει και εκτελεί αυτά που αποφασίζουν οι ευρωβουλευτές. Κύριε Αντιπρόεδρε, απευθύνομαι σε εσά. Όσον αφορά τα πολιτικής φύσεως θέματα, ας πούμε τα καταποκοπή ποσά, μπορείτε να μας ενημερώσετε, υπάρχει κάτι στο Προεδρείο, κάποια εξέλιξη που να πρέπει να γνωρίζουμε ή μήπως θέλετε να λάβει το, το λόγο καταρχήν ο Γενικός Γενικός Γραμματέας και μετά εσείς. Τι θέλετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με τα χαράς δέχομαι το έτοιμά σας και θα ήθελα να υπερθυμίσω ότι για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις δαπάνες, την αποτελεσματικότητα των δαπανών και την πραγματοποίηση εξοικονομήσεων που δεν θα επηρεάζουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των εργασιών μας Δηλαδή, συστάθηκε μια ομάδα εργασίας που αποτελείται από εκπροσώπους του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμού και του Γενικού Γραμματέα που τα τελευταίους μήνες εργάστηκαν εντατικά και για μέτρα τα οποία ζητήσει η Ολομέλεια και τα και η σχετική ομάδα εργασία ε, αποδίνει το αποτέλεσμα αυτού των ε, εργασιών, αυτού του προβληματισμού. Ο Γενικό Γραμματέα υπενθύμησε πω ε, έχουμε και συγκριτικέ μελέτε σχετικά με τι εργασίε, τι δαπάνε αλλά και τα μέτρα των αποσμίωσεων για του βουλευτέ σε ό,τι αφορά τους βοηθούς του, το κόστος ε, ταξιδιών κλπ. Γίνονται λοιπόν συγκριτικές μελέτες για τα όσα συμβαίνουν στον Νίκο μας και στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών και στο ε, ε, Γερμανικό Κοινοβούλιο, το Ιταλικό Κοινοβούλιο και ούτω καθεξής. Αυτές οι μελέτες λοιπόν, οι δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, αλλά καταρχά δείχνουν ότι το Κοινοβούλιο μας είναι από μακριά το λιγότερο δαπανηρό φυσικά έχει κάποιες δαπάνες ε, που δεν ε, αναλαμβάνουν τα άλλα κοινοβούλια. Η πολυγλωσία είναι μια δαπάνη που αφορά εμάς, αλλά δεν υπάρχει ανάγκη να, στα άλλα κοινοβούλια που πρέπει να διασφαλίσουν την διερμηνία και τη μετάφραση για τόσες γλώσσες όπως συμβαίνει σε εμάς ε, μετά από τις αλλαγές που κάναμε και υλοποίησαμε κάποιες εξοικονομήσεις ε, τώρα. Οι συγητές ε, που έθιξαν κάποια προβλήματα ε, για τις καινοτομίε που πρότεινε και υλοποίησε η ομάδα εργασίας, εντάξει θα τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη, υπόψη μας, θα γίνουν αντικείμενο εργασιών αυτής της ομάδας εργασίας και επιφυλασσόμεθα να τις εφαρμόσουμε εάν οι προτάσεις αυτές σε σχέση με τα έξοδα ταξιδίου, αποζημιώσεις κλπ. θα θεωρηθούν ε, ως αποδεκτές από την ομάδα εργασίας φυσικά μετά από συνεννόηση με την ε, διοίκηση του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αντιπρόεδρε για όλα αυτά που είπατε και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Γενικό Γραμματέα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ε, προσπάθησα να σημειώσω όλες τις ερωτήσεις και ελπίζω να είμαι σε θέση να απαντήσω ε, ικανοποιητικά σε αυτές. Καταρχήν, προς τον κύριο Βον, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά κατά την προετοιμασία αυτού του προϋπολογισμού ε, και οι εξοικονομήσεις ε, που παρουσιάζουμε τώρα στο πλαίσιο του ελέγχου των προϋπολογισμών είναι το αποτέλεσμα της δικής μας συνεργασίας. Όσον αφορά τώρα πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι έχουμε τρεις θεσμούς που και τρεις είναι κοινοβουλευτικής φύσεως. Δηλαδή, έχουμε πολύ πιο στενή συνεργασία εμείς αυτοί οι τρεις θεσμοί από ότι με άλλα όργανα. Και μάλιστα αυτοί οι τρεις θεσμοί είναι και γείτονέ μας στις Βρυξέλλες. Άρα δηλαδή αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε εγώ και ο συνάδελφός μου από την Επιτροπή των Περιφερειών, η την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, για να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα. Υπάρχουν κάποια θέματα που είναι δικές μας επιθυμίες, αλλά υπάρχουν και άλλα επιθυμίες ε, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Παραδείγματο χάρη, εμείς διαθέτουμε τις αίθουσε ε, που είναι πολύ σημαντικές για τους υπαλλήλους τους. Αλλά μπορώ να φανταστώ ότι από τη δική τους ε, την πλευρά επιθυμούν να υπάρχουν καλύτερες υπηρεσίες στον τομέα της διερμηνίας και της μετάφρασης όπου το Κοινοβούλιο πράγματι έχει την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα δυνατότητα να προσφέρει όλα αυτά. Όσον αφορά το video conferencing, ε, δίκιο έχετε, ε, ίσως μπορούμε λιγάκι να το οργανώσουμε αυτό πολλές φορές. Ε, δεν είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτό το θέα. Τώρα, όσον αφορά τη μεταφορά κονδυλίων. Εκεί θέλω να πω ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε τώρα, στο τέλος του 2012 εκτελέσαμε το 99,2% του προϋπολογισμού. Και αυτό είναι ρεκόρ. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι κατά τα επόμενα έτη θα έχουμε πλήρη χρήση των κοντιλίων του προϋπολογισμού γιατί θα προσθεθούν κονδύλια ε, για το κτίριο Κόνρατ Αντενάουρ. Βέβαια δεν θέλουμε να ε, αναλάβουμε χρέη, δεν θέλουμε να καταφύγουμε στα δάνεια. Ε, και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Η κυρία Γιάλα ε, ρώτησε σχετικά με την οροφή στις Βρυξέλλες. Προς ενημέρωσή σας θέλω να πω ότι ούτε το κτίριο στο Στρασβούργο ούτε το κτίριο στις Βρυξέλλες κατασκευάστηκαν από εμάς. Ε, πρόκειται για κατασκευαστές, στην περίπτωση αυτή ο Δήμος του Στρασβούργου που κατασκεύασε το κτίριο με δική του του ευθύνη εμείς αναλάβαμε τα κτίρια αυτά στις Βρυξέλλες. Το κτίριο PHS ε, είναι πάνω από 20 ετών και μετά από 20 έτη ε, παραγράφονται η αστική ευθύνη. Άρα δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να εγκαλέσουμε τον ε, κατασκευαστή ούτε και κανέναν άλλον. Αναφερθήκατε σε σύγκριση κοινοβουλίων. Πράγματι, το αποτέλεσμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Εμείς εντοπίσαμε τέσσερις τομείς όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκριτικά είναι υποεξοπλισμένο. Ο ένας τομέας είναι η επιστημονική ε, παροχή ειδικών υπηρεσιών σε σύγκριση με το γερμανικό Bundestag αλλά και με τη Βουλή των Αντιπροσώπων της, ε, των ΗΠΑ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υποεξοπλισμένο. Στον δεύτερο τομέα, scrutiny αναφέρεται αυτός, ε, λέγεται στα αγγλικά, κοινοβουλευτικός δηλαδή έλεγχος. Ε, το, στις Ηνωμένε Πολιτείε η Βουλή των Προσώπων έχει δικό του accounting office ε, όπου ελέγχονται οι ε, νομοπαρασκευαστικές πράξεις, τα νομοθετήματα για ε, να υπάρχει έλεγχος και δυνατόν και βελτιώσεις. Και εκεί μιλάμε για 3.300 υπαλλήλους σε αυτήν την υπηρεσία. Δεν είναι εκτελεστική μονάδα, μονάδα δηλαδή της εκτελεστικής υπηρεσίας, αλλά υπάγεται στο κοινοβούλιο. Εντάξει, εμείς δεν χρειαζόμαστε τόσους πολλούς υπαλλήλους, αλλά το ερώτημα ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του δικού μας του κοινοβουλευτικού έργου, αυτό πρέπει να το μελετάμε και μέχρι τώρα δεν επενδύσαμε αρκετά σε αυτό. Αυτός λοιπόν είναι ένας ε, τομέας ε, όπου θεωρώ ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Στον τομέα της ασφάλειας, οι συμβάσεις ε, που προσφέρονται τώρα είναι συμβάσεις έργου αρκετά ε, ευνοϊκές είναι μια συνδυάσεως μορφής ε, συμβάσεις έργου. Δηλαδή είναι αορίστου χρόνου αλλά μπορούν να καταγγελθούν. Και αυτό ε, προσφέρει μια ευελιξία. Νομίζω ότι είναι μια καλή λύση. Όσον αφορά τι αντιπροσωπείς, η κυρία Αγιάλα ερώτησε πώς μπορούμε να προβούμε σε εξοικονομήσει. Δικαιολογημένο το ερώτημα. Κατά τη συνεδρίασή του του Ιανουαρίου, το Προεδρείο έλαβε μία απόφαση η οποία αναμφίβολα σε συνεργασία με τη διάσκεψη των Προέδρων θα συμβάλλει έτσι ώστε στα ταξίδια των αντιπροσωπιών να συμμετέχουν μόνο τα μέλη και οι αναπληρωτέ. Δηλαδή, ε, την τελευταία στιγμή, παρότι κάποιο δεν ανήκει ε, σε μία αντιπροσωπεία, εντάξει, μπορεί να έχει ειδικέ γνώσει για μία χώρα, δεν μπορεί να προσθεθεί στην αντιπροσωπεία. Θα πρέπει κανεί, αν θέλει να κάνει το ταξίδι τη αντιπροσωπεία, να ασχολείται ε, για μεγάλο χρονικό διάστημα με την αντιπροσωπεία αυτή. Και βεβαίω και στόχο είναι η μείωση των δαπανών. Ο κύριο Ρούμπιχ είπε πολύ καλά λόγια για την εξοικονόμηση κονδυλίων και για το πρόσωπό μου και τον ευχαριστώ θερμά αυτό. Όσον αφορά τη διερμηνία, νομίζω αυτό που μάθαμε με το περίφημο κρούα, δηλαδή με ε, την μετάφραση των πρακτικών σε όλες τις γλώσσες, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε με το ε, σύστημα προσφέρουμε την υπηρεσία μόνο εφόσον ζητηθεί. Ακόμα και αν ένας μεμονωμένος ευρωβουλευτής θέλει τη μετάφραση, να του την προσφέρουμε. Αν όμως κανένας ευρωβουλευτής δεν ζητάει πρακτικά, γιατί να του τα προσφέρουμε μεταφρασμένα. Αυτή είναι μια πολύ σωστή αρχή, η οποία βεβαίως και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με διακριτική μεταχείριση. Ένας και μόνο να το θέλει, βεβαίως, του το προσφέρουμε. Αλλά αλλιώς ε, δεν έχει κανένα νόημα να προσφέρουμε μια υπηρεσία που είναι αχρηστή. Και επίσης το θέμα της ε, παθητικής ε, διερμηνίας ε, στα ταξίδια των αντιπροσωπιών και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Ο κύριος Ντεγιούγκ μίλησε θετικά και κατόπιν έφυξε μια σειρά συγκεκριμένων ερωτήσεων. Όσον αφορά τα καταποκοπή ποσά, εγώ ως διοίκηση μπορώ να σας πω ότι αν αρχίσουμε σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση να ελέγχουμε τα καταποκοπή ποσά, ως διοίκηση πρέπει να σας πω ότι μιλάμε για ένα τεράστιο φόρτο εργασίας, ο οποίος ε, θα αντανακλάται με αυξημένες δαπάνες. Αν το θέλετε, αν είναι αυτή η πολιτική σας βούληση, ευχαριστώ να το κάνουμε. Αλλά μέχρι τώρα η απόφαση που ισχύει είναι ότι στα καταποκοπή ποσά δεν γίνεται περαιτέρω έλεγχος και ε, διατηρούνται αυτά. Ε, μιλήσατε επίσης και για το καταποκοπή ποσό, στα ταξίδια, στις δαπάνες ταξιδίων. Ε, όσον αφορά τους ε, πόντους ε, που μαζεύουν οι ευρωβουλευτές από τις ακτιτικές εταιρείες, τα μπόνους αυτά, εμείς δεν μπορούμε αυτά να τα ελέγξουμε και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να ελέγξουμε κατά πόσο χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς. Για το Web TV έχουμε χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης ε, λόγω της συνεργασίας ε, που θα έχουμε με άλλα κανάλια. Αυτό το θέμα συζητήθηκε ε, από τον αρμόδιο αντιπρόεδρο και η Ολομέλη αποφάσισε για το τέλος του 2013 να διατεθεί σε αυτό τον τομέα το ποσό των 8 εκατομμυρίων. Βεβαίως μπορούμε να σκεφτούμε κατά πόσον μπορούμε να χρησιμοποιούμε περισσότερο τέτοιου είδους παραγωγές και αυτές να γίνονται και περισσότερο με δικούς μας συνεργάτες. Γιατί με τον τρόπο αυτό θα εξοικονομούμε κονδύλια και οπωσδήποτε είναι και ένα κίνητρο για τους υπαλλήλου μας. Θα το κοιτάξω λιγάκι αυτό. Από την άλλη πλευρά βέβαια χρειαζόμαστε και τέτοιου είδους εργαλεία λόγω των επικείμενων ευρωπαϊκών εκλογών. Ε, επίσης ε, όσον αφορά το ερώτημα στη μετάφραση ε, ποιος είχε την ιδέα να ελέγξει το σύστημα. Για δύο ολόκληρες εβδομάδες ασχολήθηκα μόνος μου, γιατί ήθελα να ξεφύγω από αυτά τα καταποκοπή ποσά για τη μετάφραση. Έχουμε 23 σε διαφορετικές μονάδες, με διαφορετική απόδοση. Σίγουρα ε, υπάρχουν κάποιες μονάδες που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές και άλλα, άλλα πάλι τμήματα, όχι μονάδες τμήματα, λιγότερο αποτελεσματικά. Ε, Έπρεπε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς γίνεται στα διάφορα τμήματα, τα γλωσσικά σε σχέση με τη μετάφραση. Μετακάναμε την αξιολόγηση και μπορέσαμε να προβούμε σε εξοικονόμηση κοντιλίων. Στο κάτω-κάτω είναι και θέμα δικαιοσύνης. Αν είμαι μεταφραστής, γιατί ας πούμε σε ένα τμήμα να πρέπει εγώ να δουλεύω 50% περισσότερο από το συνάδελφό μου. Νομίζω ότι μπορούμε να προσαρμόσουμε λιγάκι τα ποσοστά και μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Γιατί ε, για τη διερμηνία. Είχαμε μία συζήτηση με την Επιτροπή ε, Προπολογισμών. Μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση. Η Γενική Διευθύντρια, η αρμόδια, είπε, κοιτάξτε, μπορώ να επιτύχω εξοικονόμηση αν υπάρχει και καλύτερο σύστημα, καλύτερες ρυθμίσεις. Είναι σαφές ότι αν ε, υπάρχουν συνεδριάσεις μετά τις 11 ώρα το βράδυ στο Στρασβούργο, είναι απαραίτητο να υπάρχουν περισσότεροι διερμηνείς, γιατί δεν μπορούν αυτοί να εργαστούν την επόμενη μέρα. Είπε λοιπόν η Γενική Διευθύντρια ότι ε, αν σταματάει ε, η νυχτερινή συνεδρίαση στις 11 ώρα αντί 12 και 4, θα εξοικονομήσω χρήματα. Βεβαίως είπε ότι και οι μέρες δεν χρησιμοποιούνται εξίσου η Δευτέρα και η Παρασκευή δηλαδή. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι εντάξει θα πούμε εμείς πλέον σε επιτροπέ να συνεδριάζουν είτε Δευτέρα Τρίτη είτε Τετάρτη Πέμπτη. Δεν μπορούν δηλαδή οι επιτροπές να αποφασίζουν απολύτω μόνος τους. Και το τρίτο είναι ότι ε, χρησιμοποίησαμε τους δικούς μας διερμηνείς κατά τις ε, τυρκουάζ εβδομάδες. Έτσι λοιπόν πολλέ φορέ οι τυρκουάζ εβδομάδες ε, χρησιμοποιήθηκαν ω μια κανονική εβδομάδα. Αυτές οι προτάσεις έγιναν από την υπηρεσία της διερμηνίας και μας επέτρεψαν να επιτύχουμε σημαντική εξοικονόμηση. Είπατε επίσης ε, ότι αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν ad hoc, ε, θα πρέπει το σύστημα να λειτουργεί ε, στον πίνεκες. Υπάρχει ένα νέο σύστημα πληροφορικής, το ERFIS. Αυτή τη στιγμή με τα τρέπουμε το σύστημα που έχουμε έτσι ώστε να μπορούμε πιο συστηματικά να βλέπουμε τι κοστίζει το κάθε ε, στοιχείο. Και θεωρώ ότι έτσι είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ο κύριος Βαντάλεν έθιξε το θέμα ε, Βρυξέλλης και Στρασβούργο, το θέμα των εμπορευματοκιβωτίων, των μπαούλων. Ε, πράγματι, σήμερα χρησιμοποιούμε πολύ χαρτί. Και εμείς από πλευράς διοίκησης ε, ε, δεν ξέρω αν μπορούμε να αποφασίσουμε για το μοίρασμα αυτών των μπαουλών. Αν ε, δύο ή και τρεις συνεργάτες μοιραστούν ένα μπαούλο, πράγματι αυτό κοστίζει λιγότερο. Αυτά όλα ήδη τα εξετάζουμε και νομίζω εδώ υπάρχει πραγματικά ένα μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό εξοικονόμησης. Ο κ. Ζόλε επίσης έθιξε το θέμα των διερμηνέων στα ταξίδια των αντιπροσωπιών. Εγώ έχω την εντύπωση ότι μερικές φορές ε, οι ευρωβουλευτές ε, νιώθουν ότι στα ταξίδια αυτά υπάρχουν πάρα πολλοί διερμηνείς και συνεργάτες και ότι ίσως ε, μπορεί να περιοριστεί ο αριθμός τους. Ε, βεβαίως αυτό σημαίνει ότι και οι ευρωβουλευτές ε, θα πρέπει να παρετηθούν από την παθητική ακρόαση, να έχουν την ενεργητική, δηλαδή να μιλάνε τη γλώσσα τους αλλά να ακούνε κάποια άλλη Αυτά είναι θέματα που αν θέλετε μπορούμε να τα συζητήσουμε, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό πρέπει να το επιθυμούν οι ίδιοι οι ευρωβουλευτές. Είπατε επίση, ε, ρωτήσατε, γιατί χρειαζόμαστε καινούριο κτίριο στο Λουξεμβούργο. Αυτή τη στιγμή είμαστε διάσπαρτοι στο ε, Λουξεμβούργο σε οκτώ κτίρια και αυτό σημαίνει ότι είμαστε αντιπαραγωγικοί. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε και στι Βρυξέλλε και στο Στρασβούργο και στο Λουξεμβούργο να συγκεντρωθούμε σε ένα κτίριο. Επειδή το ζήτησε η Επιτροπή των Προπολογισμών, κάναμε του υπολογισμού σε 20 χρόνια ε, σύγκριση. Αν υποθέσουμε ότι κατά επόμενα 20 έτη έχουμε δικό μας κτίριο σε σύγκριση αυτό με το να νοικιάζουμε ένα κτίριο ε, τι ποια θα, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και η σύγκριση απέδειξε σε 20 χρόνια θα εξοικονομήσουμε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ, αν έχουμε δικό μας κτηρίο βεβαίως με το σημερινό προβλεπόμενο κόστος. Είναι μεγάλο το ποσό και το ε, κράτος του Λουξεμβούργου, μην ξεχνάτε, ότι μας δίνει το οικόπεδο δωρεάν. Αν συγκρίνετε τι θα μας ε, κόστιζε ένα παρεμφερές οικόπεδο στις Βρυξέλλες, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ οικονομικό το να παραμείνουν ορισμένες υπηρεσίες στο Λουξεμβούργο. Ο κύριος Μούλντε έθιξε δύο ερωτήματα του κυρίου Γκεμπράντη, τα ξέφρασε εξ ονόματός του. Ε, είπα για τον έλεγχο, είπα επίσης για το Europa TV, Web TV. Κοιτάξτε, υπάρχουν ε, και διάφορα όργανα που πρέπει να απαλλαγούν. Ε, εμείς ε, ε, παρουσιαζόμεθα στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών, παρουσιαζόμεθα σε άλλες επιτροπές. Και τελικά υπάρχει το Προεδρείο το οποίο λαμβάνει τις διοικητικής φύσεως αποφάσεις. Εμείς εργαζόμεθα μέσα σε αυτό το τρίγωνο, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι κάθε ένας από εμά έχει τις δικές του τις αρμοδιότητες στο πλαίσιο αυτού του τριγώνου. Και θεωρώ πάρα πολύ, καλά, πάρα πολύ καλό ε, το ότι γίνεται αυτή η συζήτηση για τα εξωτερικά μας γραφεία. Στο Ζάγκρεπ ε, η Κομισιόν είναι εκείνη που έχει ε, καταρχήν τον κύριο λόγο στο εξωτερικό γραφείο και είπανε δεν θα αγοράσουν, θα νοικιάσουν. Ήταν πιο φθηνό κανικό. όμως προτιμούμε να αγοράζουμε και όχι να νοικιάζουμε γιατί αυτό σημαίνει εξοικονόμηση όσον αφορά τα στηρίγματα ε, για την ε, οροφή. Ε, σας είπα ότι υπάρχει και κάποια παραγραφή ευθυνών. Κατόπιν, το να υπάρχει μία και μόνο γλώσσα, γιατί αναφερθήκατε στο γλωσσικό, να χρησιμοποιούν όλοι μία γλώσσα. Δεν μπορώ εγώ να το κρίνω αυτό. Αυτό πρέπει να το πούν οι ίδιοι ευρωβουλευτέ. Μόνοι του να πούνε σε πόσε γλώσσε χρειάζονται τα έγγραφα για να είναι αποτελεσματικοί. Η κυρία Ζομποχάτα, προφέρω σωστά το όνομά σα. Σχεδόν σωστά. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, θερμά για τα πολυφιλικά σας λόγια. Προφανώς και δεν επιθυμούμε επουδενή τη διακριτική μεταχείριση εις βάρος των ε, μικρών γλωσσών, που σημαίνει αν προσφέρουμε ε, μετάφραση ή διερμηνία εφόσον ζητηθεί, αυτό σημαίνει ότι ένας Τσέχος ευρωβουλευτής έχει την ίδια σημασία όπως ένας Γάλλος. Αν οι Τσέχοι θέλουν Τσέχικα, προφανώς και θα του τα ε, προσφέρουμε. Αυτό ισχύει και για όλες τις άλλες μικρές γλώσσες. Εγώ τουλάχιστον έτσι σκέφτομαι. Όσον αφορά τώρα τους νέους ε, κανόνες ε, ταξιδιού, προφανώς ε, και χρειαζόμαστε μια νέα αξιολόγηση. Αν θα το έχουμε επιτύχει μέχρι το τέλος του μήνα, δεν το ξέρω. να αφήσουμε λίγο χρόνο, να δούμε πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Πρέπει μετά να γίνει αξιολόγηση και ενδεχομένω να διορθωθούν και λάθη. Ο κύριος Ντόιτς είπε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την εξοικονόμηση. Σωστό και αυτό. Γιατί διαπιστώνουμε ότι μερικές φορές έχουμε μεγάλη εξοικονόμηση η οποία δεν επηρεάζει τη δουλειά μας. Και άλλου είδους εξοικονομήσεις μικρής κλίμακας που όμως δυσκολεύουν τη ζωή των ευρωβουλευτών. Άρα δηλαδή και σε αυτό το θέμα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι είδους εξοικονομήσεις θα επιλέξουμε. Σας είπα, υπάρχουν μεγάλες κλίμακες με σχεδόν καμία επίπτωση και άλλες μικρές κλίμακες που όμως δυσχεραίνουν τη ζωή και τη δική σας και τη δική μας όλων μας δηλαδή. Όσον αφορά τη μήνυ ολομέλη των Βρυξελών, νομίζω και αυτό είναι πολιτική απόφαση. Ο κύριος Ντέιβις ρώτησε κατά πόσον υπάρχει αποζημίωση των ε, δημοσιογράφων μόνο για το Στρασβούργο. Όχι, μπορεί να υπάρξει και στις Βρυξέλλες. Αλλά υπάρχουν και διάφορα προγράμματα. Υπάρχουν προγράμματα πολιτικών ομάδων, άλλα του Κοινοβουλίου. Ε, ε, όσον αφορά τα προγράμματα των πολιτικών ομάδων, αυτά είναι δικό τους θέμα, αυτές αποφασίζουν. Ε, ως ε, προς ε, τα τηλεοπτικά κανάλια, αυτά χρησιμοποιούν τη δική μας την υποδομή δωρεάν, που νομίζω είναι πολύ καλή, και βεβαίως την διασύνδεση, τη σύνδεση, δίκιο έχετε, πρέπει μόνοι τους να την πληρώνουν. Ε, να δούμε αν αυτό είναι ε, λογικό, αλλά αν θέλετε και να δίνουμε και κάποια ε, μορφή ενίσχυση, πρέπει να το εξετάσουμε. Κύριε Αντρέσεν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια και όχι μόνο για την προσπάθεια εξοικονόμηση, αλλά και για την πραγματική εξοικονόμηση που επιτύχαμε το 2012 συνολικά 24 εκατομμύρια ευρώ που θα επαναλαμβάνονται για πολλά επόμενα έτη. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό το ότι το αναγνωρίζετε. Τα στοιχεία υπάρχουν, ο Ευρωβουλευτής ε, έχει νομίζω 8,5 φορές μεγαλύτερο, ε, μάλλον με συγχωρείτε, ο Ευρωβουλευτής ε, σχετικά με το μισθό του, αυτά είναι δημοσιευμένα τα στοιχεία. Για τον κώδικα διοντολογίας, ο κώδικας ε, διοντολογίας είναι ιδιαίτερα απαιτητικός και νομίζω ότι ήταν και σωστό να δούμε λιγάκι τι συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημείωσε μεγάλη πρόοδο και υπάρχει και ειδική γραμματεία που μπορεί να συνδράμει. Νομίζω λοιπόν ότι στον τομέα αυτό, στο θέμα της διοντολογίας, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Κύριε Έπινγκ, σας ευχαριστώ πολύ για τα συγχαρητήριά σας ε, όσον αφορά την εξοικονόμηση στον τομέα της διερμηνίας. Για το σπίτι της ευρωπαϊκής ιστορίας θέλω να σας πω ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία υπέρβαση κόστους. Έχουμε κάνει υπολογισμό κόστους ε, για την ανέγερση του κτηρίου και μετά από τις ε, προσφορές που ανοίξαμε θα τηρηθεί το κόστος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Οι προσφορές είναι μέσα στο πλαίσιο κόστους που έχουμε προβλέψει για την ανέγερση αυτού του κτηρίου. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει υπέρβαση κόστους. Και κατά τα άλλα θα τηρήσουμε το business plan το οποίο έχουμε συμφωνήσει με την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ε, δηλαδή και πάλι δεν προκύπτει υπέρβαση κόστους. Βεβαίω και μπορεί να τεθεί το ερώτημα αν το χρειαζόμαστε αυτό το σπίτι. Εγώ όμω θέλω να σας πω ότι όπως και το Παρλαμεντάριουμ και εδώ έχουμε μία προσφορά για τον πολίτη. Δηλαδή δεν είναι κονδύλια τα οποία θα εκμεταλλευτεί η διοίκηση, οι ευρωβουλευτές. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία ξεκάθαρη επένδυση για τον πολίτη και διαπιστώσαμε πέρυσι 250.000 πολίτες επισκέφτηκαν το Παρλαμεντάριο. Η απήχηση ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική. Βλέπετε λοιπόν επενδύουμε στον πολίτη και πιστεύω ότι το σπίτι της ευρωπαϊκής ιστορίας ε, θα αποδειχθεί μια εξίσου, ένα εξίσου επιτυχημένο εγχείρημα όπως και το Παρλαμεντάριο. Ο κ. Σάρανεκ επισήμανε το θέμα της ε, διαφάνειας. Ελπίζω η σημερινή μας συνάντηση και αυτή να συμβάλλει στη διαφάνεια. Γιατί απαντήσαμε σε πάρα πολλές ερωτήσεις τώρα ε, προφορικά αλλά και πριν από τη συνεδρίαση σε γραπτή μορφή. Γνωρίζετε ότι δεν συμμετέχουν σε αυτή τη διαφάνεια όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και θα ήταν ε, καλό αν και το Συμβούλιο συμμετείχε σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί σήμερα είμαστε συνομοθέτες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι συνομοθέτες, άρα δηλαδή πρέπει να ανταποκρίνονται στις ίδιες απαιτήσει ως προς τη διαφάνεια. Ο κύριος Οντί, και νομίζω έτσι σιγά σιγά τελειώνω, ε, έθεσε το θέμα της πολυγλωσσίας. Ένα πολύ σημαντικό θέμα για εμάς και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η ιδέα του on demand μετά από έτοιμα είναι πολύ καλή. Αν κάποιο ευρωβουλευτής επιθυμεί κάτι, του το προσφέρουμε, αλλά αν δεν το επιθυμεί, τότε δεν το προσφέρουμε κι εμείς Δηλαδή, προσαρμοζόμαστε στις επιθυμίες του Ευρωβουλευτή. Και αν το κάναμε αυτό και σε άλλες περιπτώσεις, αυτό θα ήταν πολύ καλό για τον Ευρωβουλευτή, αλλά και για την εξοικονόμηση κόστους. Σωστά λοιπόν επισημαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση. Τώρα, δημιουργία αποθεμάτων για μελλοντικά κτίρια, για κτίρια στο μέλλον, αυτό απαγορεύεται από τον κανονισμό του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι απάντησα, ε, εξάντλησα όλες τις ε, ερωτήσεις και ε, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Γραμματέα και κύριε Αντιπρόεδρε για την διεξοδική απάντηση των ερωτήσεων. Και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια και στο ελεγκτικό συνέδριο για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Θέλω βέβαια να επισημάνω ότι ένα θέμα που μας απασχολεί στην Επιτροπή Ελέγχου Προεπολογισμών είναι ο αποτελεσματικός έλεγχος. Δηλαδή, ε, πώς μπορούμε να επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα με τα χρήματα του φορολογούμενου ε, σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν είναι θέμα ύπαρξη ή όχι κοινοβουλίου. Το ότι υπάρχουν βέβαια κάποια, κάποια πολιτικά κόμματα ή ομάδες που το βλέπουν έτσι, αυτό δεν το ε, αρνούμε. Αλλά εμεί επιθυμούμε να έχουμε τη σωστή διοίκηση και έχει αποδειχθεί ότι οι κυβερνήσεις τεχνοκρατών δεν ε, είναι καλύτερες από την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Μπας περιπτώσει, πρέπει να υπάρξει αυτή η πολιτική αντιπαράθεση, διότι ιδιαίτερα σε περίοδους κρίσης ε, τα ε, συστήματα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας δοκιμάζονται και καλούνται να αποκτούν την εύνοια των πολιτών το θέμα της ε, καλύτερης ή της ε, χειρότερης νομοθεσίας τίθεται έτσι και αλλιώ. και χωρίς ε, την βοήθεια των Ευρωβουλευτών ενδέχεται στη νομοθετική διαδικασία να προκύπτουν λάθη τα οποία όμως κοστίζουν πάρα πολύ στον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Άρα δηλαδή λείπει το οπλοστάσιο που θα μας επιτρέπει τη σωστή αξιολόγηση, δηλαδή κατά πόσον αν υπήρχαν άλλες διαδικασίες στα κοινοβούλια θα μπορούσαν να αποφευθούν ε, λάθη για τους ε, πολίτες και ε, περιορισμός του κόστους. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για το μέλλον. Ε, επέτρεψε στον εαυτό μου να κάνω αυτή την παρατήρηση και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου για να απαντήσει εφόσον το επιθυμεί σε ερωτήματα που ετέθησαν. Παρακαλώ. Ε, ε, ευχαριστώ. Δεν υπήρξε συγκεκριμένη ερώτηση που να απευθύνθηκε στο ελεγκτικό συνέδριο. Όμως υπήρξαν κάποια ερωτήματα σε σχέση με τις προμήθειες για τα κτίρια όσον αφορά την παρακολούθηση του ελεγκτικού συστήματός μας και στο, μέρος μπορούμε, στο μέλλον μπορούμε να έχουμε πιο, ε, συγκεκριμένα, πιο συγκεκριμένες αναφορές στα θέματα που θέσατε. Ως ε, τελική παρατήρηση θα ήθελα να επιμείνω στα απορίσματα της ετήσιας έκθεσής μας σε σχέση με τις διοικητικές ε, δαπάνες ε, όλων των οργάνων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, η IES θα ήθελε να επιμείνει ότι το συμπέρασμα του ελεγκτικού συνεδρίου ότι όλες οι δαπάνες ε, ήταν νόμιμες ε, και ε, κανονικές και συνάδουν με τις απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Κύριε Τομέ Μουγκουρούσα για την δήλωσή σας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον, στην εισηγήτριά μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως συμπέρασμα θα μπορούσα να πω ότι σχεδόν μετά από το πέρας τριών ωρών συζητήσεων τα πράγματα κύλησαν ε, πολύ καλά. Ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα, σε προσώπους του Ελεκτικού Συνεδρίου, τον ε, εσωτερικό Ελεκτή και τα μέλη της Επιτροπής μας και να πω ότι αποκτήσαμε την ιδέα ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά πως η Επιτροπή μας είναι πολύ δραστήρια και αποτελεσματική στις εργασίες Σας Ευχαριστώ. Äh, ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Συγήτρια, ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο κύριο Πιτέλα, τον κύριο Γενικό Γραμματέα και σας ευχαριστώ που απαντήσετε σε όλα μας τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich äh, wollte jetzt... Αγαπητοί Τώρα θα ήθελα να περάσουμε στην εκλογή του Αντιπροέδρου. Ο συνάδελφος Ντόιτς όμω απουσιάζει, γνωρίζει κανεί αν πρόκειται να επιστρέψει στη συνεδρίασή μα ε, Αποχώρησε ε, εν αναμονή. α προχωρήσουμε στην ίδια διάταξη. Α, εδώ έρχεται ο κύριο Ντόιτ. Προβλέπεται η επιλογή ενό Αντιπροέδρου τη Επιτροπή Ελέγχου, Ελέγχου Προπολογισμών. Επειδή η κυρία Ιβάνοβα φύγε και πήγε στο ελεκτικό συνέδριο του Λουξεμβούργο. έτσι και ενώθηκε μια θέση, χείρευσε και σύμφωνα με τον κανονισμό 100 και το άρθρο 191, 12, 13, 14, 161, 169 και 187, 195, 196 εφόσον υπάρχει ένας και μόνο υποψήφιος μπορούμε να ψηφίσουμε με ανάταση της χειρός. Εάν όμως το, η Επιτροπή επιθυμεί μπορούμε να προβούμε σε μυστική ψηφοφορία. Το ΕΛΚ προτείνει τον κύριο Ντόιτς και ερωτώ θέλετε να έχουμε μυστική ψηφοφορία ή όχι. Από ό,τι φαίνεται δεν επιθυμεί κανεί τη μυστική ψηφοφορία ε, κατόπιν τούτου. Νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε ανοιχτά Επιθυμείτε ε, να ψηφίσουμε διανατά στο χειρός. Μάλιστα, ποιος είναι λοιπόν υπέρ ε, του Χαμοθόσεν. Παρακαλώ να σηκώσει το χέρι. Κατά αποχές. Από ό,τι βλέπω όχι. Έτσι ο κ. Τάμας Ντόιτς ε, εκλέγεται ομόφωνο, ο κ. Ντόιτς, και τον ερωτώ κατά πόσον αποδέχεται το αποτέλεσμα της εκλογής. Ναι, το αποδέχεται. Αποδέχεστε κύριε Ντότς το αποτέλεσμα της ε, ψηφοφορίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους ε, για την εμπιστοσύνη τους. Θα προσπαθήσω να σταθώ στο ύψος ε, του καθήκοντός μου. Η κυρία Ιβάνοβα που είναι η προκάτοχός μου έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και ελπίζω ότι και οι δικές μου δραστηριότητες θα τύχουν επίσης πολύ θετική αποδοχή. Σας συγχαίρουμε ε, στην εκλογή σας ε, στη θέση του Αντιπροέδρου. Ε, το αποτέλεσμα ήταν μετά από ομόφωνη το αποτέλεσμα της ψηφορίας ήταν ομόφωνα, ελήφθη ομόφωνα και ελπίζω, όπως είπατε, να μας βοηθήσετε στην διεκπαιρέωση των εργασιών. Πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Είναι το υπερτμόν 11, απαλλαγή άλλων θεσμών. Η... Μισό λεπτό λέει ο πρόεδρος. Οι συνεισηγητές είναι Ανδρέα Τσέσκοβα και Ρίτσαρτ Τσανέτσκι και θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο επιθυμούν να λάβουν το λόγο ή μήπως θα πρέπει να ακούσουμε πρώτα το ε, ελεγκτικό συνέδριο. Η μήπω θα πρεπει να ακουσουμε πρωτα το ελεγκτικο συνεδριο η συνάδελφο κυρια τσεσκοβα εχει το λογο προεδρε θα ηθελα να πω το εξή. Με τον συνάδελφο κάναμε τη δουλειά ε, σε συνεργασία. Εγώ είμαι υπεύθυνη για την Οικονομική Επιτροπή, για την Επιτροπή των Περιφερειών, για τον Ευρωπαίο Μεσολαβητή και για τον Ευρωπαίο Επόπτη Δεδομένων. Ο συνάδελφος είναι υπεύθυνο για το ελεκτικό Συνέδριο, για το Δικαστήριο και ο κύριος Τσανέσκι μου ζήτησε να μιλήσω εγώ διότι δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί σήμερα στην συνεδρίασή μας και έχω κάποιες ερωτήσεις που μου έδωσε ο κύριος Τσερνέσκι και θα ήθελα να τις αναγνώσω στο όνομα του συναδέλφου. Αυτά ως εισαγωγή και περιμένω με περιμένω την ε, συζήτηση που θα διεξαχθεί με τους εκπροσώπους των πολιτικών ε, λοιπόν θεσμικών οργάνων. Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο κυρία Τσέσκοβα και θα ήθελα να δώσω το λόγο στο ελεγκτικό συνέδριο, στον κύριο Τόμι Μουκουρούθα. Ε, παρακαλώ πολύ για τοποθέτησή σας. Ε, thank you, Chairman. As I told you in my Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Όπω είπα και στην προηγούμενη μου παρέμβαση, κατά το σημείο 10 τη ημερήσια διάταξη, στο κεφάλαιο 9 τη ειδική διατήθεια έκθεσή του, το Ελληνικό Συνέδριο συμπεραίνει ότι οι διοικητικέ δαπάνε όλων των οργάνων και υπηρεσιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είχαν ένα συνολικό ποσοστό σφάλματο 0,1% και για τα ελεγκτικά και επεπτικά συστήματα είναι συμβατά με τι απαιτήσει του δημοσιονομικού κανονισμού. Αυτά τα δύο συμπεράσματα ισχύουν και για τα λοιπά όργανα και υπηρεσίες. Είχα ήδη τη δυνατότητα να παρουσιάσω στην Επιτροπή τα συνολικά αποτελέσματα και τις συστάσεις του κεφαλαίου, όπως επίσης και τις ειδικές παρατηρήσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στις 10 Ιανουαρίου η Επιτροπή σας συζήτησε τη διοικητική δαπάνη της, ε, εξωτερικής υπηρεσίας, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και το απόγευμα θα συζητήσει αυτή της, της Επιτροπής. Θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα για τα πορίσματά μας σε σχέση με, τους ε, λιπούς, ε, με, τα, λοιπά, όργανα και υπηρεσίες, δηλαδή Συμβούλιο, Ελεγκτικό ε, Δικαστήριο, συγγνώμη, Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. Όπως λέγεται, αναφέρεται και στην έκθεσή μας, οι λογαριασμοί του ελεγκτικού συνεδρίου ε, ελέγχθηκαν από μια εξωτερική ε, εταιρεία ελέγχου η οποία κατήρτισε ξεχωριστή έκθεση με πορίσματα και ε, γνωμοδότηση. Το κεφάλαιο 9 συμπεριλαμβάνει σχόλια για προβλήματα του συστήματος στο Συμβούλιο και στην ε, Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή. Στους υπόλοιπους, ε, στα υπόλοιπα όργανα και υπηρεσίες δεν υπήρξαν σοβαρά προβλήματα. Όσον αφορά το Συμβούλιο, το ελεκτικό συνέδριο εντόπισε προβλήματα σε δύο διαδικασίες προμηθειών από τις πέντε που ελέγχθηκαν. Σε αυτές τις περιπτώσει, οι προδιαγραφές τη προσφορά έδωσαν τη δυνατότητα στο Συμβούλιο να εκτιμήσει μία τιμή για ένα συγκεκριμένο έργο ε, αν οι προσφορές ε, δεν πρότειναν ε, κάτι τέτοιο. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα υπήρχε μια τροποποίηση του κόστους με τρόπο που δεν συμπεριλαμβάνεται, που δεν προβλέπεται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Για την ΟΚΕ, το ελεγκτικό συνέδριο βρήκε σφάλματα σε σύναψη συμβάσεων με συμβασιούχους και προσωρινούς. Σε μία από τις τέσσερις περιπτώσεις που ελέγχθηκαν, το συγκεκριμένο πρόσωπο προσελήφθη ήρθε ως ε, προσωρινός και ε, έξι μήνες ε, μετά την πρόσληψή του έλαβε και το βασικό μισθό γιατί δεν υπήρχαν επαρκείς θέσεις για προαγωγή του. Αυτή είναι η σύνοψη των πορισμάτων μας σε σχέση με τους, τα λοιπά όργανα και υπηρεσίες. Ευχαριστώ να απαντήσω ερωτήσεις αν τυχόν έχετε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ για αυτή τη σύντομη παρουσίασή σας. Ε, τώρα να δώσω το λόγο στους ε, Γενικού Γραμματείς των υπολοιπών οργάνων. Να ξεκινήσουμε με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο, παρακαλώ. Παρακαλώ, επειδή είναι μεγάλη η αίθουσα, είναι δύσκολο να διακρίνω στο βάθο. Ευχαριστώ, πράγματι είναι μεγάλη η αίθουσα. Είμαι γραμματέα του δικαστηρίου και με, τα χαρά απαντήσαμε στα ερωτήματα τη συγγήτριας για τον απαλλαγή του 2011 και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ξέρετε ότι επιθυμεί να έχει πάντα ένα ανοιχτό και διάφανο, διάλογο με την Επιτροπή σας, Επιτροπή Ελέγχων Προπολογισμών. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην διαφάνεια σχετικά με τα δαπάνες ε, που κάνουμε στο δικαστήριο. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να παρέχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πληροφορίες ε, στο πλαίσιο των ετήσιων δραστηριοτήτων και τη σχετική έκθεσης στην έκθεση για το 2011 ελπίζω να αποτελεί για μια ακόμα φορά ένα παράδειγμα αυτής της επιθυμίας ε, επικοινωνίας ε, και πληροφόρησης ε. στην έκθεση αυτή υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά δηλαδή η χρήση των πιστώσεων και, των, και το θέμα των δαπανών χρήση των ε, πιστώσεων του 2001 ξεπερνάει το 88%, το 98% συγγνώμη, και σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό και εδώ βρισκόμαστε σε επίπεδο δαπανών 98%. Ε, ε, βάλουμε στο πλάι το turnover, το Ευρωπαϊκό Δραστήριο χρησιμοποιεί στο σύνολο του πόρους διότι είναι υποχρεωμένοι στο κάτω-κάτω και αυτό επιβεβαιώνει και την καταλληλότητα των αιτήματων, των αιτήσεων που υποβάλλουμε στην αρμόδια για τον προβλησμό αρχή για την κάλυψη των υποθέσεων που εξετάζει το δικαστήριο. Επίσης αποδίδουμε ιδιαίτερη προσοχή στην τακτικότητα των ε, δραστηριοτήτων και των εσωτερικών ελέγχων. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν για μια ακόμα φορά κρίνουμε πως ε, δεν χρειάστηκε να υποβληθούν κάποιες αρνητικές κριτικές ε, για το 2011 όπως συνέβη και το 2010. Παρακολουθούμε μάλλον τις συστάσεις ε, που γίνονται από την Επιτροπή σας και να πω ότι στο πλαίσιο της απαλλαγής 2010 υπήρχαν δύο συστάσεις που είχαν απευθυνθεί στο δικαστήριο η πρώτη αφορούσε τους εσωτερικούς ελέγχους και η άλλη ενημέρωση για, τους, για το ανθρώπινο δυναμικό. Όλες, όλες αυτές τις προφορίες συμπεριλήθηκαν στην ετήσια έκθεση του 2011. Σε ό,τι αφορά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας, είναι το δραστηριότητες στο Ευρωπαϊκό Δικαστηρίο σχετικά με τι δικαιοδοσίε. Ξέρετε ότι αυτέ οι δικαιοδοσίε είναι τρει και το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να διευθυντεί κάθε υπόθεση που φτάνει ενώπιον της. Ε, σε αυτό το πλαίσιο η συνεχής αύξηση των αιτήσεων που φτάνουν μπροστά στις τρεις αυτές δικαιοδοσίες αποτελεί ε, θέμα ανησυχίας, είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί και γι' αυτό προτείναμε συγκεκριμένα μέτρα στις νομοθετικές αρχές αλλά και στις αρχές αμμόδιε για τον προπολισμό. Αυτή η αύξηση των υποθέσεων, βλέπετε τον αριθμό για το 2011 ε, παρέμενε ε, ως ήχη αλλά φυσικά ε, το 2012 αυξήθηκαν αυτές οι υποθέσεις και η τάση παραμένει αυξητική. Θα ήθελα να αναφέρω και ένα στοιχείο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα το, το όργανό σας που αφορά την διάρκεια των διαδικασιών η διάρκεια των διαδικασιών προδικαστικών διότι αφορά τις πιο σημαντικές υποθέσεις που φτάνουν ενώπιον του δικαστηρίου είναι αυτές που αφορούν εκ των εκ του ε, τους πολίτες. Ε, μπορώ να σας πω ότι το 2012 καταλήξαμε στο ελάχιστο ιστορικό ελάχιστο για τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών, διότι πέσαμε από τους 16 μήνες στους 15,7. Παλιά αυτή η διάρκεια ήταν 25 μήνες και έχουμε καταλήξει τώρα στους 16 μήνες. Τώρα το 2003 που είχαμε φτάσει στο αριθμό που προανέφερα είχε οδηγήσει σε έκθεση του Κοινοβουλίου η οποία είχε εκφράσει τι ανησυχίε τους τώρα μέτρα τα οποία έχει προτείνει το δικαστήριο για την αντιμετώπιση αποτελεσματικά αυτή της εξέλιξη του αριθμού των υποθέσεων και της περιπλοκότητα των υποθέσεων αυτών. Τα μέτρα αυτά από πλευράς οργάνωσης των δικαιοδοσιών ε, είναι μέτρα νομοθετικής φύσης, προτάσεις που έγιναν από το δικαστήριο του 2011 όταν είχα αναφέρει ήδη σε εσά πέρυσι για την χρονιά 2011 αφορούσε την ε, δικαστήριο με την ε, ε, αναθεώρηση κάποιων διαδικασιών κάτι που θα συμμετείχαν περισσότεροι δικαστές ε, απελευθερώνουν κάποιους δικαστές από την αίθουσα 5, το τμήμα 5 για να βελτιωθεί η λειτουργία αυτής τώρα σε όλη φορά τις δικαιοδοσίας με την στήριξη του Ευρωκοινοβουλίου Αυτές οι τροποποίησεις ε, εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και ήταν σε ισχύ πέρυσι τον Οκτώβριο και εφαρμόζονται ήδη. Και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις τάσεις. Είναι θετικότατα τα μέτρα. Ε, το άλλο μέτρο το οποίο είχε προτείνει το δικαστήριο, ίσως να θυμίστε, αφορούσε τα δικαστήρια της Ένωσης, το ε, δεύτερο τμήμα του οργάνου μας που αντιμετωπίζει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα σχετικά με την περιπλοκότητα των υποθέσεων, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα, στον τομέα του ανταγωνισμού και το δικαστήριο το Μάρτιο 2011 έχει προτείνει να αυξηθεί ο αριθμό των δικαστών ώστε τα δικαστήρια να μπορούν να διευθετούν μέσα σε λογικά πλαίσια χρονικά τι υποθέσει. Ε, αυτή η πρόταση του δικαστηρίου έγινε αντικείμενο σε βάθος ανάλυση από το Συμβούλιο και στον αρμόδια για νομικά θέματα Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Σήμερα βρισκόμαστε στην εξή κατάσταση, όπου με την στήριξη του Κοινοβουλίου το Συμβούλιο δεν κατόρθωσε να συμφωνήσει επί της μεθόδου που θα εφαρμοστεί για την επιλογή αυτών των επιπλέον δικαστών. Το Συμβούλιο λοιπόν δέχτηκε ότι υπήρχε όντω πρόβλημα ε, ικανότητα δημοτικότητα του δικαστηρίου. Ε, περισσότερα κράτη-μέλη δέχονται ότι η καλύτερη λύση θα ήταν να αυξηθεί ο αριθμό των δικαστών αλλά οι συζητήσεις σε αυτό το στάδιο έχουν μπλοκαριστεί λόγω αυτής της αδυναμίας των κρατών να συμφωνήσουν επί της μεθόδου για την ε, επιλογή και διορισμό δικαστών. Το θέμα έχει λοιπόν κολλήσει. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο και ελπίζουμε πως θα εξευρεθεί η πολιτική λύση προκειμένου να προχωρήσουμε για την επίλυση αυτής της εμπλοκής αυτά, αυτά είναι τα νομοθετικά μέτρα φυσικά, αυτά έτυχαν συνοδείως με την χρησιμοποίηση πόρων στο εσωτερικό και όλα αυτά τα μέτρα στοχεύουν στο αυτό αποτέλεσμα, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν οι πόροι στο μέτρο του δυνατού για το core business, δηλαδή για τις δικαστικές εργασίες, τις εργασίες των δικαστών και των εισαγγελέων. Ε, υπήρξε λοιπόν μια επαναξιολόγηση των ε, θέσεων, ε, το θέμα των ε, βοηθών. Ζητήσαμε να υπάρχουν νέοι δικηγόροι σε αυτές τις θέσεις, που θα Το θέμα της μείωσης του προσωπικού, κάτι το οποίο δουλήθηκε από το Συμβούλιο μετά από συστάσεις της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου. μείωσαμε κατά 20% το προσωπικό του τον υπαλλήλων μας ε, αλλά διατηρήσαμε τους ε, πόρους, ε, τους οικονομικούς πόρους μόλον ότι μειώθηκε σημαντικά το προσωπικό και κάτι ακόμα πρόεδρε διότι πέρυσι είχε εκφραστεί ενδιαφέρον για την πληροφορική, ιδιαίτερα για το πρόγραμμα «Η Κούρια» χρησιμοποίηση λοιπόν της πληροφορικής για την επίδοση και κοινοποίηση των ε, εγγράφων. Αυτό το Κούρια, το η κουρια τέτοια εφαρμογή τον Νοέμβριο 2011, έχετε, τα, έχετε μάλλον τα αποτελέσματα αυτών των ε, δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της εκθέσεως για το 2012, αλλά ομολογουμένως είχε πολλά ευνοϊκά αποτελέσματα για την χρήση, αλλά και στο κόστος. Μειώθηκε το κόστος. Ε, μειώθηκε η χρήση του χάρτου κλπ. Επίσης, ε, Έχουμε μια νέα μηχανή αναζήτησης ε, στην ιστοσελίδα η που επιτρέπει μια πιο εύκολη πρόσβαση στην ομολογία του δικαστηρίου και όλα αυτά τα πράξαμε προκειμένου να προσεγγίσουμε τον πολίτη και να καταστούμε πλέον διάφανοι. Και τελειώνω πρόεδρε, κυρία Συγήτρια, τονίζοντας την ε, σημασία που έχει για μας ε, η χρήση του θα φροντίσουμε να υποβάλουμε τις κατάλληλες προτάσεις για να ε, απλουστεύσουμε τις εργασίες και να ευχαριστήσω και το Ευρωκοινοβούλιο για την στήριξή του σε πολιτικό επίπεδο, την ε, στήριξη από πλευρά τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα νομικέ υποθέσει και από μέρου τη Επιτροπή σα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο Γκαρτία από το ελεγκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Επιθυμώ εξ ονόματος του ελεγκτικού συνεδρίου να σας αναφέρω μια καλή είδηση. Να σας πω ότι το 2011 ο αριθμός των εκθέσεων που δημοσίευσε το όργανό μας ε, δημοσιεύθηκε δύο, δύο, ειδικές, δύο, εκθέσεις, δύο γενικές εκθέσεις, 41 ειδικέ 16 εκθέσεις και 7 και 8 συγγνώμη γνωμοδοτήσεις. Αυτή η θετική εξέλιξη επιβεβαιώθηκε το 2012 όπου δημοσιεύσαμε 25 ειδικέ εκθέσεις. Το 2011 Κάναμε 343 επισκέψεις ελέγχου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 36 εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή για να σας δώσω μια εικόνα της προσπάθειας που έχει καταβάλει το όργανό μας ε, για την άσκηση ελέγχων. Οι εκθέσεις αυτές ε, έγιναν με βάση την ε, τον κίνδυνο και την σημασία τους. Επίσης αποδοθούσαμε ιδιαίτερη σημασία στα ζητήματα που ξέρουμε ότι ενδιαφέρουν την Επιτροπή Ελέγχων προπολογισμού, ε, όπως παραδείγματο χάρη, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, η αγροτική ανάπτυξη, η ανάκτηση των, ε, των, των, των πληρωμών που έγιναν αχρεωστήτως το δικαστήριο δείχνει την βούλησή του για να στηρίξει το κοινοβούλιο στην άσκηση ελέγχου του προπολισμού. Το όργανό μας έβαλε σε εφαρμογή την ε, διαδικασία εξέλιξης, ανάπτυξης, προχωρήσαμε σε κάποιες, κάποιους ελέγχους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, διεθνή λογιστικά πρότυπα τα οποία έχει ορίσει ε, έχουν, αρχίσει, ε, ε, έχουν εφαρμόσει οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Το όργανό μας δημοσίευσε ένα νέο κώδικα δεοντολογίας, το, οι εκθέσεις κλειδί που, που αποδεικνύουν τις εργασίες της, του οργάνου μας ήταν θετικές. βελτιώθηκαν οι εκθέσεις που, έχουν, που υποβάλλουμε και εφαρμόστηκαν οι συστάσεις των διαφόρων επιτροπών και επίσης ε, εξελίξαμε και το προσωπικό μας. Ε, ε, φυσικά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, δουλεύουμε προς την κατεύθυνση αυτή και το 2012 πετύχαμε κάποια πρόοδα και αυτή η βελτίωση θα ουσιαστικοποιηθεί αυτή τη χρονιά. Το το όργανο μας θέλει να αποτελέσει μοντέλο για την διαχείριση των οικονομικών πόρων αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού. Μειώθηκε κατά 30% ε, έλλειψη προσωπικού το σχέδιο για το νέο κτίριο K4 ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και μέσα στα πλαίσια του προπολογισμού που είχε προβλεφθεί και ήδη ε, έχουν, έχει κατασταθεί το προσωπικό. Ο προπολογισμό μα εκτελέστηκε με αυστηρότητα και μπορέσαμε να κάνουμε εξοικονομήσει ε, στον κλάδο τη ασφάλεια, ε, του καθαρισμού και σε άλλε υπηρεσίε. Ο βαθμό εκτέλεση ήταν ε, υψηλότερε από αυτόν του ε, προηγούμενη χρονιά και θα είναι καλύτερο το 2012. Οι ε, συστάσεις του εσωτερικού ελεγκτή εφαρμόστηκαν κάτι το οποίο μας επιτρέπει να βελτιώσουμε περαιτέρω διαχείριση, μια λεπτομεριακή έκθεση της εργασία του εσωτερικού ελεγκτή υποβλήθηκε στον Επιτροπή σας και θα ήθελα να τονίσω ότι πέρυσι εδώ στην ίδια αυτή αίθουσα είχαμε μιλήσει για την βούληση του οργάνου μας ε, στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης να καλωστούμε αποτελεσματικότητα, αποτελεσματικότητα να υποβάλουμε καλύτερες εκθέσεις αλλά και ταυτόχρονα να εξοικονομήσουμε πόρους, να περιορίσουμε τις δαπάνες Και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να βελτιώσουμε τις εργασίες και να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Αυτό το πράξαμε το 2012 και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε το 2013. Έκθεση των δραστηριοτήτων και το παράρτημα του που σας ε, απεστάλλει χορηγεί λεπτομερείς ε, πληροφορίες ε, αλλά παραμένω στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Westlake έχει το λόγο από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τα μέλη της Επιτροπής ε, για την πρόσκληση και ε, για τη δυνατότητα που δίνει στην ΟΚΕ. Ε, θα προσπαθήσω να είναι εδώ μαζί σας. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Πριν από 4-5 χρόνια η ΟΚΕ ανέπτυξε ένα στέρεο μηχανισμό ελέγχου για μεγαλύτερη διαφάνεια, μέγιστη διαφάνεια και μέγιστη αποτελεσματικότητα. Επίσης η ΟΚΕ έχει και ένα μηχανισμό υποβολής εκθέσεων για τον οποίο έχετε συχνά ε, πει θετικά ε, πράγματα, με ε, σκοπό βέβαια πάντοτε τη μέγιστη διαφάνεια και αυτό βέβαια σημαίνει και εξπόστε έλεγχο των δικών μας δραστηριοτήτων. Θα ήθελα να κάνω δύο γενικές παρατηρήσεις. Πρώτον, ε, η συνεργασία με την Επιτροπή Περιφερειών που αναφέρθηκε και στην προηγούμενη συζήτηση ε, με τον κύριο Βόν και τον Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου Κλάους Φέλε. Η ΟΚΕ ε, και οι πολιτικές αρχές της εξακολουθούν να φρονούν ότι αυτή η συμφωνία συνεργασίας η οποία έθεσε, ανέφερε πολύ θετικά αποτελέσματα στα μεσο, στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρησή της μπορεί να ε, επιφέρει τεράστιες οικονομίες, ε, τεράστια εξοικονόμηση χρημάτων. Είναι κάτι το οποίο καταφέραμε από κοινού και δίνουν ένα πολύ καλό παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο κυρίαρχα ε, ε, κυρίαρχη, κυρίαρχα όργανα μπορούν να ε, διεξάγουν τα ε, οικονομικά τους. Ελπίζω να ακολουθήσουν σε αντίστοιχο πλαίσιο και άλλα τέτοια παραδείγματα. Μία τέτοια συνεργασία πρέπει να βασίζεται σε μία σχέση εμπιστοσύνης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά απολαμβάνουμε με τους συναδέλφους από την Επιτροπή των Περιφερειών που είναι και εκείνοι εδώ παρόντες. Θα ήθελα να πω επίσης ότι τα αιτήματα των ε, προϋπολο... του προπολογισμού ήταν πάρα πολύ υπεύθυνα τα τελευταία χρόνια. Έτσι θα συνεχίσουν και θα είναι και πλήρω συμβατά με τι κατευθυντήριε γραμμέ ε, με ε, τι επιστολέ του Επιτρόπου Λεβαντόφσκι. Ε, εμείς κατά παράδοση έχουμε πάρα πολύ στενές σχέσεις με τα μέλη της Επιτροπής μας. Ε, ο Γιάτσε Κράφτσεκ ε, συναντήθηκε με τον εισηγητή για την απαλλαγή εκθές και είμαστε βεβαίως στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε τυχόν ερωτήσεις. Όσον αφορά τώρα την έκθεση 2011 θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στην εξαιρετική εργασία των συναδέλφων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τους οποίους είχαμε πάντοτε εξαιρετική συνεργασία Πράγματι, ε, μας έδειξαν ένα πολύ σημαντικό ε, πρόβλημα που έχουμε και εμείς ε, ευθύ αμέσω προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε κατόπιν συστάσεων του συνεδρίου. Στις 12 Οκτωβρίου πέρυσι η Επιτροπή μας εφάρμοσε συγκεκριμένες κατευθυντήρες γραμμές σε σχέση με το συγκεκριμένο, με το συγκεκριμένο θέμα ε, λαμβάνεται έτσι υπόψη και η περίοδος της ε, λιτότητας και οι περικοπές του προπολογισμού και προσπαθούμε να εξορθολογικεύσουμε τις, ε, τα οικονομικά μας και προσπαθούμε να έχουμε και μια καλή ισορροπία μεταξύ των υπαλλήλων και των προσωρινών που προσλαμβάνουμε στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να πω επίσης ότι είμαστε ευγνώμονες στο ελεκτικό συνέδριο γιατί πραγματικά έδειξε ένα όχι πολύ σοβαρό αλλά ένα πραγματικό πρόβλημα. Ε, ευχαριστούμε πολύ αν ε, θεωρείτε ότι είμαστε κάθαροι και ευχαρίστω να απαντήσω σε ε, τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ το Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Βέσλικ και θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Γενικό Γραμματέα Στάλ από την Επιτροπή των Περιφερειών. Κύριε Στάλ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω εσάς και τον κύριο Λεμπρόν, τον πρόεδρο της ε, διοικητικής μας επιτροπής ε, που παρακολουθεί ε, πολιτικά τις εργασίες, να δώσετε το λόγο στον συνάδελφο για να κάνει μια γενική παρουσίαση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπε ο κύριος Στάλ, θα μοιραστούμε τη δουλειά ανάμεσα στο Γενικό Γραμματέα και μου, που είμαι ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσιονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων της Επιτροπής των Περιφερειών. Και η εδώ παρουσία μου μαρτυρεί την σημασία που αποδίδουμε την επαφή με την Επιτροπή σας, Πρόεδρε, και ιδιαίτερα με το Κοινοβούλιο. Θα έχω λοιπόν κάποια σχόλια πιο πολιτικής φύσης αναφορικά με τις δραστηριότητες μας για το 2011, διότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η τοπική αυτοδιοίκηση να εισακούεται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ε, περιφερειακής πολιτικής και την μεταρρύθμιση των ε, περιφερειακών ταμείων σε συνεργασία με την Προεδρία της Ένωσης και του Προεδρείου ε, επικεντρώσαμε την προσοχή μας στο πλαίσιο του δημοσιονομικού πολιτικού και σε συνεργασία με την Πολωνική και την Ουγγρική Προεδρία ε, εκδώσαμε γνωμοδότησεις για το θέμα τη ε, συνοχή, ε, την ΠΑΚ, την ΚΑΠ του 2020, την ΕΠΣ του 2020, το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και ούτω καθεξή. Δημιουργήθηκαν κάποια δίκτυα για την παρακολούθηση τη Ευρωπαϊκή Στρατηγικής 2020 και τη Επικουρικότητα. Και με λίγα λόγια σα πω ότι αυτέ οι πολιτικέ κατευθύνσεις ε, παρατάθηκαν και το 2012 διότι μπορούσαμε να καταγράψουμε αποφάσεις ε, που ε, συμφωνούν με τις ε, απόψεις και νομοδρήσεις της Επιτροπής των Περιφερειών. Αναφέρομαι στην πολιτική συνοχής με την αναγνώριση των ενδιάμεσων περιφερειών την θέμα της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας, τις συμβάσεις για την κοινή στρατηγική που αφορά στα την κοινή πολιτική. Επιμείναμε τώρα για τον ρόλο των περιφερειακών και ε, αρχών και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκηση, Κύριε Πρόεδρε, κυρία Συγκήτρια, θα ήθελα να τονίσω τις εξαιρετικές επαφές που είχαμε με του συζητητές της Επιτροπή των Περιφέρειων και του Ευρωκοινοβουλίου. Ε, ειδικά μεταξύ της, ενάμεσα στην Επιτροπή Ρέτζη της, ε, του Κοινοβουλίου και της ΚΟΤΕΡ της Επιτροπής των Περιφερειών. Σε όλες αυτές τις επαφές υπάρχει ένας εμπλουτισμός των ε, γνώσεων και βοηθάει στην ενίσχυση των πολιτικών περιφερειακών ζητημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, καταλήγει να σας προσκαλέσω σε μία από τις προσεχείς συναντήσεις της Επιτροπής θεσμικών ζητημάτων, διοικητικών και δημοσιονομικών. Ε, αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τις ανησυχίες μας στο πλαίσιο του προπολογισμού, αλλά και το πώς λειτουργεί το όργανό μας. Και τώρα θέλω να δώσω το λόγο στον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής των Περιφερειών για θέματα τεχνικά, τεχνικής φύσης που άπτονται της απαλλαγής 2011. Πολύ ωραία, αγαπητέ συναδελφέ, και δίνω το λόγο στον ε, Γενικό Γραμματέα. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Εισηγήτρια, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε κάποια διοικητική φύσεως ε, θέματα και ξεκινάω με το ότι η Επιτροπή των ε, Περιφερειών τόσο την σύσταση του ελεγκτικού συνεδρίου όσο και τη σύσταση της ε, αρχής απαλλαγής και αυτά τα δύο τα ε, παρακολουθεί εκ του σύνεγγης. Και έχουμε συστήσει μία τράπεζα δεδομένων όπου περιλαμβάνονται αυτές οι συστάσεις και όπου ελέγχουμε τη διαδικασία. Για το 2011 η Επιτροπή των Περιφερειών δεν έλαβε καμία σύσταση από το ελεγκτικό συνέδριο κατόπιν τούτου δεν τοποθετηθήκαμε. Για το 2010 είχαμε τρεις συστάσεις και τις εξετάσαμε. Θέλω να επισημάνω ένα θέμα το οποίο έπαιξε κάποιο ρόλο το 2011 δηλαδή την έκθεση που ζήτησε το Κοινοβούλιο σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας ανάμεσα στην Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η έκθεση σας έχει κατατεθεί, ο κύριος Βέστλικ ήδη το επισήμανε και η έκθεση αυτή περιλαμβάνει νομίζω μια πολύ σημαντική επισήμανση ότι η συνεργασία των δύο οργάνων οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση. Όσον αφορά άλλες συστάσεις σχετικά με τη διαδικασία της απαλλαγής, εδόθησαν κάποιες συστάσεις στην Επιτροπή των Περιφερειών. Ε, πρώτον το αίτημα ε, τα μέλη μας να δηλώσουν τα οικονομικά τους συμφέροντα. Εμείς το δεχτήκαμε και το Προεδρείο μας αποφάσισε ότι τα μέλη του Προεδρείου θα πρέπει να προβαίνουν σε μια σχετική δήλωση και η δήλωση αυτή αναφέρεται στο φάκελο κάθε μέλους μας. Ένα άλλο σημαντικό θέμα ήταν βέβαια για τη διοίκηση το να υπάρχει καλύτερος δημοσιονομικός προγραμματισμός. Γι' αυτό το λόγο η Επιτροπή μας ενίσχυσε τον μηνιαίο έλεγχο το 2011 η εκτέλεση του προϋπολογισμού πήγε πολύ καλά. Το 97,5% των υποχρεώσεων μας και το 95% ε, των πληρωμών μας ε, υλοποιήθηκαν. Και πέρα από αυτό, κατά την κατάρτιση του προπολογισμού του 2012, προσπαθήσαμε να είμαστε ιδιαίτερα συγκρατημένοι στον προγραμματισμό μας και γι' αυτό το λόγο προτείναμε σε σημαντική περικοπή κονδυλίων. Συνολικά λοιπόν το 2012 μας εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός από την αρχή προεπολογισμού η αύξηση είναι χαμηλότερη από εκείνη που έπρεπε να προϋπολογίσουμε για να διατηρήσουμε τις ε, συνήθεις ε, εργασίες μας. πάνω από 65% των δαπανών μας στην Επιτροπή των Περιφερειών αφορούν μισθούς και πληρωμές για τα κτίρια. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η απαραίτητη οικονομική διαχείριση μπορεί να επεκταθεί σε ένα μικρό τμήμα του προϋπολογισμού. Και αυτό όμως είναι μια πρόκληση πολύ σημαντική για ένα μικρό όργανο όπως είναι η Επιτροπή δική μας. Και είναι και επίσης ένας λόγος γιατί η Επιτροπή των Περιφερειών θεωρεί ότι η βελτίωση της διοίκησής της είναι ένα μόνιμο, σημαντικό θέμα. Βεβαίω και μπορέσαμε να συζητήσουμε με την Επιτροπή Ελέγχου ε, προπολογισμών, Η Επιτροπή των ε, Περιφερειών προέβησε αυτοαξιολόγηση. Εμεί επωφεληθήκαμε από την εμπειρία του ελεγκτικού συνεδρίου και με βάση αυτή την αυτοαξιολόγηση ε, μπορέσαμε να επιτύχουμε περαιτέρω βελτίωση από τη σχέση ανάμεσα στην πολιτική και τη διοίκηση. Και έτσι λοιπόν, ε, στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος μας ε, διαχείρισης ε, αναφέρουμε τις προτεραιότητές μας. Επίσης έχουμε συμφωνήσει με τη διοίκηση και με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται κατά πολύ η σωστή εφαρμογή του προϋπολογισμού και η βούληση για εξοικονόμηση. Και εφόσον το επιθυμείτε, είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Στάλ και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Γενικό Γραμματέα κύριο Χάρντεν. Ο κύριος Χάρντεν από την υπηρεσία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και ευχαριστώ να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Έχω στείλει ένα σημείωμα στην κυρία Τσέσκοβα απαντώντας ε, στο αίτημά της για πληροφορίες σε σχέση με την παρακολούθηση του ε, διαμεσολαβητή ε, στο ψήφισμα της απαλλαγής του Μαΐου σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2010. Το 2011 ήταν το πρώτο πλήρες έτος εφαρμογής της στρατηγικής του διαμεσολαβητή η οποία ε, υιοθετήθηκε το Σεπτέμβριο του 2010. Η ε, στρατηγική έθετε κάποιους στόχους ε, και όριζε κάποιους βασικούς δείκτες επιδόσεων σε σχέση με τους στόχους αυτούς. Δύο από τους στόχους της στρατηγικής είναι η παραγωγή καλύτερων αποτελεσμάτων και γρηγορότερων αποτελεσμάτων. Καλύτερα λοιπόν και ταχύτερα αποτελέσματα. Όσον αφορά τα καλύτερα αποτελέσματα αναφέρεται ένα σημείο, ότι δηλαδή εμπνευστήκαμε από τη δουλειά των ε, Σουηδών συναδέλφων μας ε, που κάνουν επιθεωρήσεις ε, των υπηρεσιών και οργανισμών και καταρτίζουν ένα πρόγραμμα επισκέψεων του διαμεσολαβητή ε, σε αυτούς τους οργανισμούς που είναι κάτι το οποίο στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και είναι πάρα πολύ ισχυρό μέσω εντοπισμού και διάδοσης των ε, βέλτιστων πρακτικών. Όσον αφορά τα ταχύτερα αποτελέσματα, θέλουμε να ε, επισπεύσουμε τη διαχείριση των υποθέσεων ε, ε, και αυτό βέβαια ούτως ή άλλως αναφερόταν και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την απαλλαγή για το 2010. Εδώ εμπνευστήκαμε από τους Γάλλους συναδέλφους και αλλάξαμε τη διαδικασία, την ευθυγραμμίσαμε τη διαδικασία αντιμετώπισης των ε, και έχουμε μια νέα διαδικασία παραδεκτότητας την οποία καταφέραμε να βελτιώσουμε, να φτάσουμε στο 70% το 2011 και ε, και πρέπει να πω ότι έχουμε φτάσει ήδη στο 85% για το 2012. Ο βασικός δείκτης που έχουμε θέσει εμείς είναι το 90% και ελπίζω να το φτάσουμε ή τέλος πάντων να πλησιάσουμε πολύ το στόχο αυτό του 90% το 2013. Επίσης, σχεδιάσαμε το 2011 ε, μια ουσιαστική αναδιάρθρωση του ε, γραφείου που εφαρμόστηκε από 1η Ιανουαρίου 2012 γιατί ο, η δουλειά του προγραμματισμού είχε ξεκινήσει από το 2011. Δεν θα πω σε πολλές λεπτομέρειες. Αναφέρεται και στην έκθεση, στην έκθεση δραστηριοτήτων του διατάκτη για το 2011. Ε, συμπερασματικά θα ήθελα να σχολιάσω ένα ακόμη θέμα το οποίο ετέθη στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την απαλλαγή όσον αφορά το ποσοστό αξιοποίησης ε, των ε, ε, πιστώσεων υποχρεώσεων. Το 2010 ήταν 86,5%. Το 2011 το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε στα 92,5%. 54% και με πολύ χαρά θα σας πω ότι το προσωρινό αριθμητικό στοιχείο που έχω για το 2013 είναι πάνω από 95% και ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε ε, το ποσοστό αυτό και να το βελτιώσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Γραμματέα και θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Γενικό Γραμματέα ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων, στον κύριο Ντόξη. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι τελευταίο αλλά φαντάζομαι ότι είμαι εξίσου σημαντικός. Όπως γνωρίζετε, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ε, είναι το μικρότερο και το νεότερο ε, όργανο που αναφέρεται στο δημοσιονομικό κανονικό. Είμαστε μια ανεξάρτητη υπηρεσία προστασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και όπως αναφέρεται Αναφέρθηκε και σήμερα πρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες ε, είτε ευρωβουλευτών είτε ε, άλλου προσωπικού και πρέπει να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ε, συνεργαζόμαστε με το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για νέες προτάσεις. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε όλο και περισσότερες υποθέσεις να αντιμετωπίσουμε για πολλούς λόγους. Τα αποτελέσματα καταρχάς της συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία έδωσε μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής ε, στην ομοθεσία για την προστασία δεδομένων, μεγαλύτερες εξουσίες στο Κοινοβούλιο και μεγαλύτερη έκκληση ε, για συμβουλές στη δική μας υπηρεσία και ηλικιώδης αύξηση των τεχνολογικών εξελίξεων. Το βλέπετε αυτό ε, και στην ψηφιακή ατζέντα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες είχαν ως αποτέλεσμα τεράστια αύξηση της συμβουλευτικής μας εργασίας. Από πλευράς εποπτείας τώρα υπάρχει αυξανόμενη ευαισθητοποίηση προστασίας δεδομένων ε, στα όργανα και τις υπηρεσίες της Ένωσης και από δικής μας πλευράς αυξάνουμε το βαθμό ε, συμμόρφωσης της δραστηριότητά μας με τον υπολείπον οργάνων και υπηρεσιών και αυτό σημαίνει ότι έχει αυξηθεί και η δουλειά μας σε σχέση με τις κοινοποιήσει, για παράδειγμα. Υπάρχει επίσης αύξηση της δουλειά μας λόγω της συνεργασίας με τις Εθνικές Υπηρεσίες Προστασίας Δεδομένων για την εποπτεία μεγάλης κλίμακας προστασίας δεδομένων που λειτουργούν και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Το λέω αυτό κύριε Πρόεδρε για να μπορείτε κι εσείς να κατανοήσετε για ποιο λόγο είχαμε μια πολιτική μετριοπαθούς αλλά ε, προοδευτικής σταθερής αύξησης κατά τα τελευταία χρόνια γιατί υποστηρίχθηκε αυτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάτι για το οποίο είμαστε ευγνώμονες. Το 2010 10, συγγνώμη, είχαμε ένα πρόγραμμα 39 ε, και για το 2013 ε, θα είναι 45. Δηλαδή τα τελευταία τρία χρόνια έχει υποστηρίξει κατ' εξαίρεση ε, τα δικά μας αιτήματα για αύξηση που ζητήσαμε και για το 2014-2020 για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο εννοώ πάνω από 50% λοιπόν αύξηση του προσωπικού, κάτι το οποίο δείχνει μόνο 7,8% στον προϋπολογισμό, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δουλεύουμε πολύ σκληρά να αξιοποιήσουμε, ε, να απορροφήσουμε το κόστος αυτής της αύξησης του προσωπικού στο πλαίσιο των οικονομικών περιορισμών μας. Δεδομένου λοιπόν ότι αυτή η σταδιακή αύξηση υποστηρίχθηκε από το Κοινοβούλιο κάθε χρόνο, γιατί οι μισθοί δεν έχουν προκαλέσει αύξηση στον προπολογισμό, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου ιδιαίτερω τα μέλη τη Επιτροπή σα, τα οποία τόσο αποτελεσματικά εργάστηκαν προκειμένου να μα υποστηρίξουν. Και θα ήθελα να πω ότι είμαι ιδιαίτερο ε, ευγνώμων στον Derek Βόν. Όσον αφορά το 2013 ε, και το οποίο θα ήθελα να το πω σε σχέση με όσους εργάζονται στην εποπτεία και στην τεχνολογία των πληροφοριών, γράψαμε στην κυρία Τσέσκοβα πέρσι ένα γράμμα σε σχέση με την ε, χορήγηση απαλλαγής του 2010. Τα συμπεριλάβαμε όλα αυτά. Δεν θα το επαναλάβω, θα συμπεριλάβαμε στην έκθεσή μας. Όμως θα ήθελα να σας πω ορισμένα πράγματα σε σχέση με το πού πηγαίνουμε, πού οδεύουμε στο μέλλον. Από το 2009 αναδιοργανώνουμε την υπηρεσία μας. Ολοκληρώθηκε να διοργάνωση το 2011 με έναν ε, ε, τομέα πολιτικής ε, πληροφορικής που συμπεριλήφθηκε στα τμήματα μας. Βελτιώνουμε το επίπεδο εκτέλεσης του προπολογισμού μας 76% το 2010, 85% το 2011, 2012 περίπου 90%. Η Μαριάν εδώ δίπλα μου κάθεται, η οποία φιλοδοξεί για μεγαλύτερο, για πιο καλό ποσοστό για αυτό το έτος, για το 2013. Θα ήθελα να πω ένα πράγματα και τη στρατηγική μας το 2013-2014. Το 2011 δρομολογήσαμε μια στρατηγική αναθεώρηση με διαβούλευση ε, του προσωπικού μας και πολλών ε, ε, εξημών που είστε παρόντες εδώ σήμερα, εξωτερική διαβούλευση με όργανα και υπηρεσίες και θα ήθελα να ευχαριστήσω ειδικότερα τους συναδέλφους στο ελεγκτικό συνέδριο και στο διαμεσολαβητή γιατί μας έδωσαν πάρα πολύ καλές συμβουλές πώς να οργανώσουμε οργανώσουμε την αναδιάρθρωση. Δύο στόχοι. Πρώτον, πώς μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά αυτό που κάνουμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όταν το κάνουμε και που μπορούμε, πώς μπορούμε να αυξήσουμε τον αντίκτυπο στην προστασία, της προστασίας δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η αναθεώρηση είχε ως αποτέλεσμα αυτό εδώ το έντυπο που σας δείχνω και το οποίο θα σας το παρουσιάσουμε ε, σήμερα το απόγευμα. Ε, θα το παρουσιάσουμε επισήμω. Είναι η στρατηγική μας, ε, η μεσοπρόθεσμή μας στρατηγική 2013 με 2014 και συμπεριλαμβάνει σημεία τα οποία συζητήθηκαν στο Κοινοβούλιο στο παρελθόν, ε, ένα σύνολο 10 ε, βασικών δικτών ε, επιδόσεων και 16 δικτών εσωτερικών που εμείς από την πλευρά μας θα παρακολουθούμε και θα αξιολογούμε. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. We now listened to the statements of the General Secretaries. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Οντί, στον Ζαν Πιέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν συντομία, θα θέλαμε να έχουμε περαιτέρω επαφές με την Επιτροπή των Περιφερειών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, αξιολόγησή τους αναφορικά με την κοινή διαχείριση. Ε, θα θυμίσετε την κριτική που είχα που αναφέρει σχετικά με αυτή την κοινή διαχείριση και προσωπικά με ενόχληση η συζήτηση που είχαμε επί του διορθωτικού προπορισμού 2012 όπου μετά από κάποιο λάθος υπολογισμού μας έλειπαν 9 δις για να μπορέσουμε να ε, ανταποκριθούμε. Τώρα, ε, δεν είμαστε σε θέση να εκπληρώνουμε σωστά τις ε, υποχρεώσεις μας. Ε, δεν είναι κάτι το οποίο μας τιμά και δεν τιμάται οι δημοσιονομικές δομές των οργάνων μας. Πώς θα μπορούσαμε ανάμεσα στην Επιτροπή Περιφερειών και την Επιτροπή μας Ενέργου Προπολισμού να εξετάσουμε το κύκλωμα το οικονομικό. Θα ήθελα, είχα προτείνει μάλλον στον Πρόεδρο Καλτέρα, δεν ξέρω αν το ε, ελεγχτικό συνέδριο το σκέφτηκε, διότι θα μπορούσε να διαρματίσει έναν ρόλο προειδοποιητικό, θα έλεγα, όταν προκύπτουν τέτοια προβλήματα, προκειμένου να μην επαναληφθούν στο μέλλον και τα κυκλώματα αυτά να μπορούν να λειτουργούν ορθά. Αυτή είναι μια πρόταση που κάνω στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα έλεγα εμπλέκονται ιδιαίτερα στην ε, λειτουργία και διαχείριση ε, των ε, περιφερειακών αρχών. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που δεν έδωσα το λόγο στην εισηγήτρια και Τσέσκοβα, έχετε το λόγο. E, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι το θέμα της διαδικασίας. Ο εκπρόσωπος του ελεκτικού συνεδρίου αναφέρθηκε στο Συμβούλιο, αλλά το Συμβούλιο δεν ήταν αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης, οπότε θα το παραλείψω αυτό. Επίσης αναφερθήκαμε σε μία μόνο παρατήρηση του ελεκτικού συνεδρίου που αφορά την ΟΚΕ. Είναι γεγονός ότι αυτό αφορά ε, τους... Ε, την περίπτωση ενός ε, εργαζομένου, όπως μας την παρουσίασε ε, ο εκπρόσωπος. Ε, το συζήτησα αυτό εχθές με τον εκπρόσωπο της ΟΚΕ. Να επιστρέψω τώρα σε ερωτήσεις που θέλω εγώ να θέσω γιατί από ό,τι κατάλαβα το πρόβλημα της ΟΚΕ, από ό,τι κατάλαβα διορθώνεται ή τέλος πάντων θα διορθωθεί. Θα λοιπόν μερικά ερωτήματα για την ΟΚΕ και για κάποια άλλα ε, όργανα για τα οποία εγώ είμαι αρμόδια. Για την ΟΚΕ καταρχάς. Με ποιο τρόπο χρησιμοποιείτε το κόστος ε, επικοινωνίας. Έχετε καταγράψει το κόστος της βελτίωσης ε, ε, απορρόφησης των κομβιλίων στην Επιτροπή σας. Η συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών το είπαμε πολλές φορές. Υπάρχει μια δυνατότητα να καταλήξουμε στις ε, ίδιες, να, να δούμε τι ύψους οικονομίες έγιναν από τη συνεργασία των δύο αυτών οργάνων. Υπάρχουν κάπου διαθέσιμα αυτά τα στοιχεία. Επίσης, ε, πώς συμμετέχει η Επιτροπή σας ε, στις εγκαταστάσεις της πρόσχολικες του Συμβουλίου και σε ποιο βαθμό μπορούν οι συνάδελφοί σας να τις χρησιμοποιήσουν. Μία ακόμη ερώτηση θέλω να κάνω σε σχέση με τις οικονομίες που γίνονται με τη χρήση των ε, κτηρίων ε, για, τις, ε, για εξωτερικά γεγονότα και πώς επιλέγετε αυτά τα εξωτερικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις σας. Για το 2010 τώρα προτείναμε ένα νέο σύστημα αποζημίωσης των εξόδων ταξιδίων επί τη βάση πραγματικών εξόδων δηλαδή. Η διαδικασία αυτή ακόμη την χάνει επεξεργασία ε, από το Συμβούλιο. Από ό,τι κατάλαβα, αν εγκριθεί θα υπάρχει ένα παράλληλο διάστημα, ένα διάστημα παράλληλης αποζημίωσης, ε, δηλαδή το σύστημα πραγμα... αποζημίωσης επί τη βάση πραγματικών εξόδων και το παλιό σύστημα με τα καταποκοπήν ποσά. Για αυτή την περίοδο μετάβασης ε, παράλληλης χρήσης των δύο συστημάτων μπορεί να γίνει επιλογή του ενός ή του άλλου συστήματος. Ε, όσον αφορά τώρα τον εξυγχρονισμό ε, του συστήματος ε, διαχείρισης και αποθήκευσης των εγγράφων, μιλάω δηλαδή για τις υποδομές της τεχνολογίας των πληροφοριών. Σε ποια φάση βρίσκεται αυτό το σύστημα. Να περάσω τώρα στις ερωτήσεις για την Επιτροπή Περιφερειών. σε σχέση με το CISPER 2 και το σύστημα ίντρανετ. Πώς έχουν τα πράγματα, αν υπάρχουν πολλά ε, αιτήματα μεταφράσεων, κάνετε εξωτερική ανάθεση. Και ποιοι είναι οι κανόνες επιλογής τότε των, ε, της παροχής αυτών των υπηρεσιών. Πώς γίνεται αυτή η εξωτερική ανάθεση των μεταφράσεων. Όσον αφορά τώρα την απαλλαγωγή για το 2010, μιλήσαμε για τη βιντεοδιάσκεψη. Η βιντεοδιάσκεψη χρησιμοποιείται και πώς γίνεται η αποζημίωση των εξόδων ταξιδίων σε αυτή την περίπτωση. σε σχέση με τα έξοδα ταξιδίων, πώς γίνεται η αποζημίωση σε επίπεδο Επιτροπή Περιφερειών. Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο βέβαια για να λάβουμε τις απαντήσεις. Να περάσω τώρα στο διαμεσολαβητή. Θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το κόστος ε, για την γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του διαμεσολαβητή. Ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με το βίντεο κλιπ, με τη χρήση του ηλεκτρονικού ε, ενημερωτικού φυλαδίου, του newsletter, γιατί αυτά τα δύο ε, θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ε, προβολή του γραφείου του διαμεσολαβητή στο κοινό. Μιλήσατε επίσης για ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξέλιξης. Μήπως μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα γι' αυτό τι σημαίνει επακριβώς και επίση ε, τι προγράμματα τεχνολογία των πληροφοριών έχουν ολοκληρωθεί και ποια έχουν αναβληθεί για το μέλλον. Όσον αφορά τώρα τον, ε, την ε, προστασία δεδομένων, έχετε ένα νέο εσωτερικό εγχειρίδιο που διέπει την πρόσληψη νέων εργαζομένων. Συμπεριλαμβάνει άραγε τη συνεργασία με την ΕΨΟ, ερωτώ και για ποιο λόγο έχετε προβλέψει δύο συγκεκριμένες θέσεις για τη σεξουαλική παρενόχληση. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης και πώς ε, τις ε, ε, επιλύεται αυτές τις περιπτώσεις σε επίπεδο εσωτερικό. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο λογισμικό για τον έλεγχο ή συγκεκριμένα της προστασίας δεδομένων. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του λογισμικού και πώς εξασφαλίζεται την επεξεργασία, τη μεταχείριση των ευαίσθητων δεδομένων. Αυτά είναι τα ερωτήματα που ήθελα να θέσω για ε, τις, ε, τα όργανα για τα οποία είμαι υπεύθυνη. Τώρα να περάσω στα ερωτήματα του κυρίου Τσερνίσκη για το δικαστήριο και το ελεγκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να τα παρουσιάσω. Ναι, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, σε πέντε λεπτά δεν θα έχουμε άλλη διερμηνία. Προτιμάτε μήπως μία απάντηση στις ερωτήσεις σας γραπτός, ίσως ενδεχομένως να είναι μια καλύτερη λύση αυτή. Σας δίνω το λόγο και για τον κύριο Τσαρνέσκι, αν θέλετε. Ναι, μπορούμε να λάβουμε γραπτές απαντήσεις στις ερωτήσεις που έθεσα. Το ίδιο ισχύει και για τις ε, ερωτήσεις του κυρίου Τσαρνέσκι. Μπορούμε και πάλι να ζητήσουμε γραπτές απαντήσεις και να δώσουμε το λόγο στους υπόλοιπους ε, συναδέλφους αν θέλουν να θέσουν και άλλα ερωτήματα. Μάλιστα. Πολύ καλά. Ναι. Ε, ο κύριος Κάλφιν ήθελε βέβαια να θέσει ένα ερώτημα και ευχαριστώ που είστε πραγματικά τόσο συνεργάσιμοι και επίκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις ε, για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ελεκτικό Συνέδριο. Για το δικαστήριο γνωρίζουμε ότι το δικαστήριο ε, αναζητάει γλωσσομαθείς νομικούς για τη μετάφραση διαφόρων υποθέσεων. Θα ήθελα να ρωτήσω ότι το εξής. Αυτή τι οι μελλοντικοί συνεργάτε θα πρέπει να βρίσκονται στο Λουξεμβούργο ή μπορούν να βρίσκονται και σε άλλες χώρες και να έχουν επαφή μέσω ε, υπολογιστών. Τώρα προς το ελεγχτικό συνέδριο έχετε τη δυνατότητα να επανεξετάσετε τα αποτελέσματα Εξετάζεται όμως και την, την εφαρμογή των ε, συστάσεων. Ε, πώς κάνει γίνεται αυτή η παρακολούθηση και κάτι ακόμα. Οι εξωτερικοί ελεγκτές ε, συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχων Προϋπολογισμού. Και τέλος, θα ήθελα να λάβω αυτές τις ε, απαντήσεις γραπτός. Κάτι που φορά όλα τα όργανα. Αυτά που είπε ο διαμεσολαβητής για τους δείκτες αποτελεσματικότητας θα ήθελα να ζητήσω, να ρωτήσω. Προβλέπετε την εφαρμογή αυτού του δείκτη και την υποβολή σχετικών εκθέσεων. Και κάτι ακόμα. Καλύτερη χρήση της πληροφορικής θα μπορούσε να καταστήσει πιο αποτελεσματικές εργασίες αλλά και πιο διάφανες. Προβλέπετε να λάβετε κάποιο μέτρο σχετικό. Ευχαριστούμε πολύ ε, κύριε Κάλφιν, αγαπητές συνάδελφοι. Τώρα πλέον δεν μπορούμε να δώσουμε προφορικές ε, απαντήσεις. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω τους εκπροσώπους των άλλων οργάνων κατά πόσον μπορούν να μας καταθέσουν μία γραπτή απάντηση. Βλέπω νεύεται καταφατικά. Ε, κατόπιν τούτου ευχαριστώ εκ μέρους της εισηγήτριας της Επιτροπής για την ε, γνωμοδότησή σας, για αυτά που μας είπατε και ε, θεωρούμε ότι είναι πολύ καλό το ότι θα μας δώσετε γραπτές απαντήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ που συμμετείχατε στη σημερινή συνεδρίαση. Η συγγήτρια θέλει το λόγο. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το ηλεκτρικό συνέδριο, το δικαστήριο, αλλά και όλους όσοι συμμετείχαν στις εργασίες μας. Μόνο ότι δεν είχαμε και πολύ χρόνο τη διαθέσή μας για αυτό το κομμάτι. Ευχαριστώ και τη γραμματεία της Επιτροπής, διότι η συνεργασία ήταν άψογη όλες οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι απαντήσεις ε, των συναδέλφων θα συμπεριληφθούν στην ε, έκθεσή μου. Ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια, την κυρία Τσέσκοβα. Ευχαριστούμε ε, τους γενικούς γραμματείς και τους άλλους ε, εκπροσώπους των οργάνων ε, και θα πάμε τώρα για μεσημεριανό γεύμα και το πρώτο θέμα θα είναι η ειδική έκθεση την οποία αναβάλαμε. Στις 3 ε, η ώρα ε, θα συνεχίσουμε. Γεια σας.